αλλά θα ήθελα να παρουσιάσω αλλά συγχαρητήρια στους Ισπανούς συναδέλφους. Ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τους φίλους μας τους Ισπανούς που κέρδισαν ε, το παγκόσμιο κύπελο στο ποδόσφαιρο. Καλά το πάλεψαν οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί κάπως λιγότερο. Τέλος πάντων θα έχουν... πάλι την ευκαιρία σε κάνα δύο χρονάκια και πάλι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχω να καλωσορίσω έναν προσκεκλημένο τον Υπουργό Εθνική Ανάπτυξη τη Ουγγαρία, τον κύριο Μπέλγκη. Καλώς ήρθατε. Θα παρακολουθήσει εργασίες μας ο κύριος Μπέλγκη. Φέλεγγι. Καθώς είναι ο επόμενος στη σειρά για την Προεδρία και καλωσορίζω και τους υπουργούς που έχουμε σήμερα παρόντες από το Βέλγιο, τον κύριο Ζων Κλοντ Μαρκούρ και τον κύριο Βερμά Σερέξ. Καλώς ήρθατε. Θα πρέπει όμως να ρωτήσω πρώτα τους συναδέλφους αν υπάρχουν παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Όχι από ό,τι βλέπω. Ας ξεκινήσουμε το πρώτο θέμα της τη διάταξη τότε. Οι δύο Υπουργοί. Σας καλωσορίζω θερμά και εύχομαι κάθε επιτυχία για τη Βελγική Προεδρία. Δύσκολη στιγμή αναλαμβάνετε την Προεδρία και μόλις ένα μήνα πριν από τις διακοπές ή στο ξεκίνημα των διακοπών έχετε δύσκολη δουλειά. Αλλά από την άλλη, επιστρέφοντας από τις διακοπές, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, έχουμε μπροστά μας και μεγάλα θέματα να επιλύσουμε. Και γι' αυτό εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Ποιος θέλει να ξεκινήσει πρώτος, ε, ο κύριος Σεγέξ, ο κύριος Μαρκούχ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μεγάλη χαρά για μένα και το συνάδελφό μου να είμαστε μεταξύ ανάμεσά σας να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα, διότι εδώ και ένα χρόνο, σαν Ευρωβουλευτής, στις 14 Ιουλίου, είχα αναλάβει τα καθήκοντά μου, είμαι σχεδόν ένα χρόνο μετά, ε, πήγα μαζί σας ε, στο Στασβούργο με κάποιους από εσάς, να ξεκίνησε τη του Κοινοβούλιο, παρετήθηκα το σημαντικότατο αυτό αξίωμα να είμαι Ευρωβουλευτής, διότι μου έδειξαν εμπιστοσύνη και έγινε την πρόεδρος της κυβερνήσεως της Βαλονίας και της γαλλιόφωνης κοινότητας. Αλλά πάντα με ενδιέφεραν τα ευρωπαϊκά θέματα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι σαν επικεφαλής του κόμματός μου έκανα προκλητική εξατία ευρωπαϊκή πριν από ένα χρόνο και είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά που είμαι μεταξύ σας σήμερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας, ενισχύθηκε όσον αφορά τις αρμοδιότητές του και δεν είναι ένα πρώτο βήμα που και θα ακολουθήσουν και άλλα. Ε, θα έχει μεγάλη σημασία το Κοινοβούλιο κατόπιν της εφαρμογής της συνθήκης αυτής. Και σαν υπουργό ενός, ενός ομοσπονδιακού κράτους θέλω να πω ότι έχουμε μεγάλη, μεγάλη χαρά για το Μπενουά Σενέξ και μένα να είμαστε εδώ διότι είμαστε δύο υπουργοί περιφερειακοί που αντιπροσωπεύουμε όμως όλο το Ομοσπονδιακό κράτος και σαν υπουργοί που εκπροσωπούμε το Βέλγιο είμαστε εδώ ενώπιον σας και όχι απλώς σαν ε, υπουργοί που εκπροσωπούμε ένα τμήμα του κράτους. Είναι μικρό κράτος το Βέλγιο και όπως είπε ο Πρόεδρος ε, δεν έχει ομοσπονδιακή κυβέρνηση πλήρη, αλλά λειτουργούν οι διάφοροι φορείς, ούτως ώστε η Βελική Προεδρία θα εκτελέσει τα καθήκοντά της κατά το δεύτερο εξάμεινο του 2010 και θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας όσο καλύτερα γίνεται. Είμαστε στη διάθεση του Κοινοβουλίου, ανά πάσα στιγμή που θεωρεί χρήσιμο το Κοινοβούλιο αν υπάρξει κάποια επιθυμία. Για να έρθετε να μιλήσετε και σε μένα ή να έρθετε σε επαφή με κάποιους συναδέλφους για να σας δώσουμε κάποιες απαντήσεις με τα χαράς να ανταποκριθούμε σε τέτοιες ε, ε, παρακλήσεις σας. Πολύ σύντομα, διότι ήδη μπορέσατε να δείτε ποιες είναι οι προτεραιότητες της Βελικής Προεδρίας Εφόσον είμαστε πολλοί, μερικά λεπτά θα αναφερθώ στις προτεραιότητες. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να μπω στα ουσιώδη. Η Βελική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα σημειωθεί από την εφαρμογή, την ελοπιστατική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το 2020. 2020-2020. Όσο μας αφορά, βασική πρωτοβουλία θα είναι προφανώς η βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης και επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε ε, Σα έδωσα πρώτα τα γερμανικά, στα γερμανικά το κείμενο. Αυτό αφορά μια μελέτη που κάναμε όσον αφορά τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέψτε μου λοιπόν στην αρχή της συνεδριάσεως να σας υποβάλω αυτό το έγγραφο που είναι στις τρεις εθνικές γλώσσες του Βελγίου, γερμανικά, ολλανδικά, γαλλικά και συνοδεύονται τα κείμενα αυτά που είναι μετά στα αγγλικά για να είναι κατανοητό το κείμενο από όλους. Θα είναι στη διάθεσή σας λοιπόν αυτό το κείμενο για όλα τα μέλη της Επιτροπής σας και θα τροφοδοτήσει τον προβληματισμό όσον αφορά την βούληση και θέληση που έχουμε να κάνουμε αυτή τη βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησεως ε, στο επίκεντρο να τη βάλουμε της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι η αναφορά, το σημείο αναφορά των εργασιών μας. Είμαστε πεπισμένοι ότι η ευρωπαϊκή οικονομία είναι και θα παραμείνει βιομηχανική. Μια βιομηχανική βάση ισχυρή θα συμπεριλαμβάνει απαραίτητα μια ανθρώπινη διάσταση, βιώσιμη διάσταση, ε, με την ευρύτερη δυνατή αποδοχή, χωρίς πολλούς περιορισμούς, κάτι που ισχύει πολλές φορές, για να μπορέσουμε να βρούμε μια απάντηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς πολλούς περιορισμούς Λαμβάνοντας λοιπόν όψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις και μετατρέποντας τους περιορισμούς και τα όρια σε δυνατότητες. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και κοινωνική διάσταση, διότι βασίζεται σε ανθρώπους η βιομηχανία και η μεταμόρφωση της βιομηχανίας και οικονομίας στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησεως δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτό το στοιχείο. Και τέλος θα συμπεριλαμβάνει και την καινοτομία σαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα πλαίσια της ε, παγκοσμιοποίησης. Η βασική προτεραιότητα του Βελγίου που είναι βασική και εγκάρσια είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω κυρίως μίας βιώσιμης ε, βιομηχανικής πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα βασίζεται επίσης στην καινοτομία και στα εργαλεία που απεδείχθησαν αποτελεσματικά στους δύο αυτούς τομείς, δηλαδή την πολιτική της ομαδοποίησης της προσπάθειας του clustering. Τις μέρες λοιπόν που τις επόμενες 14 και 15 Ιουλίου για αυτό το λόγο ετοιμάζουμε μια άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου Βιομηχανίας διοργανώνεται σε δύο μεγάλες πτυχές σε βιομηχανική πολιτική στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης αυτή είναι η μία πτυχή και η καινοτομία στη βιομηχανική της διάσταση είναι η άλλη πτυχή. Η καινοτομία θα αντιμετωπιστεί και θα συζητηθεί σε μια κοινή συνεδρίαση με τους Υπουργούς Έρευνας και Βιομηχανίας που εκεί θα τονιστεί η εγκάρση κάθε τη διάσταση της καινοτομίας. Τις 2 Ιουλίου που πέρασαν ξεκίνησε η Βελική Προεδρία και γι' αυτό το γεγονό αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε πούμε, λοιπόν με μια διάσκεψη στην Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή ΟΚΕ, επ' αυτού του θέματο ε, καινοτομία. Εκεί συμπεριλήφθησαν πολλοί, συμμετείχαν πολλοί κοινωνικοί εταίροι, το Κεντρικό Συμβούλιο τη Οικονομία για το Βέλγιο και τη Περιφέρεια που είναι στο, στην, στο Βέλγιο, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο τη Βαλονία, των Βρυξελών και τη Φλάνδρα. Που υπέβαλαν ερωτήσει και αιτήματα και Θέλουμε οι προσδοκίες οι οποίες εξεφράστησαν ε, να τύχουν ικανοποίησεως. Αυτά που αναφέρθηκαν ε, αφορούσαν κυρίως την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την καινοτομία, την εφαρμογή μιας ε, πολιτικής κόμβων ευρωπαϊκή κλώστος, μια πρόσβαση στη μη τεχνολογική καινοτομία, αλλά επίσης και την χρήση δικτών ποσοτικών και ποιοτικών. Θεωρούμε λοιπόν σημαντικό να ακολουθήσουμε οριζόντια προσέγγιση στον αφορά την πολιτική βιομηχανική και ταυτόχρονα τομεακή προσέγγιση. Οι τομεί έχουν τι ιδιαιτερότητέ του, Κάποιοι από αυτού μπορούν να αντιμετωπιστούν σε εθνικό όπω όπως επιθυμούν κάποια κράτη-μέλη, αλλά θεωρούμε όμως ότι η διεθνή διάσταση των μεγάλων επιχειρήσεων απαιτεί επίση μια ευρωπαϊκή προσέγγιση ε, για να καλυφθούν οι διάφορε ιδιαίτερότητε. Ο κ. Ζουρκέν, ο πρόεδρος της Σολβέ και υπεύθυνο της Χάρσελε Ομιτάλ ε, ασχολήθηκαν με αυτό, θα μιλήσουν ε, σε αυτό, πάνω σε αυτό το θέμα στο περιθώριο της άτυπης συνεδριάσεως. Κάποια θεματικά θέματα θα συζητηθούν σίγουρα ε, στα πλαίσια τη τομέα βιομηχανία του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας. Ο των δημοσίων αρχών είναι πάρα πολύ κομβικός και το έδειξε αυτό η κρίση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει κάποιες ανακοινώσει, οι οποίες άμεσα ή έμεσα αφορούν αυτή την ε, κρίσιμη ε, θέση και ρόλο των ε, δημοσίων αρχών όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως γιατί αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια μια αυθεντική βιομηχανική πολιτική. Για παράδειγμα, θέλω να σα αναφέρω ότι γίνεται να ανακοίνωση που αφορούσε τι δημόσιε συμβάσει πριν την θέση σε εμπορία. Ε, θεωρώ ότι υπάρχει ε, το θέμα των κρατικών ισχύων που θα πρέπει να θυγεί στα πλαίσια τη μετασχηματισμού τη οικονομία και θα πρέπει γι' αυτό το λόγο να γίνει ένα συντονισμό μεταξύ όλων των τομέων, τόσο ώστε να μπορούμε να έχουμε τι άλλε πρακτικέ και να έχουμε τέτοιου είδου συντονισμό που είναι βασικό, τόσο ώστε να έχουμε καινοτομία στην βιομηχανία. Επίση, θα πρέπει να φρεσκάρουμε, να δώσουμε νέα όθηση στην οικονομία de l'industrie européenne. Nous organisons une conférence και να γίνει πράσινη οικονομία και αυτό για να αντιμετωπίσουμε τι ενεργειακέ προκλήσει. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται μέσα στην Ευρύωση σε γίνει τη διάσκεψη στο ΣΠΑ και θεωρούμε ότι αυτό θα βοηθήσει να γίνει πράσινη οικονομία και θέλουμε να γίνει μια ομαλοποίηση και γι' αυτό και προβληματιζόμαστε γύρω από αυτό το θέμα. Θέλουμε μετασχηματισμό τη οικονομία που είναι η καρδιά τη βιομηχανική πολιτική και από αυτού έχουμε επεξεργαστεί ιδέε με κάποια ομάδα διαφόρων ερευνητών. Προέρχονται πολλέ χώρε τη Ευρώπη και τα αποτελέσματα πρόκειται σύντομα να βγουν στο φω ε, στο website τη Βελγική Προεδρία και αυτοί οι ερευνητέ έχουν επεξεργαστεί το πώς θα ταυτοποιήσουν αυτές τις προκλήσεις με τις ανάγκες των ε, επιχειρήσεων και γι' αυτό και έχουν ε, στείλει μηνύματα, μηνύματα κλειδιά και ε, θα πρέπει να δούμε και την καινοτομία για τις ΜΜΕ που είναι αυτό βασικό όσον αφορά τη συνέπεια της πολιτικές και την διακυβέρνηση και κάτι άλλο είναι πάρα πολύ βασικό για μας να εμπλακούν όλοι η κοινωνική εταίρη ε, για αυτές τις αλλαγές που πρέπει να περάσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία και αυτό επίσης ε, πρόκειται να συζητηθεί σε διάσκεψη που θα γίνει στο ΣΕΡΕΝ κοντά στην Λιέγη μέσα Νοεμβρίου και τέλος δεν μπορώ να μην θίξω κάτι το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ τις μικρομεζές επιχειρήσεις αυτές οι οποίες κυρίως έχουν φύγει από την κρίση έχουν πάνω από από 180.000 επιχειρήσεις στην Ευρώπη που κλείσανε ε, μέχρι σήμερα, την περασμένη χρονιά. Και γι' αυτό χρειάζονταν αρδιαθρώσεις πάρα πολύ σημαντικές που έπληξαν τις θέσεις εργασίας, τους εργαζόμενους, αλλά επίσης η, κλίση, η κρίση έχει πλήξει και τους προμηθευτές και αυτούς που έχουν κάποια σχέση υπεργολαβίας. μιέψουν το 10% της απασχόλησης και του ΕΕ στην Ευρώπη και γι' αυτό θα πρέπει να κινηθούμε στα πλαίσια της αναθεώρησης του Small Business Act. Οπότε να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την καινοτομία, θα γίνει με τη χρηματοδότηση και να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε ένα πλαίσιο που να διευκολύνει την καινοτομία. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του 2008 της Κομισιόν όσον αφορά <clears throat> αυτές αυτές τις ομαδοποιήσεις ε, παγκόσμια βεληνικού, θέλουμε να ξεκινήσει μια αυθεντική ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά αυτή την ομαδιοποίηση, το clustering και επίσης ε, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε είδους ε, πρωτοβουλία για αυτά τα θέματα και περιμένουμε πώς και πώς το πώς θα μας βοηθήσει το Κοινοβούλιο σε αυτές τις πρωτοβουλίες και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και παρακαλώ τώρα. Τον κύριο Μαγνιέτη να λάβει το λόγο και του συναδέλφου όταν κάνουν ερωτήσει να είναι στο δυνατόν πιο σύντομοι γιατί έχουμε πολλή δουλειά και πρέπει να είμαστε οικονόμοι με τον χρόνο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Όπως και ο συνάδελφος του ο κύριος Μαρκού, θέλω να σας ευχαριστήσω που μας δεχθήκατε σήμερα εδώ και που μας επιτρέπετε να σας εκθέσουμε ο καθένας στο χαρτοφυλάκιό του τις προτεραιότητες της Βελγικής Προεδρίας ως προς την έρευνα. Για να μπορέσει κανείς ε, να εξασφαλίσει έξοδο από την κρίση με διαφύλεξη όμω και το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης, θα πρέπει να επιλέξει η Ευρώπη ένα νέο τύπο ανάπτυξης με κινητήριες δυνάμει στη γνώση, την καινοτομία και όσο δυνατόν λιγότερη κα... κατάχρηση, εκμετάλλευση των, ε, πε... των πεπερασμένων φυσικών πόρων. Και έτσι λοιπόν η Βελγική Προεδρία ιδιαίτερα με το στόχο αυτό θα έχει σαν στόχο να ενισχύσει την έρευνα, την καινοτομία, την ανώτατη εκπαίδευση για να αναπτύξει ακόμη περισσότερο το δυναμικό για την έρευνα στην Ευρώπη και να το μετατρέψει σε συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα. Αυτό με ταπεινοφροσύνη φυσικά θα το προτείνουμε, αλλά και με ρεαλισμό θα το υλοποιήσουμε. Μέσα σε πνεύμα όμως φιλόδοξο για μια Ευρώπη της έρευνας πιο τολμηρή, πιο ενωμένη αλλά και πιο κοινοτική. Και έτσι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό τις νέες δυνατότητε που προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας και να προαγάγουμε την εμβάθυνση των συγκλήσεων και την κοινή ενδεχομένως αξιοποίηση των, των κοινωνικών ε, και εθνικών πολιτικών έρευνας και πρέπει να επισημάνω βέβαια ότι η συνθήκη της Λισαβόνας όπως πενθύμησε και ο συνάδελφος ε, σημαίνει ότι λαμβάνονται υπόψη και οι ενισχυμένες εξουσίες του Κοινοβουλίου με αμοιβαίο σεβασμό, με διαφάνεια, με συνεργασία και μέσα στην ευθεία γραμμή της προηγούμενης Προεδρίας. Ποια είναι μεγάλη, τα μεγάλα θέματα που θα εξετάσουμε. Καταρχάς η στρατηγική 2020 στο προσεχές εξάμεινο δεν προβλέπεται νομοθετική ε, πρόταση στην έρευνα πλην κάποιων ενδεχομένων διεθνών συμφωνιών. Οι προτάσεις Bonus και GMES ολοκλήρωσαν την νομοθετική τους πορεία κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας. Πλην όμως η Βελγική Προεδρία έχει υπόψη μια σειρά από μίζωνα ε, θέματα να εκκινήσει, εκ των οποίων το πρώτο θα είναι η Στρατηγική Ευρώπη 2020 και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συνομβουλίου να ε, ε, ενσκύψει το Δεκέμβριο του 2010 στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Και πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία, μια ευκαιρία που θα πρέπει να δράξουμε καθώς ναι βεβαίως το Συμβούλιο πρέπει εξάπαντος να λάβει κάθε απαραίτητη απόφαση για την οικονομική διακυβέρνηση και την σταθεροποίηση των δημοσιονομικών, πλην όμως επίσης ουσιαστική σημασία είναι να προσδιορίσει και τις προτεραιότητες και τα περιθώρια που ε, μπορούν να διατεθούν στους τομείς που προσφέρουν τις μεγάλες προοπτικές της ανάπτυξης, μέσο και μακροπρόθεσμα. Δηλαδή την επενδύσεις για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία και φυσικά και το περιβάλλον. Και έτσι θέλουμε να απευθύνουμε ένα σαφές μήνυμα, ένα ηχηρό μήνυμα για την έρευνα και την καινοτομία απευθυνόμενο προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ταυτόχρονα για να υπενθυμίσω και τον συνάδελφο το ε, μήνυμα είναι κοινό τόσο για την έρευνα όσο και για την βιομηχανία. Εξού και η άτυπη σύνοδος για την ανταγωνιστικότητα που θα έχει όχι μόνο μία πτυχή έρευνα αλλά και μία πτυχή έρευνα και πλέον αυτόν ε, έρευνα και βιομηχανία αφετέρου, αλλά πέραν αυτών θα έχει και μια κοινή πτυχή έρευνα και πλεον αυτων ερευνα και βιομηχανια φετερου αλλα περαν αυτων θα εχει και μια κοινη πτυχη ερευνα και καινοτομια για να συστήσουμε ακριβώ τα ζητήματα τη καινοτομία επί τη ευκαιρία αυτή. Έτσι λοιπόν και παρά την έκθεση, παρά την αναβολή μάλλον της έκθεσης, ή μάλλον τη συζήτηση στο Συμβούλιο ε, από τον Οκτώβριο στο Δεκέμβριο των θεμάτων αυτών, είναι απαραίτητο η Επιτροπή να διατηρήσει για το Σεπτέμβριο του 2010 στο πρόγραμμά της, όπως άλλωστε είχε προδιαγράψει, την έκδοση του σχεδίου για την έρευνα και την καινοτομία, που θα μας επιτρέψει να έχουμε μια πρώτη, ανταγω... μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων κατά το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις 5 στις 12 Οκτωβρίου και μετά για τις 26 Νοεμβρίου το ίδιο να συστήσουμε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας αυτή τη φορά με συμπεράσματα τα οποία θα διαβαστούν στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Χωρίς να μπορώ βέβαια να προδικάσω τις συζητήσεις, τα μηνύματα που σκοπεύουμε να μεταφέρουμε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι δύο τύπων. Πρώτα απ' όλα ένα πολιτικό μήνυμα, δηλαδή επιβεβαίωση, επαναδιατύπωση της σημασίας, όχι μόνο παρά την κρίση, αλλά κυρίως λόγω της κρίσης, τις σημασίες λοιπόν που αποδίνουμε στην έρευνα και την καινοτομία, το 3% το οποίο παραμένει απαραίτητο λόγω αυτής της δυνατότητας που έχει να κινητοποιήσει πόρους γνώσης και αποτέλεσμα και για την περίοδο 2006-2008, περίοδο που έχουμε, όπου έχουμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία, βλέπουμε ότι 18 κράτη-μέλη εκ των 27 ενίσχυσαν την ένταση έρευνας και ανάπτυξης που προσφέρουν. Πλην όμως αυτό το 3% θα πρέπει να συμπληρώνεται και από μια πιο ποιοτική προσέγγιση, δηλαδή στόχους αποτελέσματος και συμπληρωματικούς δείκτες. Και δεύτερος τύπος, βέβαια, το μήνυμα ότι πρέπει να διαρθρωθεί η έρευνα και ο οικονομικός αντίκτυπος και ο κοινωνικός της αντίκτυπος σε μια προσέγγιση ολοκληρωμένη με την καινοτομία. Και τρίτο τύπο, ενίσχυση τη σύγκληση των πολιτικών τη έρευνα και κοινοτομία στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο πολιτικό μήνυμα είναι ότι επιδιώκουμε μια πρώτη συμφωνία μεταξύ των Υπουργών για πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που θα περιλαμβάνονται στο σχέδιο και που σκοπεύουμε να θέσουμε σε εφαρμογή κατά προτεραιότητα. Δεύτερος μεγάλος φάκελος, θέμα της Προεδρίας μας είναι ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας με αρκετές πρωτοβουλίες που σκοπεύουμε να αναλάβουμε. Καταρχάς μια διάσκεψη προς την κινητικότητα των ερευνητών, διάσκεψη για τον κοινό προγραμματισμό, μάλιστα με πρωτοβουλία της ε, περιφέρειας της Βαλωνίας, μια διάσκεψη ε, για το ρόλο των πανεπιστημίων και των κέντρων έρευνα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνα. Γνωρίζετε φυσικά ποιο είναι ο στόχο που εξυπηρετεί ο κοινό προγραμματισμό. Είναι δηλαδή να μην γίνεται περιττή επικάλυψη προσπαθειών των κυβερνήσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη εν ώψη των μεγάλων προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στον τομέα αυτό, δεδομένου ότι μόλις ξεκινούν οι εργασίες για τους τέσσερις πρώτους θεματικούς τομείς, η Βελγική Προεδρία θα επικεντρωθεί κυρίως στις συνθήκες πλαίσιο του κοινού προγραμματισμού. Επίσης, κατά τη του προσεχού εξαμήνου, η Επιτροπή είχε εξαγγείλει την ενδιάμεση αξιολόγηση του Εβδομού προγράμματος πλαίσιου και την ε, υποβολή της έκθεσης από το Στρατηγικό Φόρουμ για την Επιστημονική και Τεχνική ε, Συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, το ΣΦΙΚ. Εν, όψη ε, και αναλόγως με την πρόοδο λοιπόν κατά την περίοδο αυτή μπορούν να, μπορούμε να συμπεριλάβουμε τα στοιχεία αυτά στα συμπεράσματα μας ή μέσα σε μια έκθεση προόδου για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας στα συμπεράσματα που, όπως έλεγα, θα παρουσιάσουν προς 26 Νοεμβρίου. Επίσης, 26 Νοεμβρίου θα έχουμε μια ε, πρότυπη πρωτοβουλία σε συνεργασία με την Ινδία που θα ασχοληθεί με τις προκλήσεις τις σχετικές με τους υδάτινους πόρους με στόχο ένα καλύτερο συντονισμό των μέσων, των πόρων και των γνώσεων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με την Ινδία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Πολύ σωστά το Κοινοβουλίο σας πάντοτε διατυπώνει το αίτημα της απλούστευσης. Πολλοί είναι οι ερευνητές οι οποίοι περνούν περισσότερο από το μισό του χρόνου τους σε ε, γραφειοκρατικές εργασίες να συμπληρώνουν ε, ερωτηματολόγια, εκθέσεις ε, και άλλα έντυπα. Για τις περιφέρειες επίσης είναι πολύ σημαντικός ο στόχος της απλούστευσης γιατί οι περιφέρειες έχουν και τη μεγαλύτερη εκείτητα είτε με τον ερευνητή, είτε με το ερευνητικό κέντρο, το πανεπιστήμιο ή τη μικρομεσαία επιχείρηση. Έτσι λοιπόν πρέπει αυτά τα προγράμματα να είναι πραγματικά προσβάσιμα και καθώς η συμμετοχή του, κόσμου, του χώρου της βιομηχανίας ε, στα προγράμματα αυτά είναι μάλλον, ε, έχει μάλλον μειωτική τάση, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει το επίπεδο αυτό να είναι στο δυνατόν πιο απλό. Η επλούστευση λοιπόν αυτή είναι απαραίτητη για να ενισχυθούν οι συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των σχεδίων που χρηματοδοτούνται υπό την έρευνα και των άλλων που χρηματοδοτούνται από τα διευθυντικά ταμεία. Εγώ προσωπικώς θέλω να συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στον σκοπό αυτό. Και γι' αυτό βεβαίως πάντοτε και προσκαλούμε τον πρόεδρο της Επιτροπής σας στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών με κύριο θέμα την απλούστευση στην ημερήσια διάταξη. Τον ε, Μάιο επίσης είχαμε μια ανακοίνωση επιτροπής ε, όπου ενέκρινε το Συμβούλιο ένα πρώτο σύνολο συμπερασμάτων με γενικές κατευθύνσεις ε, στο στόχο της απλούστευσης και επίσης σε μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την ε, τριετή αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, καθώς και με μια πρόταση σχετική με το περιθώριο σφάλματος που μπορεί να είναι αποδεκτό. Η Προεδρία μας σκοπεύει να προχωρήσει το περισσότερο δυνατό στον τομέα της απλούστευσης. Η μεγάλη πρόκληση είναι ότι πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στον ερευνητή και ότι πρέπει να βρούμε μια λεπτή ισορροπία μεταξύ του, της εμπιστοσύνης αυτής στον ερευνητή και της αξιοποίησης των δημόσιων πόρων. Λοιπόν, και μία από τις προσεγγίσεις που θέλουμε να ακολουθήσουμε είναι να περάσουμε από την προσέγγιση που ακολουθούμε τώρα με βάση το κόστος σε μία προσέγγιση που θα βασίζεται στα αποτελέσματα. Θα πρέπει ε, να γνωρίζουμε για ποια αποτελέσματα συζητούμε, διότι η έρευνα περιέχει πάντα ένα κομμάτι κινδύνου και αβεβαιότητας. Υπάρχει σειρά άλλων θεμάτων, κύριε Πρόεδρε, που θα εξεταστούν επί Βελικής Προεδρίας. Θα γίνει ένα συνέδριο τον Νοέμβριο. Θέλουμε να δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή στο Συμβούλιο αυτό για το διάστημα. Θέλουμε την έρευνα του διαστήματος, ε, δημιουργήσουμε χώρα ασφαλείας, ε, περιφερειακή διάσταση. Όλα αυτά θα συμπεριληφθούν στα προγράμματά μας, καθώς και το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης θα αντιμετωπιστεί ε, εγκάρσια, διότι θα είναι παρόν θέμα στη δική του 2020, στο πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία και στις προτεραιότητες του κοινού προγραμματισμού. Αλλά δεν θα αντιμετωπιστεί μόνο εγκάρσια, αλλά θα εξεταστούν πολλές πτυχές αυτού του θέματος, καθώς και το πρόγραμμα ΣΕΤ, στρατηγικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κρατών μελών για τις ενεργειακές τεχνολογίες, ούτως ώστε να επιταχυνθεί η έρευνα στις τεχνολογίες ε, χαμηλή παραγωγή διοξιδίου του που θα είναι στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Συνόδου κορυφής των Ενεργειακών Τεχνολογιών. Μία διάσκεψη όσον αφορά την θαλάσσια ε, έρευνα καθώς και η βιοπικιλότητα και μια σειρά εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν επί της Βελγικής Προεδρίας. Ιδού κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, βουλευτές, πολύ συχνά στιγματίζονται οι αδυναμίες οι οποίες υπάρχουν στην Ευρώπη όσον αφορά την έρευνα. Αυτές οι αδυναμίες όμως είναι γνωστές. Κατακαιρματισμός, η διάχυση και άχρηστος ανταγωνισμός μεταξύ χωρών, έλλειψη ερευνητών και εξειδικευμένου προσωπικού ε, έλλειψη κεφαλαίων κινδύνου, κενά όσον αφορά τι άδειε ευρεσιτεχνία, Όλα αυτά θα πρέπει να τα επεξεργαστούμε και θα προσπαθήσουμε να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας το επόμενο εξάμεινο. Όμως θα πρέπει και οι Ευρωπαίοι να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση και ίσως να είναι περισσότερο υπερήφανοι για τα ισχυρά του σημεία. Έχουμε τα πιο μεγάλα ερευνητικά προγράμματα στον κόσμο που επίσης είναι τα πιο ανοιχτά όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία με τους εξωτερικούς μας εταίρους. Είμαστε ο γεωπολιτικός χώρος ο πιο απαιτητικός στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος. Μακράν είμαστε οι πρώτοι ε, δανειοδότες όσον αφορά τη συνεργασία και την ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένου και του μοιράσματο του βάρους ε, με τους πιο στερημένους και να τους δίνουμε δυνατότητες όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα. Είμαστε ο χώρος που επενδύει περισσότερο στην πολιτισμική ποικιλομορφία και τη γλωσσική ποικιλομορφία, ε, κάτι που οδηγεί στην αξιοποίηση της κληρονομιάς μας. Περισσότερη εμπιστοσύνη χρειάζεται στις δυνάμεις μας και βούληση να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες η Ευρώπη χρειάζεται να αναπτύξει μεγαλύτερη νοοτροπία ε, καινοτομίας, αλλαγής κινδύνου. Ε, είμαι πεπισμένος ότι αυτό είναι απαραίτητο για να βγούμε από την κρίση εκ των άνω και δεν είναι μόνο εκείνοι που παίρνουν τις αποφάσεις που πρέπει να πείθουν, αλλά και η κοινή γνώμη εν γέννη και οι νέοι ιδιαίτερα. Όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο σημείο, όπως και τα άλλα σημεία, είμαι πεπισμένος ότι μαζί μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Σας ευχαριστώ την προσοχή σας. Ευχαριστώ θερμά κύριε Υπουργέ. Ας δούμε τώρα και τους δύο φυσικά υπουργού ευχαριστώ. Έχουμε 12 συναδέλφους το λόγο. Για να μπορέσουμε λοιπόν να μιλήσουμε όλοι, πρέπει να περιοριστεί ο καθένας σε ένα λεπτό. Παρακαλώ. Θα είμαι πολύ αυστηρός. Διαφορετικά θα μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε όλου. Η κυρία Φον παρακαλώ να δώσει το καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα λεπτό δεν είναι αρκετό, αλλά παρόλα αυτά να ευχαριστήσω τους δύο υπουργού που ήρθαν στη συνεδριασή μας. Συγχαρητήρια στην Προεδρία, γιατί ήρθαν δύο περιφερειακοί υπουργοί. Ε, θα σας στηρίξουμε για τη λίγη ώρα που έχουμε. Θα πρέπει εδώ να συζητήσουμε για την βιομηχανική πολιτική. Με μας τα είπατε. Αλλά ο Πρωθυπουργό ε, Λετέρ μίλησε και αυτό σχετικά με αυτό στο Στασβούργο την περσμένη εβδομάδα και επομένω πάρα πολύ καλά ε, έχει συλληφθεί το θέμα ότι είναι δυνατόν να προχωρήσει η κοινωνία όπως να υπάρχει μια βιομηχανική βάση γερή και επομένως να κάτσουμε και να δούμε τι είδου βιομηχανικό ιστό θέλουμε να φτιάξουμε, αυτό να συζητήσουμε. επομένω. αυτά που σα ρωτώ είναι να μου εξηγήσετε πώς ο ισχυρό βιομηχανικό ιστό ε, συμβαδίζει με την ισχυρή ε, περιβαλλοντική πολιτική. Ε, και αυτό θα σας είναι η δεύτερη ερώτησή μου. Πετε μας κύριε Υπουργέ, τι νομίζω ότι μπορεί να γίνει στην βραχία περίοδο που έχετε για την ε, Προεδρία σας. Επόμενος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Λάμπερτς. Τα ξέρετε, ήσασταν εδώ πρόσφατα, αγαπητέ συμπατριώτα. Θέλουμε μία γερή η βάση, γιατί δεν υπάρχει ευρωπαϊκή οικονομία χωρίς αυτό. Θέλουμε ανταγωνιστικότητα προς τα έξω, αλλά κατά καλά μας λέτε ότι η ανταγωνιστικότητα θα αφορά όχι το κόστος, γιατί εκεί χάνουμε, αλλά στην προσθέμενη αξία, στην, στην ποιότητα. Άρα θέλουμε αποτελεσματικότητα, ενεργειακή και όπως το κύριε Σερέξ, μια οικονομία η οποία να βασίζεται στην εκμετάλλευση των ε, πόρων. Τέτοια βιομηχανία που θέλετε να χτίσετε και η ερωτήση μου είναι η εξή. Πρώτον, σήμερα έχουμε κάποιε επιχειρήσει οι οποίε ε, λένε ότι το πλήν 20% ε, για τι εκπομπέ είναι πάρα πολύ βαρύ. Αφήστε με ήσυχο, δεν γίνεται αυτό, δεν μπορεί να μα ενταγωνιστεί και από την άλλη μεριά. Έχουμε κάποιε ευρωπαϊκέ επιχειρήσει μικρές μεγάλε που λένε ότι πρέπει να έχουμε κάποιε πιο φιλόδοξε κάποιο πιο, πιο φιλόδοξους κανόνες για πάμε για, για, ακόμα και σε ένα πλήν 30%. Τι λέτε. Και προσπαθούν αυτές οι εταιρείε να ωφεληθούν από τα έξοδα αυτά που κάνουν για το περιβάλλον. Κυρία Gutierrez, έχετε ένα λεπτό. Τι να σας πω στην ε, λεπτάκι, γιατί ε, ε, έχουμε διπλή γλώσσα. Από τη μια μεριά έχουμε τη γλώσσα του ρεαλισμού, για την άλλη της, του, του, ιδιατού και του βολονταρισμού. Τι γίνεται με αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο. Έχουμε ένα σωρό λεφτά που πάνε σε, στις μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουμε 3.300.000 ευρώ το οποίο πάνε σε μεγάλες επιχειρήσεις και από την άλλη μεριά έχουμε και, και, και τους υπόλοιπους. Παρά την πρόταση της Κομισιόν, σε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις έχουμε αντίθετη πολιτική. Δεν μπορούν οι μικρές επιχειρήσεις να συνεχίσουν το πρόγραμμά τους. Αυτές οι ενισχύσεις πάνε μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις και έτσι ούτε στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις ούτε την πανεπιστημιακή παιδεία. Danke sehr, Monsieur Jadot. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κ. Μακόρ και ο κ. Σερέξ, αναφερθήκατε στη διαφάνεια, αναφερθήκατε στις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα θέμα σας δυσαρεστεί και δεν το αναφέρω. Το θέμα ΙΤΕΡ σαν, σαν αφεντικά της Ευρώπης σήμερα υπάρχει ένα συμβούλιο το οποίο σήμερα χωρίς συζήτηση θετήσει κάποια ευρωπαϊκή θέση όσον αφορά τη χρηματοδότηση του ΙΤΕΡ στο τελευταίο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα δεν επετέφθη συμφωνία. Έχω δύο ερωτήσει λοιπόν να σα θέσω. Πώ τέλο Ιουλίου θα πάτε στο Καταρά στο Συμβούλιο ΙΤΕΡ με του Ιαπωνέζου, Αμερικανού και του άλλου και θα πείτε ότι τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να ρίξουν ευρώ στο τραπέζι και ότι αυτό το μεγάλο πρόγραμμα που όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν να υλοποιηθεί προς το τέλος του αιώνα όπου κανονικά θα έπρεπε να δοθούν 4 με 5 δισεκατομμύρια από την Ευρώπη. Ποια αξιόπιστη θέση μπορεί να κρατήσετε στο Συμβούλιο ΙΤΕΡ επ' αυτού του θέματο. Πώ μπορείτε να το προασπιστείτε αυτό έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σαν θέση και έναντι των Ευρωπαίων πολιτών. Παντού γίνονται περικοπέ όσον αφορά τι δαπάνε του ε, προπολογισμού εκτό από ένα πρόγραμμα το οποίο δεν ξέρουμε πότε θα υλοποιηθεί και πόσα ακριβώς, ποια ακριβώ είναι τα προγράμματα. Κύριοι Υπουργοί, ε, εξετίμησα δεόντως και τις δύο παρεμβάσεις και ιδίως ότι δώσατε σημασία ιδιαίτερη στη βιομηχανία. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ήπειρός μας περνάει με περίοδο από αποβιομηχανοποίησης. Μέσω μακροπρόθεσμα ξέρουμε τις λύσεις. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσης και το 2020. Αλλά μέσω μακροπρόθεσμα κινδυνεύουμε τελικά να μην μπορούμε να κινηθούμε, διότι η αποβιομηχανοποίηση προχωρά πολύ γρήγορα. Τι προτίθεστε να κάνετε για να καταπολεμήσετε κάθε μορφή dumping που είναι θύμα αυτής, του dumping η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέτω το συγκεκριμένο ερώτημα, διότι θίγει το θέμα. Όσον αφορά την, τα οικολογικά ζητήματα, είπατε ότι θα πρέπει τις, τους, να κάνουμε τους περιορισμούς περιβαλλοντικούς, να τους κάνουμε δυνατότητα. Αν είναι αποτυχία ξανά η σύνοδος του Κανκούν και τελικά δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, τι θα κάνετε. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε μονομερώς τα αναγκαία μέτρα πιστεύω, αλλά ταυτόχρονα έχουμε δικαίωμα αν δεν μας ακολουθήσουν τα άλλα κράτη που ρηπαίνουν, η και κάποιοι άλλοι, έχουμε δικαίωμα εμείς να επιβάλλουμε μια εισφορά για την ενέργεια και το κλίμα για να ε, εξισωθούν οι όροι του ανταγωνισμού. Τι σκέφτεστε εσείς για άμυνα έναντι αυτής της μορφής ε, του ντόμπινγκ. Εγώ ανέφερα μόνο μερικούς, αλλά υπάρχουν βέβαια και άλλοι. Ο κύριος Λάγκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, και εγώ θεωρώ πολύ θετικό το ότι η βιομηχανική πολιτική και η πολιτική για την καινοτομία είναι στο επίκεντρο της Προεδρία σα. Δύο ερωτήσει. Η βιομηχανική πολιτική έχει διάφορους παράγοντες μέσα της. Έχει δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη κτλ. Πώς σκοπεύετε να εξασφαλίσετε μια κοινή πορεία της βιομηχανικής πολιτικής. Φερρυπίν, στο άρθρο 173 βλέπετε τη δυνατότητα ενδεχομένω να την ενεργοποιήσετε έτσι ώστε να βοηθήσετε στην ανάπτυξη μιας κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής βιομηχανικής ή πώς θα πείσετε τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν μια κοινή γραμμή. Δεύτερον, για την ε, ερευνητική πολιτική. Πολύ καλά ε, το ότι, πολύ θετικό βρίσκω το ότι προσανατολίζετε προς το στόχο του 3% και ότι θέλετε να ε, ενισχύσετε τις αλυσίδες της καινοτομία. Πολύ καλά όλα αυτά, αλλά στο προσεχή προϋπολογισμό, από ό,τι φαίνεται το Συμβούλιο, σκοπεύει να περικόψει τις δαπάνες για την έρευνα και τεχνολογία. Όλα αυτά πώς συνάδουν με τις περικοπές. Δύσκολο είναι να συζητήσουμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, σε ένα λεπτό. Δεν μπορούμε να προβάλλουμε ορθολογικές σκέψεις, όμως έχω μια ερώτηση που είναι απλή. Ε, όσον αφορά τη βιομηχανική και οικονομική στρατηγική για την ανάπτυξη κλπ. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, το πρόβλημά μας είναι η ανεργία και γίνεται μια κοινωνική σύγκρουση, γίνεται κοινωνικό πρόβλημα. Εγώ δεν ακούω στο σύντομο αυτό χρόνο τον συνάδελφο Βέμπερ που μίλησε προηγουμένω, δεν, δεν ακούω τι, κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες θα εφαρμοστούν ε, σε αυτό το τομέα, όπως διαφορετική πολιτική οικονομική του προπολογισμού, ε, τι γίνεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά τα, τη στρατηγική που θα εφαρμοστεί. στρατηγική καλή, κάνουμε βήματα προς τα πίσω και ας εφαρμόσουμε όμως ε, κάτι αμέσως. Τώρα. Ο Καρβάλιο. Ο κ. Καρβάλιο. κυρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Υπουργή. Σαν εισηγήτρια για την έκθεση περί απλούστευσης παραδέχομαι την προτεραιότητα που δίνει η, Ευρωπαϊκή, η Βελική Προεδρία. Θεωρείτε ότι θα συζητηθεί την Τετάρτη σε διάσκεψη που διοργανώνει η Βική Προεδρία Επλούστευση, όπου εκεί έχω προσκληθεί να παρουσιάσω τις βασικές ιδέες της ε, έκθεσης. Μοιράζομαι, συμμερίζομαι, κύριε Υπουργέ, τις ανησυχίες που εκφράσατε, την ανάγκη για την προσέγγιση που θα βασίσει τα αποτελέσματα και πώ θα ακολουθηθεί αυτή που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειαζόμαστε διευκρινήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την έννοια αυτή που θέλει να χρησιμοποιήσει. Η απλούστευση είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους τους ε, τομείς. Όμως, βασικά, αν θέλει κανείς να δημιουργήσει αποτελεσματική και ανοιχτή Ευρώπη και ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, η απλούστευση είναι ύψης της ε, σημασίας. Αναφέρατε και είπατε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες που σας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας για να δημιουργήσετε τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Θα σας ρωτήσω, Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που προβλέπετε μέσω του κοινού προγραμματισμού θα χρησιμοποιήσετε κοινού φορείς, θα χρησιμοποιηθεί και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας για να συνενωθούν τα προγράμματα 100 μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιες είναι οι πραγματικές ρεαλιστικές ιδέες που έχετε υπόψη σας διότι αναφέρατε πολλά ρεαλιστικά προγράμματα και κατά τη διάρκεια των λίγων ημερών της Προεδρίας σας. Σας ευχαριστώ. κυρία Χέρτσοκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε ε, Υπουργέ. Σ' άκουσα και συμφωνώ με αυτό που είπατε, αλλά όταν διαβάζω τα συμπεράσματα του, ε, Συμβουλίου γενικά και ιδίω του ΕΚΟΦΗΝ που θέλει να κόψει 800 τόσα εκατομμύρια, ε, τι γίνεται. Εδώ θέλουμε το αντίθετο, θέλουμε αύξηση σήμερα στην Λισαβόνα και σα ρωτώ το εξή. Τι θα πρέπει να κάνουμε ούτως ώστε το Συμβούλιο των Αρμοδίων την ανταγωνιστικότητα να σταματήσει να, να έχει αυτή την οτροπία τόσο συντηρητική και στενή του ΕΚΟΦΗΝ. Μεσάρος. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ και εγώ και να καλωσορίσω τους δύο υπουργού και να κάνω τις ερωτήσεις μου για την ε, έρευνα. Μόλις είδαμε την ε, αξιολόγηση του 7ου προγράμματος έρευνας, διάμεση αξιολόγηση και βέβαια μας δίνει και κάποια ιδέα για το 8ο πρόγραμμα. Άκουσα λοιπόν τις παρατηρήσεις σας, οι οποίες σε έναν βαθμό περιλαμβάνουν και κάποιες επικρίσεις. Εσείς λοιπόν για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο βλέπετε περιθώριο βελτίωσης και τι για την έρευνα, την ε, καινοτομία, ιδιαίτερα την ανάπτυξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς μπορούμε να τις εμπλέξουμε στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Έχουμε προγράμματα πολύ σημαντικά για την έρευνα και την καινοτομία που στόχο έχουν να διαφυλάξουν την πρωτοπορία της Ευρώπης. Μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες αυτές. Ευχαριστώ. Μπέλετ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στους δύο υπουργούς της Βελικής Προεδρίας, καλωσορίζω. Καταρχάς, για τον κύριο Μαχκούχ. Συνεχίζεται, κύριο Υπουργέ, μετά την Ισπανική Προεδρία, η οποία επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην ε, ενέργεια, την προαγωγή νέων τεχνολογιών και κυρίως τα ε, την ανάπτυξη της ηλεκτρικής τεχνολογίας στα, στην βιομηχανία Έχετε στις αντίστοιχες ε, προθέσεις, θα συνεχίσετε τις προσπάθειες αυτές ε, και τις πρωτοβουλίες της Ισπανικής Προεδρίας, γιατί αν είναι έτσι βεβαίως θα σας υποστηρίσουμε 100%. Επίσης για τον κύριο Σερέξ, είπατε ότι χρειάζεται και περισσότερο συντονισμό συνεργασία από πλευράς των κρατών μελών για να διαφυλαχθεί και να τηρηθεί το όριο του 3% για την έρευνα αν κατάλαβα καλά από τα όσα είπατε, θέλετε ω Υπουργή Καιροτομία να αποστείλετε σαφή μηνύματα για το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Έχετε κάτι πιο συγκεκριμένο να μα πείτε, γιατί και πάλι και εδώ θα σα στηρίξουμε. Ευχαριστώ, κύριε Σουκαλά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τους δύο κυρίους Υπουργούς για τις πολύ χρήσιμες εισηγήσεις τους. Είμαι πολύ χαρούμενος ότι στην Επιτροπή μας Όλα ένα και συχνότερα γίνονται συζητήσεις για την έρευνα και την τεχνολογία. Άκουσα τις παρατηρήσεις του Δευτέρου των εισηγητών. Ε, φυσικά και ελπίζω και εγώ ότι θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Όμως παρά τα αυτά πρέπει να τον ειδοποιήσω ότι υπάρχει μια αυξημένη δυσπιστία σε σχέση με το εάν η Ευρώπη με την στρατηγική του 2020 θα έχει καλύτερη τύχη από την στρατηγική της Λισαβόνας. Και μολονότι υπήρξαν κράτη-μέλη που χρησιμοποίησαν αυτή τη στρατηγική πάρα πολύ αποτελεσματικά και με πολύ καλά αποτελέσματα, οι μέση, ώρες, οι μέση όροι και οι τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό εξακολουθούν να είναι ποσοτικά και ποιοτικά κατώτερες του αναμενωμένου. Σχετικά με αυτό υπάρχουν προτάσεις να ακούσουμε. Ακόμα δύο συνάδελφοι έχουν στήσει το λόγο. Έντσου και Τσίκαου. Ε, ε, παρακαλώ όμως πολύ στόμα γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους δύο προσκεκλημένους υπουργού για την παρουσίαση του προγραμματός τους και των στόχων της Βελικής Προεδρίας. για, την επόμενη, για το επόμενο εξάμεινο στους τομείς της έρευνας και της ε, καινοτομίας. Πιστεύω ότι θα επιτύχει το στόχο της, ε, του επαναπροσδιορισμού των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη η Βελική Προεδρία. Για, του, για τα νέα κράτη-μέρη λοιπόν, Θέλω να ρωτήσω αν έχετε κάποια συγκεκριμένα σχέδια, γιατί ξέρουμε ότι έχουν ιδιαίτερε ελλείψει στι υποδομέ τα νέα κρατημέλη. Κυρία Τσίκαο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ να ευχαριστήσω του ε, υπουργού που ήρθαν εδώ για να συζητήσουμε, για να μα παρουσιάσουν το πρόγραμμα τη Βελγική Προεδρία. Θα ήθελα τώρα να συνεχίσω στην μητρική μου γλώσσα, που την αγαπώ τόσο πολύ. Η ερώτηση λοιπόν που θέλω να κάνω εγώ έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό σχέδιο για τις οικονομικές συνεργασίες. Ένα σχέδιο το οποίο μας είχε υποβάλει αρχικά, αρχικά με μια ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία μεταξύ του τομέα της έρευνας, της ενέργειας κτλ. Που όμως δεν, ήταν δεν είδανε συγκεκριμένη υλοποίηση. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει αυτή η οικονομική στήριξη και η συνεργασία, πώς μπορούμε να περιμένουμε ανάπτυξη οικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Οι δύο υπουργοί τώρα έχουν την ευκαιρία να δώσουν σύντομες και συγκεκριμένες απαντήσεις και πάλι παρακαλώ να περιοριστείτε ο καθένας σε μερικά λεπτά, δύο-τρία λεπτά. Κύριε Μαχκούχ, παρακαλώ εσείς πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τη βιομηχανία. Θα ήθελα να ανταποκριθώ στις ευχές του Προέδρου και να είμαι συνθετικό, συνοπτικό. Να πω ότι πρώτα απ' όλα στη συνάντηση μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Βελική Προεδρία, στου βασικού άξονε που θέλει να αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η βιομηχανική πολιτική είναι κάτι που αναφέρθηκε. Νομίζω ότι εδώ και πέντε χρόνια αυτό το στοιχείο της βιομηχανικής πολιτικής δεν θα αποτελούσε το αντικείμενο συνένεσης τόσο μεγάλης μεταξύ των διαφόρων κλάδων της ενώσεως και αυτό για μένα είναι σημαντικό θέμα. Δηλαδή ότι θεωρούμε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να υπερασπιστεί τη βιομηχανία της. Για να απαντήσω, δεν θα αναφερθώ σε όλους βέβαια, προς την κυρία Βαν Μπρέντ να απαντήσω, είναι σαφές ότι η αλλαγή του κλίματος είναι ένας περιορισμός και μια έξοχη δυνατότητα και ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί για τις επιχειρήσεις, απαντώντας σε άλλους τώρα το λέω αυτό, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί η αλλαγή του κλίματος σαν ένα εμπόδιο για την ανάπτυξη των βιομηχανιών μας, θα πρέπει να δούμε ποιο μονοπάτι θα πρέπει να ακολουθήσουμε και συνοδέσουμε τις βιομηχανίες μας και το κάνουμε αυτό και στη Σύνοδο Κορυφής την ανεπίσημη αυτής εβδομάδας και στο πλαίσιο της διασκέψεως για τις βιομηχανικές αλλαγές που θα λάβει η χώρα επί Βελικής Προεδρίας. Θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις βιομηχανίες μας να αντιμετωπίσουν την αλλαγή του κλίματος, να έχουν σημαντικότερους στόχους, ώστε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Όσον αφορά τις ποσοστώσεις, πάντα ήμουνα πολύ επιφυλακτικό όσον αφορά τι ποσοστώσει διοξιδίου του άνθρακο και του συστήματο που δημιουργήσαμε, ιδιωτικοποίησεω των ποσοστώσεων διοξιδίου του άνθρακο, ενώ θα πρέπει προφανώ να έχουμε ένα στόχο μειώσεω των εκπομπών, λαμβάνοντα υπόψη την εξέλιξη τη τεχνολογία παρακινώντας την χρήση των πλέον οικονομικών ε, τεχνολογιών που θα μειώνεται η κατανάλωση της ενέργειας μέσω αυτών των τεχνολογιών, αλλά αυτό θα πρέπει να ακολουθηθούν, να επιτευχθούν μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων. Θα έχουμε εκεί να το συζητήσουμε. Όσον αφορά το dumping, ε, θέλουμε να αξιολογήσουμε ποια είναι η εξωτερική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αφού αξιολογηθεί αυτή η εξωτερική ανταγωνιστικότητα να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος χωρίς να γίνει να δώσουμε χώρο στους ανταγωνιστές μας να μας αφαιρέσουν μερίδιο της αγοράς. Θέλουμε να παραμείνει η ανταγωνιστικότητά μας κυρίως ε, μέσω της, των εξαγωγών μας. Δηλαδή πετυχαίνοντας τους στόχους που έχουμε θέσει έναντι των ανταγωνιστών μας και έναντι ε, των γενικών εξελίξεων. Είναι σαφές ότι κάθε οικονομική δράση έχει νόημα, κατά την άποψή μου, μόνο αν δημιουργεί θέσει απασχόληση. Αυτό είναι ένα στοιχείο θεμελιώδου σημασία, να υπερασπιστούμε την απασχόληση, να υπερασπίσουμε του τομεί εκεί που δημιουργούν απασχόληση και να του υποστηρίξουμε. Υπάρχει και ανάγκη άμεσων μέτρων, αλλά δεν μπορούμε να καλύψουμε ε, όλο το χρόνο που χάσαμε. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας, να δώσουμε κίνητρα και για να πω ότι δεν έχουμε οικονομική και κοινωνική πολιτική ε, ενιαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να έχουμε πολιτικές συγκλήσεις σε που θα εφαρμόσουμε, ώστε να πλησιάσουν τα κράτη-μέλη και να υπάρχει κοινή βούληση. Αν θα μπορούσαμε να επανεξισορροπήσουμε το Συμβούλιο Βιομηχανίας και να γίνει πολύ σημαντικός χώρος, όπως είναι και το Συμβούλιο για κοινωνικά θέματα και ΕΚΟΦΗΝ, τότε αυτό θα ήταν ωφέλιμο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ήθελα να πω ότι προφανώς και χαιρετίζω εδώ το έργο της Ισπανικής Προεδρίας κατά διάρκεια του πρώτου εξαμήνου όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα θα πρέπει λέγω τα αυτοκίνητα ο αυτοκινητοβιομηχανία που είναι σημαντικός τομέας και θα παραμείνει σημαντικός τομέας αλλά όχι μόνο σαν απλή αυτοκινητοβιομηχανία αλλά σαν ένα τομέα που μπορεί να μειώσει την κατανάλωση της ενέργειας να, να φτιάχνει αυτοκίνητα καθαρά στα πλαίσια λοιπόν της μεταμόρφωσης της βιομηχανίας που εξετάσουμε πώς μπορούμε να αποθηκεύουμε ενέργεια τι γίνεται μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, πώς μπορεί να αποθηκεύεται. Πρέπει να εξεταστεί αυτό. Χαιρετίζω τα όσα έκανε η Ισπανική Προεδρία. Θα συνεχίσουμε και εμείς την ίδια προσέγγιση. Για να αλλάξουν τα αυτοκίνητα. Να γίνουν ηλεκτρικά ή να βρεθούν και άλλες λύσεις. Διότι το Συμβούλιο Βιομηχανία ζήτησε να εξεταστούν όλες οι λύσεις. Το 2011 θα πρέπει να υπάρξει μια τυποποίηση όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων για να προσαρμοστεί δεόντως η Ευρώπη. Θα απαντήσω και σε άλλες ερωτήσεις αν τυχόν υπάρξουν ή το επιθυμείτε. Αυτά είχα να πω μέχρι τώρα. Ε, Ευχαριστώ θερμά τον ε, Υπουργό κ. Μαρκούρ για την πολύ σύντομη και σαφή του απάντηση. Και τώρα ο κ. Ε, Σέαξ παρακαλώ. Προσπαθήσω πρόεδρε να σας το πω όσο κρατεί ο συνάδελφος Μαρκούρ όσον αφορά τις ΜΜΕ και το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο όντως η συμμετοχή των ΜΜΕ έχει μειωθεί και ε, να, δούμε γιατί το θέμα της συμμετοχής αυτού του 15% ΜΜΕ είναι κάτι το οποίο ως στόχο δεν το πιάσαμε και τελικά ε, χρειάζεται να έχουν περισσότερη απλούστευση, απλούστευση ε, να μειωθούν τα κονσόρτσια, να μειωθούν οι, οι ομαδοποιήσεις και αυτό και θα μας απασχολήσει. Τώρα, όσον αφορά το ΙΤΕΡ γνωρίζετε ότι το Συμβούλιο Βιομηχανής και Ανταγωνιστικότητας είπε ε, τον Ιούνιο ότι δεν αποφασίζει όσον αφορά ε, αυτά που θέλαμε και θα, θα γίνει στο ε, Κάνταρας μία έκτακτη σύνοδος, γιατί θα πρέπει αυτό το Συμβούλιο να καθορίσει μια θέση μέχρι τα τέλη Ιουλίου και κανένα ε, κράτος μέλος σήμερα δεν θέτει να αμφιβόλω αυτό το, το όραμα. Γιατί το θέμα είναι από πλευρά ε, δημοσιονομικής, από πλευράς χρηματολόγησης και έχουμε και την Task Force της Ισπανικής Προεδρίας που ε, ξεκίνησε και συγκροτήθηκε επί τη βάση απόφαση της ε, κορυφές τη 30 Ιουνίου, κατόπιν είχαμε δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι θέμα α ε, του σημερινού Συμβουλίου Γεωργίας. Ε, σημειώθηκε συμφωνία στο Συμβούλιο όσον αφορά την ουδέτερη στάση της Προεδρίας, αλλά θέλουμε να είμαστε εγγυητέ αυτής της θέσης που αποκρισταλώθηκε. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει όλες υπόψη την εμπλοκή που μπορεί να φέρει στην υπόθεση του Κοινοβουλίου. Άρα εμείς θα πρέπει να πασχίσουμε, να βρούμε κάποιο είδους συμβιβασμό και θα πρέπει επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει 100% ε, τη δυνατότητα ε, και αρμοδιότητα υποβολής της ε, πρότασης που έχει τώρα για το κατά πόσον χρειάζεται να έχουμε παραπάνω επενδύσεις για την έρευνα και ε, τι θα γίνει με τις περικοπές στον προπολογισμό. Νομίζω ότι το 3% στόχος δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί εάν δεν έχουμε προσπάθεια από πλευράς προϋπολογισμού. Και να γίνει προσπάθεια και από τα κράτη-μέλη, τις περιφέρειες, τα, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει να πάει αλλού η αυστηρότητα και οι περικοπές. Αλλά επίσης θεωρώ ότι το θέμα δεν είναι το αν κάποιο ε, εκταμιεύει περισσότερα, αλλά πώ χρησιμοποιεί αυτά τα οποία διαθέτει. Και άρα θα πρέπει να βρεθούν κάποιου δείκτε ποιοτικοί. Είναι αυτό κάτι το οποίο σα το εξήγησα προηγουμένω. Τώρα, με την Τετάρτη στο σεμινάριο, όντω, θα δούμε τι γίνεται όσον αφορά την πιστοποίηση. Και όπως σας είπα, θέλουμε να έχουμε μια προσέγγιση βάσει των αποτελεσμάτων αλλά υπάρχουν εδώ πέρα κάποια, ε, κάποια ρίσκα εγγενή όσον αφορά την έρευνα. Θέλουμε να δούμε πώς θα έχουν κινητικότητα οι ερευνητές, πώς θα έχουμε κοινό προγραμματισμό, πώς θα έχουμε διεθνή συνεργασία. Όντως, εγώ επέμεινα όσον αφορά την καινοτομία και όσον αφορά το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να στείλουν οι Υπουργοί Βιομηχανίας και Έρευνας τον Δεκέμβριο με το Συμβούλιο. Από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα πλαίσιο το 1984 η Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Έρευνα έχει ε, οδηγήσει σε καλύτερη γνωριμία και συνεργασία των επιστημόνων στην Ευρώπη. Και σήμερα θα πρέπει να δούμε περισσότερο τι έχουμε όσον αφορά τις εθνικές προσπάθειες ε, συγκεκριμένες προτάσεις να έχουμε που να τεθούν επιτάπητο στο Συμβούλιο και να δούμε τι γίνεται στις προτεραιότητες μας, πρώτα πρώτα με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ε, εταιρική σχέση, ε, τυποποίηση ε, και εν κατακλείδη πρώτα να δούμε τι θα γίνει με τα καινούργια κράτη-μέλη. Γιατί οργανώθηκε εκείνη η συνάντηση υπό την Ισπανική Προεδρία στην Ισπανία. Εκεί κάναμε βήματα πρόοδου για να αναδείξουμε το πόσο χρειάζεται να υπάρχει καλύτερη συνέργεια μεταξύ έρευνας, πολιτικής συνοχής και της περιφερειακής διάστασης. Για τη στρατηγική του 2020 θέλουμε οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές να ασπαστούν αυτή τη στρατηγική αλλά και να την εφαρμόσουν σύμφωνα με την αρχή της επικορικότητας και επίσης να χρησιμοποιήσουν την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο υπουργούς. Ήταν σύντομη, ναι, πολύ σύντομη, αλλά πάντως σαφής νομίζω ξεκάθαρη συζήτηση η πρώτη αυτή επαφή μας. Δυστυχώς όμως ε, είχαμε λίγο χρόνο σήμερα και υποχρεωτικά περιορίσαμε το ε, χρόνο που μπορούσαμε να σας διαθέσουμε. Θα σας ξαναδούμε όμως σύντομα πιστεύω. Καλή αρχή και σας εύχομαι και καλή επιτυχία στη Βελγική Προεδρία. Εμείς θα συνεχίσουμε και με τον επόμενο Υπουργό που θα έρθει να μας επισκεφθεί τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ.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 6, μάλλον 5, προβλέπει την επιχείρηση του κυρίου Πολ Μανιέτ, Υπουργού Κλίματος και Ενεργειακής Πολιτικής, αρμοδίου για την προστασία των καταναλωτών, ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε την ευκαιρία τώρα να ακούσουμε μια σύντομη παρουσίαση από τον κύριο Μανιέτ. Μετά δε θα έχουμε με τις ερωτήσεις και τις ε, την ευκαιρία να εμβαθύνουμε στο θέμα σας. Κύριε Μανιέτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας όπου θα αναφέρουμε τις προτεραιότητες της Βελικής Προεδρίας, της Ευρωπαϊκής Ενώσης στον τομέα της ενέργειας. Είναι στιγμή σημαντική για μένα. Θέλω ειλικρινά να πω ότι περιμένω στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ήδη μπορέσαμε να ξεκινήσουμε συνεργασία, ήδη είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε με τις πολιτικές ομάδες τέλος μηνός Ιουνίου εν την προετοιμασία της αναλήψεως της Προεδρίας. Είχα τη μεγάλη χαρά να μπορέσω να πάω στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα εις για να συζητήσουμε την ασφάλεια των ε, διαφόρων πετρελαϊκών ε, εξορίξεων στη θάλασσα και το φθηνό που το θέμα και θέλω αυτός ο διάλογος να μπορέσει να διατηρηθεί ε, και να είναι εξίσου πλούσιο όπως τώρα που ξεκίνησε. Θα ήθελα να πω ότι οι νέοι κανόνες της συνθήκης της Λισαβόνας οδηγούν σε ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι έχουμε κάποια προηγούμενα γεγονότα που δείχνουν ότι η σχέση μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου μπορεί να είναι εξοχές όπως στην ολοκλήρωση του κανονισμού για το φυσικό αέριο που, θα, που ενεκρίθη με τους καλύτερες δυνατές συνθήκες πρόσφατα. Αυτή η Προεδρία λοιπόν από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να την προετοιμάζουμε με τους Ισπανούς και Ούγγρους φίλους μας ασχολήθηκε με τις εργασίες του Κοινοβουλίου και υποχρεώθηκε να βάζει στην ημερήσια διάταξη διάφορα θέματα που ίσω να μην συμπεριλαμβάνονταν μέχρι τώρα και που αποτέλεσαν αντικείμενο εργασιών και προβληματισμού από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέματα που συνδεόταν όλο ιδιαίτερω με την προστασία των καταναλωτών. Στον τομέα τη ενεργειακή πολιτική, και θα επανέλθω σε αυτό το θέμα σε λίγο. Πριν αναφερθώ στα συγκεκριμένα σημεία, ξεχωριστά σημεία επί των οποίων θα θέλαμε ε, να κινηθούμε ιδιαίτερω ε, σε αυτό το, στην Προεδρία μας, να πω κάτι εν συντομία. Πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η στιγμή στην οποία βρισκόμαστε όσον αφορά την ιστορία της ευρωπαϊκής πολιτικής. Είμαστε λοιπόν δέκα χρόνια μετά την αρχή της απελευθερώσεως του ενεργειακού τομέα και του ανοίγματο της ενεργειακής αγοράς, των ενεργειακών αγορών, όπως θα θυμόσαστε. Μας δόθηκαν πολλές υποσχέσεις όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της απελευθέρωσης ενέργειας. Μας λέγανε ότι αυτό θα οδηγούσε στην τεχνολογία, την καινοτομία, την τεχνολογική, μεγαλύτερο ανταγωνισμό που θα οδηγούσε σε καλύτερες υπηρεσίες, πιο ποιοτικές, χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. Δηλαδή, όπως και σε άλλους τομείς ότι ε, δοθήκανε πάρα πολύ καλές υποσχέσεις σε όλους τους Ευρωπαίους. Όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε χωρίς να θέλουμε λοιπόν να μπούμε σε επίμαχα θέματα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως ότι δεν φτάσαμε εκεί που θα έπρεπε και ότι όλοι οι στόχοι που είχαν τέθει όσον αφορά την πολιτική της απελευθερώσεως δεν επετεύχθησαν. Το επίπεδο της συγκεντρώσεως των αγορών παραμένει ψηλό. Όσον αφορά τους μεγάλους προμηθευτές φυσικού αερίου για 10 κράτη-μέλη οι τρει μεγάλοι προμηθευτέ έχουν πάνω από 90% τη αγορά όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό ο έλεγχο είναι μεγαλύτερο από το 80% σε 14 κράτη-μέλη, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά τη. Η έκθεση του καθηγητού Μόντι όσον αφορά την εσωτερική αγορά δείχνει επίση ότι στον τομέα των ενεργειακό ακόμα πόρο απέχουμε από τη δημιουργία πραγματική εσωτερική αγορά. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει κάποια ορμή ε, όπου μπορούμε να αναλύσουμε πού βρισκόμαστε όσον αφορά την υλοποίηση του τρίτου ενεργειακού πακέτου και κλίματος όταν τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει και κάποιε εθνικέ δράσει όσον αφορά τι ανενώσιμε πηγέ ενέργεια. Υπάρχει λοιπόν κάποια όθηση, παρένεση για να αναλύσουμε αυτή την ενεργειακή αγορά και να διορθώσουμε εκεί που χρειάζονται διορθώσει. Και μετά άλλη σκέψη έτσι ακροθυγό, Ξέρετε ότι η Ευρώπη έχει ηγηθεί όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική και κυρίως το Δεκέμβριο του 2008 υιοθετώντα το πακέτο ενέργεια κλίμα τις παραμονές πολύ σημαντική συνεδριάσεως στο Πόσναν όσον αφορά τις διεθνείς συζητήσεις για το κλίμα έδειξε η Ευρώπη τη βούλησή της να ηγηθεί σε αυτά τα θέματα και να εφαρμόσει μια πολιτική πραγματικά που θα έχει όραμα στον αυτή την ενέργεια. Ποια είναι η ηρωνία τη ιστορία, και υπενθυμίζω για τα γεγονότα, σα το είπα ήδη την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια, ότι τη στιγμή όπου οι Ευρωπαίοι ετοιμάζαν αυτό το πακέτο ενέργεια και το κλίμα που είχε στόχο να μειώσει την κατανάλωση της ενέργειας και να τονώσει πραγματικά, να δώσει ζέση στην ανάπτυξη των νοσημών τεχνολογιών και ενέργειας. Η προηγούμενη Αμερικανική κυβέρνηση ακολούθησε διαφορετική πολιτική γεωτρήσεων πάρα πολύ περιπετειώδη στην Αλάσκα με συνέπειες που ξέρουμε σήμερα. ως φορά τις γεωτρήσεις. Λοιπόν, θέλουμε να ιδρύσουμε αυτό το πνεύμα το οραματικό που είχαμε εδώ και 18 μήνε. Δηλαδή, θέλουμε ένα ευρωπαϊκό όραμα όσον αφορά την ενέργεια, γεμάτο υποσχέσει για την ασφάλεια φωδιασμού, για την ανεξαρτησία μα την ενεργειακή, για τον οικονομικό και βιομηχανικό συγχρονισμό, για τη δημιουργία απασχόληση επίση. Και βεβαίω αυτό το όραμα θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητα από τι χρονικέ πιέσει ή και τα εμπόδια που θα αντιμετωπίσουμε στο μονοπάτι μα. Αυτή είναι, σε αυτή τη φιλοσοφία κινούμεθα σαν Βελική Προεδρία. Διπλή φιλοσοφία να αξιολογήσουμε και να διορθώσουμε τα ελλείψει μέσω της απελευθερώσεως και να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε το ισχυρό μας όραμα όσον αφορά το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης απ' την άλλη. Όλα αυτά προϋποθέτουν καταρχάς κατά την άποψή μας να ασχοληθούμε με το θέμα της καταστάσεις που κρατήσουν όσον αφορά τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Διάβασαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενεπνεύστην από το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σας στις 19 Ιουνίου 2008 όσον αφορά τη Χάρτα των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών. Κάποια στοιχεία μπορούν να επηρεάσουν και τη σύνταξη του τρίτου πακέτου ενέργειας και κλίματος, όπου εκεί βλέπουμε ακόμα και από μετά μερικά χρόνια πολλά απομένουν να γίνουν, κυρίω όσον αφορά το θέμα των τιμών. Από το 2005 μέχρι το 2007 η τιμή του φυσικού για την νοικοκυριά αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 18% σύμφωνα με τη σχέση του Γεροστάτ και τη ηλεκτρική ενέργεια κατά 14% μια συζήτηση όσον αφορά τα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ούτως ώστε να καταστήσουμε την ενεργειακή πολιτική πιο ευνοϊκή για τους καταναλωτές είναι τώρα περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Αυτό προϋποθέτει βεβαίως ενίσχυση των πολιτικών, της πολιτικής ενημέρωσης του καταναλωτού. Αυτό προϋποθέτει και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να συντονίσουμε τις εργασίες των εθνικών διαμεσολαβητών που προσπαθούν να συντονίσουν τους προμηθευτές με τους καταναλωτές και θα πρέπει να ενισχύσουμε με δυναμικό και συνεχή τρόπο τα δικαιώματα των καταναλωτών με αυτό που κάνει και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής με επικοδομητικό τρόπο ε, στη συνεργασία με τους εθνικούς ομολόγους του. Ε, υπό αυτή την οπτική γωνία θέλουμε να εξετάσουμε αυτή την πρόταση οδηγίας που θα δημοσιεύσει το Θηνόπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το wholesale market trading, νέο ρυθμιστικό πλαίσιο ευρωπαϊκό για τις ενεργειακές αγορές χοντρική πωλήσεως, ένα βασικό στοιχείο όσον αφορά έναν αποδοτικό ανταγωνισμό που θα είναι επωφελής προς τους καταναλωτές. Λοιπόν, στο φάσμα του καταναλωτέ, θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή για του καταναλωτέ ευαλώτου, όπω αποκαλούνται, και είναι ένα νέο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σα που μα ενέπνευσε και μα έδωσε τροφή τη 25η ε, Σεπτεμβρίου του 2008 όσον αφορά τον έλεγχο τη κρίσεω. Όσον αφορά την ενεργειακή ανασφάλεια, υπάρχει σήμερα στην, ε, υπάρχουν στην Ευρώπη ανάμεσα στου 50 και 125 εκατομμύρια ε, πολίτε που υποφέρουν από φτώχεια ενεργειακή. Δεν έχουμε καθόλου αυτόν τον όρο, δηλαδή ότι δεν μπορούν να ζεσταθούν επαρκώ και δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους ή πρέπει να δώσουν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός τους για να καλύψουν ενεργειακές τους ανάγκες έστω και στοιχειώδεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε πλέον να αγνοήσουμε και θα πρέπει πάση θυσία να το επιλύσουμε και κυρίως αυτή την Ευρωπαϊκή Χρονιά Καταπολέμησης της Στόχιας το 2010 και αυτή την χρονιά της οικονομικής κρίσης όπου ξέρουμε ότι έχουμε 23 εκατομμύρια άνεργοι που αυξήνουν τον αριθμό των οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ειδικέ δυσκολίες και θέλουμε να αποφύγουμε μεγάλη επιδείνωση του φαινομένου αυτού. Σαν Εθνικό Υπουργό τη Ενέργεια, θέλω να πω ότι αυτά τα θέματα σίγουρα, αυτό το θέμα ήταν ένα από εκείνα που δημιούργησε την ενδελεγέστερη συζήτηση στη χώρα μου και γνωρίζω ότι, διότι έχω συζητήσει με Ευρωπαίου συναδέλφου, ότι η ίδια συζήτηση έχει γίνει και σε πολλά κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και θα γίνει η πρώτη συζήτηση κατά τη διάρκεια του ατύπου συμβουλίου που θα γίνει σε 6 και 7 Σεπτεμβρίου και μετά τα συμπεράσματα του επισήμου συμβουλίου θα είναι έτοιμα το 2 Δεκεμβρίου και θέλουμε να καθορίσουμε ποιο είναι το φαινόμενο αυτό της ανασφάλειας της α, ενεργειακής, να προστατικοποιήσουμε αυτό το φαινόμενο και θέλουμε ένα σύστημα αξιολογήσεως των μέτρων που εφαρμόστηκαν από τα διάφορα κρατημέλη, ανταλλαγή να γίνει των βελτίστων πρακτικών τους ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ένα από τα άλλα σημεία τα οποία θα θέλουμε να συνδέσουμε με την ενεργειακή ανασφάλεια είναι και το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας και πιο συγκεκριμένα στις κατοικίες. Αυτοί οι πολλοί συμπολίτε μα που αντιμετωπίζουν δυσκολίε να θερμανθούν ή να πληρώσουν του λογαριασμού του, πολύ συχνά είναι εκείνοι που ζουν σε ε, παλιά σπίτια. Ξέρετε ότι στην Ευρώπη, στα 27 κράτη-μέλη, 60% των κατοικιών οικοδομήθηκαν χωρί να ληφθεί υπόψη κανένα κριτήριο ε, για την θέρμανση ε, και υπάρχει μόνος πολύ κακή καθόλου μόνος. Οι αυτοί που ζουν εκεί αντιμετωπίζουν πρώτε δυσκολίε και προ αυτού θα πρέπει να κατευθυνθούν οι προσπάθειέ μα και η προσοχή μα. Η ενεργειακή λοιπόν αποδοτικότητα σίγουρα είναι η βασίλισσα των πολιτικών. Κάθε φορά που καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια, είμαστε λιγότερο, λιγότερο ρηπαντές, λιγότερο εξαρτημένοι, λιγότερο υπεύθυνοι για την αύξηση της θερμοκρασία. Αυτό ίσχυε και θα πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα των προτεραιοτήτων. Υπάρχει λοιπόν ακόμα στην Ευρώπη, υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά τη βελτίωση τη αποδοτικότητα. Υπάρχουν πολλέ μελέτε και στη στέγαση και στα δημόσια κτίρια, στη θέρμανση, στι βιομηχανικέ διαδικασίε, στι μεταφορέ. Και η πολιτική μα ευρωπαϊκή στον τομέα κατέδειξε την αποτελεσματικότητά Θυμηθείτε τη συζήτηση καμιά φορά που ήταν δύσκολε ο άφο περιγραφέ για τι εκπομπέ των οχημάτων. Θα θυμηθείτε τι συζητήσει που έγιναν για την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακο και αερίων του θερμοκηπίου. Που Θυμηθείτε αυτή τη συζήτηση. Δύσκολη ήταν. Έγιναν πολλέ αξιολογήσει, τι έχουμε στη διάθεσή μα και δείχνουμε ότι η Ευρώπη σε αυτό το τομέα έκανε πάρα πολλέ πρόοδου και οι Ευρωπαίοι αυτοκινητιστές καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια χάρη σε εξυγχρονισμό των, του στόλου των οχημάτων που είναι κάτι υποφελές και για την αυτοκινητοβιομηχανία μας. Από αυτή την έποψη θα ήθελα να πω με χαρά ότι θα έχετε τη χαρά μάλλον να εθετήσετε τι τέσσερι πρώτε ε, εκχωρηθήσει πράξει όλη τη ιστορία τη Ευρωπαϊκή Ολοκληρώσεω, διότι είναι νέο είδο πράξη που προβλέπεται από τι συνθήκε τη Αβώνα, που ακόμα δεν είχε εφαρμοστεί πλήρω και θα προτείνει κατά διάρκεια του θέλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτω ώστε το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να, ε, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τοποθετηθούν και να γνωμοδοτήσουν και να προωθηθούν αυτέ οι κορυφήσει πράξει όσον αφορά την κοιτοθεσία των προϊόντων όπω τα ψυγεία, οι τηλεοράσει ε, κλπ. Αυτό είναι ένα πρώτο στάδιο που θα κάνουμε με τις συνεργασίες της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Το Συμβούλιο περιμένει Όπω και το Κοινοβούλιο, τα πρώτα στοιχεία αξιολογήσεω του σχεδίου δράση όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, ούτω ώστε να διεξαχθεί στι 6 και 7 Σεπτεμβρίου στο Άτυπο Συμβούλιο με πρώτα συζήτηση. Συζήτηση που θα πρέπει να τροφοδοτήσει τη δημιουργία του σχεδίου δράση όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα που θα ακολουθήσει. Κάποια λόγια για να κλείσω όσον αφορά τι επενδύσει, διότι στο Συμβούλιο συζητήσει που διεξήχθησαν πρόσφατα, όσον αφορά τι έξοχε συζητήσει που έγιναν επί Ισπανική Προεδρία, πρέπει να πω ότι είναι ένα θέμα που το συζητήσαμε εκτενώ, το συζητήσαμε πάρα πολύ, διότι είναι επίκαιρο, οι επενδύσεις, πάρα πολλές επενδύσεις χρειάζονται όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση για τις μεταφορές, για την διανομή, για τον εξυγχρονισμό των δικτύων και για, τα, για τους μετρητές, για την ίδια την παραγωγή. Για να έχουμε δυνατότητες παραγωγής πιο καθαρής υπάρχουν και άλλες περιοχές του κόσμου που παράγουν απορριχτά καύσιμα, ενέργεια που είναι απαραίτητη για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζονται κολοσσίες επενδύσεις στους τομείς αυτούς τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη δεκαετία, χωρίς να μετρήσουμε τα 75 με 80 δισεκατομμύρια ευρώ που χρειάζονται για την έρευνα και την ανάπτυξη, κάτι που καθορίσαμε στο 7 ε, ε, ε, προ, άξονες προτεραιότητες. Λοιπόν, στα πλαίσια του προγράμματος της ενέργειας για επαναπρόθεση οικονομίας, το Recovery Plan, της ενέργειας και εκεί μπορέσαμε να εντάξουμε μια ουσιαστική, μια σημαντική ενεργειακή πτυχή. 4 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις δόθηκαν τότε Ξέρουμε και ξέρετε καλύτερα από μένα ότι όλα αυτά τα ποσά δεν δαπανήθηκαν και ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα σχέδιο κανονισμού που έχει σαν στόχο να επαναπροωθήσει τα μη καταναλωθέντα ποσά προς το Recovery Plan, προς ιδιωτικό ταμείο που θα έχει σαν στόχο όχι τα ιστορικά ιδιωτικά ταμεία, αλλά ένα άλλο ταμείο τέλο πάντων που θα βοηθήσει τη χρηματοδότηση διαφόρων προγραμμάτων σχετικών ενεργειακών προγραμμάτων συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία θα είναι αποκεντρωμένα. Είναι ένα πρόγραμμα που το θέλουμε πάρα πολύ η κυρία Κατρίν Βανπρέν την εισηγήτρια του Κοινοβουλίου και πάνω σε αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε ούτω ώστε να προχωρήσει το χαρτοφυλάκιο θα γίνει συζήτηση πολιτική στο άτυπο Συμβούλιο 6 και 7 Σεπτεμβρίου και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων θα συζητήσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο και τα οικονομικά θέματα. Είναι ένα πρόγραμμα, πιστεύω, που είναι πάρα πολύ καλό, διότι ίσω είναι το στοιχείο που λείπει από όλη την ενεργειακή νομοθεσία που έχουμε σήμερα. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε να έχουμε μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, εάν θέλουμε να το κάνουμε τόσο ώστε οι καταναλωτέ να το εκμεταλλευτούν, κυρίω οι πλέον ευάλωτοι καταναλωτέ, οι τοπικοί εμπορευόμενοι είναι εκείνοι οι οποίοι είναι πιο χρήσιμοι και πιο αποδοτικοί για να προχωρήσουμε. Παραδείγματο χάρη, Δήμοι καθώς και ε, κοινωνική πρόνοια για τη στέγαση. Όλοι οι φορεί για τη στέγαση είναι βασικοί φορεί που μπορούν να βοηθήσουν να επιταχύνουμε τι επενδύσει αυτέ και να φροντίσουν τόσο ώστε η ενεργειακή μα κατανάλωση και το μερίδιο τη ενέργεια που πηγαίνει στα νοικοκυριά να μειωθεί δραστικά τα επόμενα χρόνια. Θα έχουμε επίση τη χαρά στη συζήτηση επί των επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση να περιμένουμε τον Φιλίπ Μιστά, τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Τάπεζα Επενδύσεων, που μαζί με τον Μάριο Μόντιν, ονόμα για να παρουσιάσει την, ε, παρουσιάσουν τι εκθέσει τους. Θα είναι παρόντες στο Συμβούλιο το επίσημο. Κάποια λόγια να πω όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια, αιωλική, offshore. Ε, είναι, κάτι, είναι το πάθο τη Βελική Προεδρία, διότι έχουμε οικοδομούμε στη Βόρεια Θάλασσα τέτοιο, ε, τέτοιες αιωλικά μηχανήματα υπεράκτια και στη Λέγη υπεγράφει συμφωνία του περσμένο Αθηνόπορου για να δημιουργηθεί ένα κοινό δίκτυο, ένα υπερδίκτυο σε όλη τη Βόρεια Θάλασσα, ούτω ώστε να συνεργαστούν οι διάφορες εγκαταστάσεις και να μοιραστεί και το κόστος. Ε, ήδη μας υποστήριξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό και θέλουμε να υπογράψουμε στα περιθώρια του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ 10 κρατών μελών ούτως ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο κατασκευής των αιωλικών αυτών εγκαταστάσεων το μεγαλύτερο πρόγραμμα όσον αφορά την ανανεώσιμη πηγή, ανανεώσιμες ενέργειες. Και τέλος η Προεδρία θα θέλει να μπορέσουμε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου να συζητήσουμε και τα μακροπρόθεσμα οράματα. Έχουμε πρώτη ευκαιρία να το κάνουμε. Το σχέδιο δράσεως Ενέργεια 2011-2020, σχέδιο δράσης και για τις εσωτερικές πολιτικές και τις εξωτερικές μας πολιτικές. Και εκεί ε, θέλουμε να μπορέσουμε σε αυτά τα πλαίσια να φροντίσουμε να δώσουμε σάρκα και οστά σύντομα στην, ε, στην, στα προγράμματα αυτά για το πακέτο ενέργεια που εγκρίναμε το 2008 θέλουμε να δρομολογηθούν συγκεκριμένε πράξεις. Οι συζητήσεις ήταν ιδιαίτερα πλούσιες επί Ισπανική Προεδρία. Εμείς θέλουμε να συνεχιστούν. Και τώρα θα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίω και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάθε φορά που το επιθυμεί να συμμετάσχει, θα ξεκινήσει η συζήτηση όσον αφορά την πραγματική πολιτική, τη μακροπρόθεσμη, όσον αφορά τον οριζόντα του 2050. Όλοι πρέπει να γνωρίσουμε ότι 2050 είναι η ημερομηνία γύρω από την οποία θα πρέπει να διαμορφώσουμε την ενεργειακή πολιτική, τη μακροπρόθεσμη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει τι εργασίε ούτω ώστε να καθοριστεί ένα οδικό χάρτη για το 2050, Ένα προβληματισμό για το ενεργειακό μα μείγμα όσον αφορά την ε, ολοκλήρωση ενιαία αγορά τη σχέση με τι εξωτερικέ χώρε, όσον αφορά τι αναγκαίε επενδύσει, όσον αφορά τι υποδομέ, όσον αφορά τη ρύθμιση, όλα αυτά είναι απαραίτητα. Θα είναι μια συζήτηση εξαιρετικά σημαντική και ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση με τον ύψιστο βαθμό απαιτήσεων και φιλοδοξιών. Ε, κάποιοι επιστήμονες είναι πεπισμένοι το 2050 η Ευρώπη θα μπορούσε αν το αποφασίσει σήμερα να διαθέσει τα μέσα ε, να 100% ή 80-90% να απαλλαχθεί από τα ορυκτά καύσιμα ε, δεν θα τα καταφέρουμε το 2050, παραμένουν να κάνουμε σήμερα τι πολιτικέ στρατηγικέ επιλογέ θα επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ειδού και αυτή μια συζήτηση που θα θέλαμε να ξεκινήσει από τι προεδρίε μα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να μην κρυγόρισα όσον αφορά την παρουσίαση των βασικών αξώνων και τι προτεραιότητε που έχουμε θέσει. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ, για την παρουσία σας. Περίπου μισή ώρα στη θέση μας τώρα και δέκα συναδέλφους που ζητούν το λόγο. Παρακαλώ λοιπόν να είμαστε στο δυνατόν πιο σύντομοι. Η κυρία Χόλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Βελγική Προεδρία. Ιδιαιτέρως, με ικανοποίησαν αυτά τα οποία είπατε, όσον αφορά την παινία, όσον αφορά τα καύσιμα και όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αποδοτικότητα στη χρήση της ενέργειας γιατί προηγουμένως δεν αναφέρθηκε τίποτα σχετικό. Οπότε επιτέλους άκουσα κάτι τέτοιο και κατάλαβα ότι θέρατε την ενέργεια να τη συζητήσετε στο Συμβούλιο στις 6 και 7 Ενάτου. Συγκεκριμένα, τι θέλει να κάνει για το πρόγραμμα δράσης η Βελική Προεδρία. Είπατε ότι τώρα θα πρέπει να πείσετε τα κράτη-μέλη κάτι να κάνουμε και αυτό θα το κάνετε με το που θα τάξετε κάποιους στόχους σε ενωσιακό επίπεδο. Και έτσι να δώσετε μια στην ε, σχετική οδηγία τώρα. Όσον αφορά το πρόγραμμα αυτό Τι γίνεται με την χρηματοδότηση. Γιατί υπάρχει εδώ ένα μεγάλο χρηματοδοτικό κενό. Τι γίνεται με αυτό το σχέδιο ανάκτησης. Εσείς Από πού θεωρείτε θα προέλθουν οι πόροι αυτοί, ούτω ώστε να μπορούμε να έχουμε νέε πράσινε θέσει απασχόληση σε όλη την Ένωση. Λάμπατς. Λάμπερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλώ ήρθατε, κύριε Μανιέτ. Πολλά ενδιαφέροντα ακούσαμε κατά την ομιλία σα. Εγώ θα αναφερθώ στα εξή δύο. Μίλησατε πολύ για την προστασία του καταναλωτή. Η καλύτερη προστασία βέβαια του καταναλωτή είναι η αποφυγή των μονοπωλίων ή ιονή μονοπωλίων που καταχωρούνται τη αγορά. Και επίση γνωρίζετε πολύ καλά ότι ε, η ε, Προμηθευτέ ενέργεια και κυρίω αυτοί που έχουν κάνει τι επενδύσει του στην πυρηνική ενέργεια που έχουν τεράστιο περιθώριο κέρδους, έχουν τεράστια συγκέντρωση. Βλέπουμε όμως από αυτό που κάνετε στο Βέλγιο εσείς ότι επιβεβαιώνετε την καταδυνάστευση της αγοράς για ακόμη μεγαλύτερη χρονική περίοδο για τις συγκεκριμένε αυτές εταιρείε. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν, κάποιες από απόπειρε στο Βέλγιο δεν εστέφθησαν με επιτυχία και ενισχύω ιδιαίτερα για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Και επίσης, ισχυρίζεστε ότι θα περάσετε από, ε, σε, σε ένα ενεργειακό μείγμα ανεξάρτητο σχεδόν από, το, από τα καύσιμα τα ορυκτά, ε, πράγμα το οποίο χαιρετίζουμε, βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι και το ουράνιο, το οποίο είναι ορυκτό, δεν θα το, θα το συμπεριλάβετε και αυτό στην κατηγορία των ε, ορυκτών καυσίμων από τα οποία πρέπει να είναι απαλλαγμένη η ε, ενέργειά μας. Και θα ήθελα να ρωτήσω για το 2020 τι στόχους έχετε. Κύριε Φανμπρέμπτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχή για τα όσα άκουσα. Ερωτήσεις για το σχέδιο ανάκαμψης δεν έχω. Ξέρω κύριε Υπουργείο ότι το παρακολουθείτε με πολύ ενθουσιασμό. Τώρα βέβαια θα πρέπει να ανασκουμποθούμε για να πείσουμε το υπόλοιπο Συμβούλιο. Όμω ένα θέμα το οποίο ιδιαίτερα με ενδιαφέρει και με ανησυχεί είναι το εξή. Το, το Βέλγιο δείχνει ιδιαίτερη, υψηλή φιλοδοξία στα θέματα τα κλιματικά και θέλει να εγγυθεί τη Ευρώπης στην προσπάθεια για μια νέα ανάκαμψη κλιματική στην πρωτοπορία. Αλλά πρέπει αντίστοιχα να είμαστε και εμεί στη δική μας ε, εσωτερική πολιτική συνεπής και πρέπει να αναθεωρήσουμε το ενεργειακό μας μείγμα. Θα πρέπει για το μέλλον να επανεξετάσουμε την χρήση του άνθρακα και βέβαια των άνθρακορυχείων. Πρόσφατα, όπως ίσως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ανακοίνησε το θέμα λέγοντας ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η εκμετάλλευση του άνθρακα το 2023 και διαθέτοντας 23 δισεκατομμύρια ευρώ η συνέχιση της εκμετάλλευσης των ανθρακοργείων. Ένα-δύο λεπτά, Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και ως εκ τούτου είναι παράλογο το να υποστηρίζουμε με τέτοια κονδύλια τα ανθρακοργεία. Το θέμα αυτό θα έρθει και στο Συμβούλιο, από φαίνεται η Βελγική Προεδρία τι θα σκοπεύει να κρατήσει. Το ΔΕ Συμβούλιο στο σύνολό του. Δεν θα πρέπει πια να δώσουμε τέρμα σε τέτοιου είδου επιδοτήσει, να μην χρησιμοποιούνται τα κονδύλια αυτά παρά μόνο για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και την αναδιάρθρωση βέβαια του τομέα. Ευχαριστώ, κύριε Ζαντού. Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω ότι και εγώ ιδιαίτερα εκτιμώ τα όσα μας είπατε για το Ε, μέλλον της ενέργειας. Στην Ευρώπη όμως έχουμε μεγάλη μεγάλες περικοπές ως προς τα κίνητρα που δίνονταν για τις ανανεώσιμες πηγές. Και αντίστροφα βλέπουμε τις Ηνωμένες, πηγές, τις Πολιτείες και την Κίνα μαζικά να, επενδύσουν, να επενδύουν σε τέτοιου είδου ε, τεχνολογίες, οι οποίες και εσείς υποστηρίζετε και επιδιώκετε. Τώρα βλέπουμε να προτείνονται επενδύσεις για 4,5 ε, δισεκατομμύρια ε, σε σχέδια τα οποία δεν έχουν απτά αποτελέσματα και άλλα 3 δισεκατομμύρια για τον άνθρακα. Ερωτώ λοιπόν εάν είστε διατηθειμένος να δεσμευτείτε για πιο αποτελεσματικούς στόχους, πιο δεσμευτικούς στόχους. Μιλήσατε επίσης για ε, σήμανση στις ε, ε, τηλεοράσεις, στις θερμάστρες και τους λέβητες καύσης. Πράγματα όμως τα οποία δεν προχωρεί από ό,τι φαίνεται σε συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε την αποφασή να προχωρήσετε κατά τρόπο σαφέστερο για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κυρία Τσικάου, παρακαλώ. Και εγώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν σκοπεύετε να αξιοποιήσετε την ε, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών για να διαθέσετε επιδοτήσεις για την θερμική προστασία των ε, κτηρίων. Γιατί τέτοιο πράγμα δεν προβλέπεται. Καταρχάς λοιπόν προβλέπετε την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση για τις δημοσιονομικές ε, προοπτικές να την αξιοποιήσετε για την ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα των κτηρίων. Και επίσης, κάνατε λόγο για κάποιες πράξεις ανάθεσης. Σε σχέση με τη σήμανση των ηλεκτρικών συσκευών. Ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο διαφώνησε πέρυσι με τις θέσεις της Επιτροπής. Γι' αυτό θα παρακαλέσουμε να ακολουθήσετε τις θέσεις του Κοινοβουλίου στο μέλλον, στην υπόθεση αυτή. Κύριος Μπέλετ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλή επιτυχία στο έργο σας κύριε Υπουργέ. Ήδη Μα αναφέρεται για την περιβαλλοντική τραγωδία στον κόλπο του Μεξικού. Την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα πρέπει να συγκροτηθεί ένα εργαστήριο, ούτω ώστε να μπορούμε να δούμε τι γίνεται όσον αφορά με κάθε διαρροή πετρελαίου στα χωρικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα όμω θα γίνει ένα, το μορατόριο, θα έχουμε μια ομάδα υψηλού επίπεδου. Για πετε μα, όσον αφορά αυτό το μορατόριο για την εξόριξη πετρελαίου, ε, πόσο θα κρατήσει, πώ θα λειτουργήσει ακριβώ αυτή η ιδέα. Έχετε έρθει σε επαφή με τις ε, ε, εταιρείε που ασχολούνται με την εξόριξη. Καβαίου. Uh, Κύριε Γραβάλιο, ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για το πρόγραμμα το οποίο με κάθε λεπτομέρεια μας εξέθεσε και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι μια μακρόπνοη ενεργειακή πολιτική συνδέεται άρρηκτα με την καταπολέμηση της ε, αλλαγής του κλίματος και ένα από τα πιο σημαντικά είναι η διεθνής διαπραγματεύση για την αλλαγή του κλίματος. Είναι πάρα πολύ βασικό να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε όσον αφορά το περιβάλλον. Επίσης όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό όσον αφορά και την ανταγωνιστικότητά μας και ιδίω την ε, βιομηχανία έντασης ενέργειας. Γι' αυτό και σας ερωτώ, τι έχετε προγραμματίσει όσον αφορά αυτή την ε, βιομηχανία ένταση ενέργειας. αν δεν καταφέρουμε να έχουμε κάποιο είδους ε, σύμφωνια, πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια τέτοια βιομηχανία και τι θα γίνει, γιατί ε, ταυτόχρονα προετοιμάζονται για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και τι νέε τεχνολογίες η Ιαπωνία, η Κίνα και άλλοι ανταγωνιστέ. Τι λέτε. Ευχαριστώ. Λάγκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κεντρικό σημείο για την νέα παραγωγή ενέργεια στην Ευρώπη είναι τα δίκτυα. Τα συζητήσατε ακροφυγώς. Μιλήσατε βέβαια και για την παραγωγή μέσα στα τα offshore τα πάρκα offshore. Το σημαντικό μου στοιχείο σε όλες αυτές τις νέες προσπάθειες είναι τα δίκτυα. Ο εξυγχρονισμός των δικτύων, πώς μπορεί να προχωρήσει, ποια είναι τα πρώτα βήματα και βέβαια πού θα βρούμε τα κεφάλαια. Ο Γκούρκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ θερμά για την ε, παρουσία σα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα παρά το, την πίεση του χρόνου και πλήρες. Από ό,τι βλέπω, η Βελική Προεδρία σκοπεύει να συνεργαστεί με, με την προηγούμενη, την Ισπανική, αλλά και με την επερχόμενη, την Ουγγρική Προεδρία. Αυτό είναι πολύ βασικό Ξέρουμε ότι τα προβλήματα ε, στον εφοδιασμό σε ενέργεια δεν γνωρίζουν προεδρίες και ίσως ακόμη η προσεχής προεδρία, η Ουγγρική δηλαδή, να αντιμετωπίσει νέα προβλήματα εφοδιασμού σε αέριο, σε φυσικό αέριο. Με την Αυτογκάση λοιπόν και την Κασπρόμ, τι είδους συμφωνίες νομίζετε ότι μπορούν να αναπτυχθούν, έχουν χαρακτηριστεί αυτές ε, ιστορικής σημασίας, έχουν χαρακτηριστεί συμφωνίες που θα εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό σε ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η Βελγική Προεδρία πιστεύει ότι μπορεί να συνδιαμορφώσει αυτές τις συμφωνίες, δηλαδή να είναι παρούσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επεξεργασία τους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, μίληξατε για διάφορα θέματα. Εγώ είχα υπόψη τον κύριο Μον τις απαντήσεις του ως προς τις παρατηρήσεις ε, του κυρίου Μπαρός ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ενιαία αγορά και τον ανταγωνισμό. Εσείς είπατε ότι χρειαζόμαστε αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην ε, χίδιν παραγωγή και διανομή ενέργειας. Φαντασμό ότι εννοείται την ηλεκτρική και το φυσικό αέριο. Πώς σκοπεύετε αυτό να το επιτύχετε, ο ρόλος της Προεδρίας σας ποιος θα είναι θα ε, δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στην ε, ενέργεια, στα δίκτυα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολύ ωραία φαίνονται όλα αυτά. Ανταγωνισμός στην ε, ε χίδιν εμπορία ενέργειας, αλλά πώς θα το καταφέρετε αυτό. Κύριος Ουντζή. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και... Ουντζή και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ για, την, για το δυναμισμό που επιδεικνύεται ύστερα από την Ολομέλεια που μόλις ολοκληρώθηκε νομίζω ότι ξεκινάμε τους καλύτερους σιωνούς, η Βελγική Προεδρία. Έχουμε όμως ένα πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Καριλαίο και με άλλα ε, υλοποίησης σχεδίων. Εσείς από το Συμβούλιο, από την Προεδρία, Ποια είναι η που έχετε αποκομίσει για το Desert Tech, γενικά για την ενέργεια και την οικονομία. Βλέπετε να υπάρχει η δυνατότητα και οι ικανότητες να ξεπεράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους διχασμούς της και να προχωρήσει στην υλοποίηση μεγάλων σχεδίων. Και δεύτερη ερώτηση ως προς τη ρύθμιση των αγορών ενέργειας. Έχουμε 27 εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Έχουμε και την Ευρωπαϊκή. Αλλά πώς μπορεί Χρειαζόμαστε μάλλον μια ευρωπαϊκή, εάν δεν υπάρχει ε, ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή με πραγματικές όμως εξουσίες, πόσο θα εξασφαλίσουμε τη ρύθμιση των αγορών. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Μανιέτ, ασφαλώς πολλές και ποικίλε ερωτήσεις. Έχετε το χρόνο να απαντήσετε και αν δεν προλάβετε σήμερα τους προσεχείς, τις εβδομάδες και μήνες ασφαλώς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ας προσπαθήσουμε όμως να δώσουμε μια πρώτη σειρά απαντήσεων. Κύριε Μανιέτ. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι βουλευτές για τις τόσες ερωτήσεις σας. Τόσο ενδελεχείς, ούτως ώστε και εγώ θα μπορέσω να σας απαντήσω όμως για μεγαλύτερη ακρίβεια. Ναι, θα πρέπει πάντοτε να μπορεί κανείς να συγκεράσει το, το όραμα με το συγκεκριμένο ε, πρόγραμμα, ε, αυτό θα πει πολιτική και οπότε δεν θα πρέπει όμω ε, να μην παραπονούμε ούτε το ένα ούτε το άλλο και με αυτό ήταν το πνεύμα το οποίο διαπνέει την Προεδρία όσον αφορά την προεδρία. Ξέρουμε ποιο είναι το όρομα, το έχουμε, το έχουμε δει, έχουμε, το έχουμε επεξεργαστεί και θέλω να δούμε τι μπορεί να γίνει μέσω αυτού του εγγράφου που είναι τόσο βασικό το 2005 για να ξεκινήσει η προβληματική και αυτό έγινε μέσω διαβουλεύσεων προσκλήσεων ε, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όσο γίνεται πιο πολλές φιλοδοξίε και βέβαια εμεί πάρα πολύ συγκεκριμένα θα ε, ασχοληθούμε με τα συγκεκριμένα ε, προγράμματα για να δούμε πώς όλα αυτά εντάσσονται στο σύνολο και να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Είναι αυτό το οποίο σας είπα στην συνοπτική εισαγωγή για τις υποδομές και όχι μόνο για τα δίκτυα που βέβαια ε, θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με το σχέδιο ανάκτησης που και αυτό κατά κάποιο τρόπο θα γίνει ένα έμβριο ε, της δομής της πολιτικής που θα φτιάξουμε και λέμε για 114 εκατομμύρια πάνω κάτω, αλλά πρόκειται τέλο πάντων για ένα λογικό προπολογισμό. Το σημαντικό είναι να μπει το πόδι στην πόρτα, να υπάρχει ένα μέσο το οποίο στη συνέχεια να είναι δυνατόν στα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών να μπορούμε κάτι να κάνουμε. επίση και όσον αφορά το πρόγραμμα δράση για την ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι η κορονίδα τη πολιτική μα και πριν αρχίσουμε να, τη συζήτηση για το τι θα γίνει όσον αφορά την ε, αποτελεσματική της ενέργειας, θα πρέπει η Κομισιόν να μας πει τι θα κάνει. Τι, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι, ε, τι, τι είναι όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε. Να, τι θέλουμε να μας απασχολήσουν και κατόπιν 6 ε, και 7 Σεπτεμβρίου θα συζητήσουμε το Συμβούλιο να δούμε τι κανόνες χρειάζονται, αν χρειαζόμαστε περισσότερα αυτά τα οποία συζητούμε, αναφέραμε όσον αφορά τις ε, κατανάδες κατουξιοδότηση πράξης και υπάρχουν και άλλα θέματα όσον αφορά τα προϊόντα που χρησιμοποιούν και δεν καταναλώνουν ενέργεια, έρευνα, ανάπτυξη, προβληματική. Ήδη έχει αρχίσει ε, στο πλαίσιο του προγράμματος. Ε, έχουμε κάποια δισεκατομμύρια και για όλα αυτά έχουμε πει ότι είναι δυνατόν και για την ε, ανακύκλωση, να ξέρουν τι μπορεί να γίνει και είπαμε ότι οι ανανεώσιμε μορφές ενέργειας είναι πάρα πολύ βασικές και στην επιλογή μας για το πού θα επενδύσουμε θα πρέπει να τα κάποιες προτεραιότητες και τα είπαμε αυτά στα πλαίσια των προοπτικών για να μπορέσουμε να προωθήσουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε συγκεκριμένους στόχους και όσο μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς μπορούμε να μειώσουμε ή να νομίζουμε ότι ξέρουμε τέλος πάντων να μειώσουμε τις ε, επιβλαβείς ε, εκπομπές για το θέμα του θερμοκηπίου, τότε θα ξέρουμε καλύτερα να, το, αξιολογήσουμε το πώς μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους, να έχουμε μετρήσιμους στόχους. Και αυτό είναι τελικά το ζουμί και βέβαια είναι και το θέμα της ε, οικονομικής υποστήριξης όταν είναι της αξιολόγησης αυτού του προγράμματος και παραπέρα θα πάμε σε ένα δεύτερο πρόγραμμα δράσης που θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ένωση πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία του Συμβουλίου να γίνει ένα συμβούλιο έκτακτο για τα ενεργειακά στις 4 Φεβρουαρίου για να δούμε πώς θα συνεχιστούν αυτά τα οποία θα χαράξει η Βελγική Προεδρία, πώς θα απεμπλέξουμε κάποια θέματα που έχουν κολλήσει και πώς θα υπάρξει κάποιο του συνεννόηση. Ανταγωνισμός, μονοπόλια, πώς θα, θα έχουμε περισσότερη ποικιλία και πολυφωνία στην ενεργειακή αγορά και στα δίκτυα. Όλα θα βγαίνουν από το πρόγραμμα της, ε, της Προεδρίας και αφορούν και ταυτόχρονα και ερωτήσεις σας. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη δράση για όλα αυτά, δεν υπάρχει συγκεκριμένο θέμα, συγκεκριμένο φάκελος που να έχει ανοίξει. Ε, και θα πρέπει έτσι καλλιώ το α ή το β θέμα ε, θα πρέπει να, να, δούμε ότι για να είναι κάποιος αποτελεσματικός δεν μπορεί να έχει 17 προτεραιότητες, έχει 3-4. Όμως εμείς κατά το άτυπο ε, συμβούλιο τα θέματα των ευάλωτων ε, καταναλωτών ή μορφών ενέργειας θα τα συζητήσουμε από πλευράς όχι των μεγάλων εταιριών, από πλευράς των καταναλωτών. Κάποια στιγμή θα υπάρξει και το επόμενο τέταρτο πακέτο ενεργειακό, γιατί έχουμε την, ε, είχαμε την τρίτη οδηγία που ανέδειξαν σωρό θέματα και κάποια μέρα θα, θα έχουμε κάτι παραπάνω από έναν απλό συντονισμό των ε, εθνικών ρυθμιστικών αρχών, ας πούμε για τα τιμολογιακά. Και εδώ στο Βέλγιο θα ξέρουμε ότι όταν υπάρχουν δύο μεγάλοι φορείς που δρούν στη χώρα, τότε οι ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν αρκετή ισχύ ώστε να εξασφαλίσουν μια διαφανή, πλήρως διαφανή λειτουργία της αγοράς. Να, ποια είναι η ουσία του προτινασμού για την ενεργειακή πολιτική. Ε, μιλούμε για δίκτυα, τα είπαμε και στα πλαίσια των υποδομών, στα πλαίσια του σχεδίου ανάκτησης, στα πλαίσια αυτών των πρωτοβουλειών που είναι περιφερειακές, διακυβερνητικές και ταυτόχρονα, ταυτόχρονα αφορούν ε, και τις βιομηχανίες όπως ε, η υπόθεση της Βόρειας Θάλασσας αλλά θέλουμε να υπάρξει διασύνδεση μεταξύ των εθνικών ε, υποδομών. Αλλά αυτό να αφορά και συνόηση με τους γείτονες και να μπορούμε έτσι να έχουμε μια διαφοροποίηση Είχαμε κάποιε ερωτήσει που δεν μπορώ να τι απαντήσω γιατί είναι εθνικέ πολιτικέ ε, για άνθρακα, επενδυτική ενέργεια. Κύριε Μπέλε, τόσο αφορά τι εξορίξει, αρχίσαμε όλα αυτά να τα διερευνούμε. Νομίζω ότι υπάρχει πρόοδος. Έχουμε την Επιτροπή Διαβούλευσης με τη Βιομηχανία. 18 Ιουνίου υπάρχει Συμβούλιο. 8 Μαΐου, 8 Μαΐου έγινε. 31 Μαΐου επίσης ε, έγινε συνεννόηση και τα είπαμε και στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα, οπότε αρχίσαμε να εκπονούμε ε, μια, μια τέτοια προβληματική τη συζήτηση για το τι γίνεται στη Βόρειο Θάλασσα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάποιοι ήδη υπάρχουν όσον αφορά την ασφάλεια στις πλατφόρμες τους εργαζομένους για την άλλη μεριά, πώς θα είναι οι μηχανισμοί αντίδραση σε περίπτωση ατυχήματος και είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να, να, παγώσει η μετάφραση της Βόρειας Θαλάσσης ε, μέχρι ότου ολοκληρωθούν αυτές οι κινήσεις, και αναλύσεις. Ακόμα δεν έχει αποφασίσει το Συμβούλιο, αλλά συμφωνούμε να συνεχιστεί ο προβληματισμός και να αποφανθούμε στο μέλλον. Τώρα, όσον αφορά το κλίμα, όσον αφορά τους κλιματικούς στόχους, Βέβαια αυτό δεν αφορά τόσο στενά το Συμβούλιο Ενέργειας, αλλά είναι βέβαια κάτι πάρα πολύ σχετικό και πρέπει να ακολουθήσει το Συμβούλιο τι γίνεται, από το 20 το 30% να προχωρήσουμε, λέγει μια ερώτηση και άλλη είναι τι θα κάνουν. Επί Ισπανικής Προεδρίας, τα είπαμε στην Σεβίλη, έγινε πάρα πολύ αξιόλογη συζήτηση και είπαμε στην Επιτροπή ότι το λάθος της Κοπενχάγης είναι λιγότερο σχέση με το πώς, πώς κατεβήκαμε και από την άλλη ε, περισσότερο ήταν το ότι είπαμε ότι τι θα γίνει το 30% που εμείς θα κατέβουμε αν δεν κατέβουν οι άλλοι. Ίσως πρέπει να πούμε ότι αν περάσουμε μονόπλευρο, τόσο ώστε να δημιουργήσουμε μια τάση, μια όθηση. Να, τι έγινε. Οι άλλοι δεν προχώρησαν, είδατε τι έγινε σε Κίνα, Ινδία, είπα. δεν υπήρχε σύνεση για να πάμε το 23%. Και έτσι θα έκλεινε συζήτηση. Και έτσι κάτι θα γινόταν από μέρους μας στην Κανκούν και στο μέλλον, παραπέρα. Επί τη βάση των φάσεων της Κοπενχάγης. Αλλά κατόπιν δεν θα θέσουμε ότι έκλεισε το θέμα παρά μόνο να τολμήσουμε να έχουμε απόφαση για το αν θέλουμε να έχουμε έναν μηχανισμό ή θα προχωρήσουμε, ε, ε, αποφασίσουμε θα ρισκάρουν οι βιομηχανίες μας. Αυτό είναι το βασικό για τη συζήτηση. Και το δεύτερο είναι το αν γίνει μονόπλευρη αλλαγή από 23% θα είναι αυτό κακό για τους Ευρωπαίους. Τα είπαμε τον Ιανουάριο. και λέγαμε τότε ότι το 23% είναι καλό για την Ευρώπη μεν και θα, θα εντυπωσιάσουμε. Καλό είναι, αλλά δεν εντυπωσιάζουμε κανέναν. Πρόοδο τεχνολογική υπάρχει, από την άλλη μεριά έχουμε επιβράδυνση τη βιομηχανική παραγωγή και θα θέλει επιπλέον προσπάθεια από το 23%. Και άρα έτσι θα υπάρξει ένα πλεονέκτημα. Πλεονέκτημα να κάνουμε πρώτη τη ρύθμιση, αλλά παράλληλα να μην πλήξουμε τι βιομηχανίε μα έναντι του υπολείπου κόσμου. Να δούμε πώς θα ε, πώς αρμόσουμε αυτά τα μέτρα στη βιομηχανία μας και τι θα κάνουμε γιατί κατά 80% αυτό είναι θέμα ενεργικής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για τα όσα μας είπατε, για τις απαντήσεις σας δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε περισσότερο τα θέματα αυτά. Έχουμε ολοκληρώσει το θέμα τη ημερήσια διάταξης, αλλά προφανώς στι προσεχείς εβδομάδε και μήνες θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διάφορα θέματα. Ευχαριστώ θερμά λοιπόν για την παρουσία σα εδώ και τις πληροφορίες σας. Merci beaucoup. darf Sie alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, aufrufen, direkt Αγαπητοί συναδελφέ, περάσουμε απευθεία ε, στο προσεχή θέμα τη μαριστική διάταξη με την κυρία Φαν Μπρέντ. Δεν έχουμε χρόνο, προχωρούμε. Ακόμα και χωρί την κυρία Φαν Μπρέντ, γιατί δεν τη βλέπω εδώ. Κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Το πρόγραμμα δύσκολο. Κυρία Φαμπρέμπτ, σημείο 6 σχέδιο ανάκαμψης του έχουμε ήδη συστήσει μια φορά. Υπάρχει τίποτα καινούριο. Όσο το δυνατόν. Σύντομα παρακαλώ. Έτσι το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, μπορώ να είμαι σύντομη. Χάρηκα που ο υπουργό ο κ. Μανιέτ επιβεβαίωσε εκ νέου ότι θεωρεί ότι η πρόταση αυτή είναι σημαντική διότι καινοτομεί και καινοτομή όσον αφορά την χρήση των πόρων, όσον αφορά τις επενδύσεις για ενεργειακή απόδοση και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι έχω να πω. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικότατη πρόταση, διότι για πρώτη φορά διάφοροι παράγοντες συνδυάζονται. Τα ημί χρησιμοποιηθέντες πόροι που κανονικά θα επεστρέφονται 114 εκατομμύρια ευρώ μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο μέσο χρηματοδοτικό που θα χρησιμοποιείται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στα κράτη-μέλη και μπορεί να γεννά επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι καλό για την απασχόληση, είναι καλό για τους στόχους μας σχετικά με το κλίμα και πάνω απ' όλα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο να μην υπάρχουν μετεγκαταστάσεις. Τρίτον, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η προσέγγιση δημιουργώντας και άλλους πόρους. Ο στόχος της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποιος είναι. Ότι μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρήματα ευρωπαϊκά μπορούν να μπουν σε ένα ταμείο για να δημιουργηθούν επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε αυτή την προσέγγιση σαν κοινοβούλιο. Και αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε είναι η διαφάνεια. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τα οικονομικά και το πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει και εμπιστοσύνη όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καινοτομήσει. Όπως είπε και ο Υπουργό, είναι ένα μικρό βήμα, αλλά ένα πρώτο βήμα το οποίο μακροπρόθεσμα ίσως να απελευθερώσει πολλούς πόρους από διάφορους αθυσιμοποιητούς πόρους. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά το πρόβλημα είναι ότι σε τοπικό επίπεδο υπάρχει έλλειψη ε, κεφαλαίων. Και αυτό είναι ένα μικρό βήμα για να διορθωθεί αυτό. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι στην έκθεσή μου ε, έχουν, για την έκθεσή μου έχουν αποβληθεί κάποιες τροπολογίες. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κοντά στις επιθυμίες του Κοινοβουλίου, αλλά και εγώ ήθελα να στείλω και κάποιο μήνυμα μέσω των τροπολογιών που συμπεριλαμβάνω. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό αυτή η πρόταση να υιοθετηθεί τάχιστα. Θα ψηφίσουμε εμείς εδώ το Σεπτέμβριο και μετά μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και να προσπαθήσουμε να περάσει το κείμενο στην πρώτη ανάγνωση. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να υποβάλλετε τροπολογίες και ότι δεν μπορεί να βελτιωθεί το κείμενο. Το θέμα είναι να υποστηριχθεί το κείμενο, να πετύχουμε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση και να έχουμε αυτό το ειδικό οικονομικό εργαλείο και να συμφωνήσουν και οι πολιτικές ομάδες και να υιοθετηθεί τον Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, κύριος Πρεσίνα, από τις πολιτικές ομάδες αρχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστώ την εισηγήτρια. Είναι, νομίζω, πολύ καλή η ευκαιρία και η πρότασή της. Φυσικά μπορούμε να αξιοποιήσουμε κονδύλια για την ε, αναζωογόνηση της οικονομίας. Κονδύλια που διαφορετικά θα χάνονταν και νομίζω ότι με το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να συνδυάσουμε τα, την ε, ανάκαμψη της οικονομίας με τους στόχους, τους περιβαλλοντικούς και τους ε, ενεργειακούς. Ερωτώ όμως το εξής. 114 εκατομμύρια ευρώ. Από ό,τι φαίνεται είναι το ελάχιστο ποσό το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να έχουμε κάποια ικανοποιητικά αποτελέσματα, έτσι δεν είναι. Και δεύτερον, δημοσιονομικό μέσο. Για πόσο χρονικό διάστημα θα χρησιμοποιείται αυτό και πότε θα το έχουμε στη θέση μας. Το ταχύτερο δυνατό δηλαδή πότε θα τεθεί σε ισχύ. Ευχαριστώ η κυρία Χόλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, θα είμαι συντομότατη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια πάρα πολύ για τη δουλειά που έκανα. Συμφωνώ με τις τροπολογίες που προτείνει. Ε, έχω κάποια ανησυχία. Φοβάμαι ότι κάποια στοιχεία στο Συμβούλιο φαίνεται ότι είναι συγκεχημένα όσον αφορά κάποια στοιχεία του προγράμματος. Παραδείγματο χάρη. Λένε δεν μπορούμε να έχουμε ανοιχτό σχόλιο για μελλοντικέ αναλήψει υποχρεώσεων, ενώ αυτό απελευθερώνει άλλου πόρου που ίσω είναι διαθέσιμοι. Δεν ήταν έτοιμα να υπολογιστούν, ξέναν θα είναι διαθέσιμα αυτά τα χρήματα Τα κράτη-μέλη θέλουν πάντα επιστροφή των χρημάτων. Επικρατεί αυτή η νοοτροπία και το κλίμα. Πριν από τις διαπραγματεύσεις, θέλω να ρωτήσω σε θέση να δώσετε κάποιο υλικό ή να αρχίσετε κάποιες ανεπίσημες συζητήσεις με τα κράτη-μέλη ακόμα και τώρα ούτως ώστε να μην επικρατήσουν αυτές οι απόψεις που ακούγονται τώρα περί επιστροφής των χρημάτων στα κράτη-μέλη, να μην επικρατήσουν έστω και σε ανεπίσημη φάση. Ευχαριστώ, Κάντσιον. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Κάντσιον. Ω κοιόδης εισηγητής του ΕΛΚ, αισθάνομαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και συμμερίζομαι αυτή την πρόταση ενός καινοτόμου ταμείου, σημαντικού ταμείου, θα μπορούσε να είναι το πέρασμα προς μια αρχή που παγιώνει, μάλλον δημιουργεί ε, δυνατότητες επενδύσεων και επιτρέπει και την προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων στη λογική συνεργασίας partnership επιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Άκουσα πριν τον Υπουργό που έλεγε ότι όσον αφορά το μόνιμο Ταμείο Συμφωνία Πόλητα, εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία, αν και αν είναι ε, περιορισμένο το ταμείο στα 114 εκατομμύρια. Στο τέλος αυτά τα υπόλοιπα τα 114 εκατομμύρια θα είναι πολύ περισσότερα διότι περίπου 4 δισεκατομμύρια είχαν δοθεί στο πρώτο τμήμα του προγράμματος ανάκαμψης και πιστεύω ότι θα επιστραφούν και άλλα χρήματα. Και αντί να γυρίσουν στα κράτη, καλό θα ήταν να πάνε και να γεμίσουν αυτό το ταμείο. Αυτό είναι καινοτόμο το ταμείο διότι θα προσελκύσει και ιδιωτικούς πόρους εκτός από διεθνείς οικονομικούς φορείς και αν θέλουμε να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ε, να είναι κερδοφόρο. Εδώ μιλάμε για δάνεια, μιλάμε για υποβολή εγγυήσεων, μιλάμε για συμμετοχή σε διάφορα αξιόγραφα και ομόλογα για σημαντικά προγράμματα. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το startup, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το αρχικό οικονομικό τμήμα, το χρηματοδοτικό, Αφού φτάσουμε στον ισοσκελισμό, στο break even, θα πρέπει λοιπόν μετά να έχουμε μια ανάκτηση των πόρων. Δεν θα πρέπει να συμμετέχει μόνο το Ταμείο στις διάφορες πρωτοβουλίες. Υπάρχουν διαθετικά ταμεία, υπάρχουν διάφοροι ιδιωτικοί φορείς όπως το ΕΣΚΟ. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες που μαζί όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν πηγή για τα μεγάλα προγράμματα που σήμερα ε, συμμετέχουν κυρίως η τοπική αυτοδίκηση και οι δημόσιοι πόροι. Θα πρέπει λοιπόν να προωθηθούν καινοτόμα προγράμματα και όχι μόνο από τον ε, δημόσιο τομέα αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι ένα εργαλείο πιλωτικό, κάτι που ξεκινά, αλλά θα πρέπει να φτάσουμε τελικά σε διαθρωμένο εργαλείο, διαθρωμένο μέσο για το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η θα μπορούσε μαζί με μας μέσω του πολλαπλασιαστικού φαινομένου που ανέφερε η συγγήτρια να συμμετάσχει και μετά από αυτό πιστεύω ότι σίγουρα θα εφαρμοστεί το μέσο. Σε πόσο χρόνο. Σωστό το ερώτημα που ετέθη από τον συνάδελφο. Αντιμετωπίζουμε ανάγκες τώρα και χρειαζόμαστε να δαπανίσουμε αμέσως. Είναι και το ερώτημα που έβαλα πριν, πριν στους υπουργούς. Πιστεύω ότι αν ξεκινήσουμε αμέσως τη δημιουργία ενός απλού ταμείου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα, θα πρέπει να κινηθεί αρκετά γρήγορα. Και μετά θα μπορέσουμε να το αναπτύξουμε αυτό το εργαλείο και θα μπορέσουμε να το αναπτύξουμε και να έχει περισσότερε δυνατότητε και να έχουμε και εμεί περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μα. Να λάβουμε υπόψη ότι όσον αφορά τη τεχνική πτυχή υπάρχει το πρόγραμμα Έλενα και μέσω αυτού μπορούμε και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι απαιτείται για τις υπηρεσίες. Να περιοριστούν όμως αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να, έχουμε, να καλύψουν προγράμματα με μέγιστο 10%. Να λάβουμε υπόψη επίση ότι όταν μιλάμε για προγράμματα που χρησιμοποιούν νέε τεχνολογίε, θα πρέπει να προσέξουμε να μην παρατείνουμε τα χρονικά διαστήματα. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις καλύτερες δυνατές τεχνολογίες που παρέχουν τα συστήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ούτω ώστε να μην ε, χρειαστούμε περισσότερο χρόνο ε, από αυτόν που είναι απόλυτα αναγκαίο. Πιστεύω ότι θα γίνει έξοχη δουλειά. Ακούσαμε και τους ε, υπουργούς και νομίζω ότι η συνοδεία των υπουργών μπορεί να ξεκινήσει κάτι σημαντικό παρόλο που οι πόροι, τα χρήματα είναι πολύ περιορισμένα για την ώρα. Ευχαριστώ. Ζαντού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστώ την εισηγήτρια για την δουλειά τη. Δεν έχουμε ιδιαίτερα να προσθέσουμε με σε σχέση με τα όσα έχει προτείνει, διότι θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Ξέρουμε ότι οι παραδοσιακέ δομέ δεν προτιμούν αυτού του τύπου την ε, χρηματοδότηση. Πρέπει να ενισχύσουμε ιδιαίτερα τις ανανεώσιμες και καινούργιες μορφές ενέργειας. Πρέπει λοιπόν όσο μπορούμε πιο γρήγορα να προχωρήσουμε έτσι ώστε οι πόλεις και οι περιφέρειες να έχουν το ταχύτερο δυνατό πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και είμαι βέβαιος, ελπίζω τουλάχιστον, ότι ε, όπως εργαστεί γρήγορα και το Κοινοβούλιο, το ίδιο και το Συμβούλιο θα λάβει τις αποφάσεις του το ταχύτερο δυνατό ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα χρηματοδότησης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσόνσκι. Ευχαριστώ και εγώ Πρόεδρε θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις ε, προσπάθειές της. Ε, εδώ γίνεται μια προσπάθεια να ενισχύσουμε τον ε, τομέα της ενέργειας, ένα θέμα μεγάλης σημασίας φυσικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεδομένων των προβλημάτων που είδαμε στο παρελθόν, ένα τομέα πολύ ευαίσθητος. Ως και ο λοιπόν θα ήθελα να συμφωνήσω πως όντως τα χρήματα αυτά πρέπει να διατεθούν και να παραμείνουν στον σχεδιασμό για την ενέργεια. Και επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι προγράμματα που έχουν μεγάλη σημασία και μακροπρόθεσμα έχουν χαρακτήρα οριζόντιο, ε, δεν θα πρέπει να τα αναμειγνύουμε με κάποια άλλα. Καλό είναι αυτά τα προγράμματα να έχουν ένα καλό προγραμματισμό και ανεξάρτητο προγραμματισμό. Δεν εξαντλούνται τα δημοσιονομικά μέσα τα οποία έχουμε διαθέσιμα, γιατί δεν υπήρχε επαρκής προετοιμασία. Γρήγορα να προχωρήσουμε και σε υλοποίηση των σχεδίων και σε ταχεία αντιμετώπιση των κρίσεων που είναι γνωστές σε όλους. Είναι πολύ σημαντικές οι προτάσεις της εισηγητρίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κυρία Φον Μπρέμ, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Η Επιτροπή. Πρώτα η Επιτροπή τότε, μάλιστα. Κύριο κύριος Καμπό. Yeah, please. If not necessary... Εάν δεν θέλετε, αν δεν είναι ανάγκη να μιλήσετε, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Κύριε Σκαμπό, όχι πρόεδρε, δύο λόγια μόνο. Θέλω μόνο να ευχαριστήσω τους βουλευτές που έλαβαν τον λόγο για την υποστήριξη προσφέρων στις προτάσεις της Επιτροπής και να ε, καταστώ ότι η Επιτροπή λαμβάνει την πρωτοβουλία χάρη σε μια πρωτοβουλία κοινοβουλίου, σε μια συμφωνία μάλλον κοινοβουλίου και συμβουλίου, όπου είχε κριθεί ότι δεν υπήρχε επαρκή χρηματοδότηση για τις ανανεώσιμες ε, πηγές και άρα, δυναμικά δηλαδή, συμφωνίες, υποθέτει ότι ε, το σχέδιο ανάκαμψης ε, γίνεται δεκτό μόνο εφόσον τα κονδύλια που μένουν αδιάθετα επανέρχονται και αξιοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές, στις νέες πηγές ενέργειας, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως είπε και η κυρία Φον Μπρέντ, για την πράσινη ανάπτυξη αυτές οι επενδύσεις είναι πολύ σημαντικό να υποστηριχθούν Είναι δύσκολο με τις συνθήκες οικονομικής κρίσης να χρηματοδοτηθούν οι πράσινες επενδύσεις εκείνες οι οποίες δεν έχουν απαραίτητα μέσω την ε, απόσβεση και το κέρδος. Ε, ακριβώς αυτό το ρόλο έχει να διδραματίσει αυτή η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή διάθεση άμεση κονδυλίων, το bankable όπως λέμε στα αγγλικά, και τη χρηματοδότηση κυρίως του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή με ένα ευρώ που θα δίνουμε από το δημόσιο κορβανά, θα έχουμε την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των χρημάτων μας και εμπλοκή βέβαια του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις. Ακούστηκαν κάποιες ερωτήσεις για το κρίσιμο όριο, το 114 εκατομμύρια. Μα ακριβώς και λόγω αυτού του, αυτού, του αποτελέσματος μόχλευσης μπορούμε ούτως ή άλλως με τα 114 ευρώ, ε, εκατομμύρια ευρώ μπορούμε να έχουμε ουσιαστική αλλαγή στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, αλλά πάντως και με περισσότερα ακόμα καλύτερα. Την ευκαιρία δεν πρέπει να χάσουμε. Εάν θα πρέπει να είναι το ταμείο μόνιμο ή όχι. Η πρόθεση δεν είναι να καταστεί μόνιμο το ταμείο, αλλά, αλλά ένα τέτοιο ταμείο εγγύσεων, εφόσον διαθέτει τις εγγύησεις του, ε, έχει ακόμη περιθώρια οικονομικά Άρα χρειάζεται αρκετός χρόνος ή χρόνια για να εξαντληθούν αυτά τα κονδύλια. Και από την άλλη θα πρέπει και η αγορά να κινηθεί εξίσου γρήγορα για να ζητήσει τα κονδύλια. Εμείς πάντως συγκεκριμένο όριο εξάντλησης του, ε, της ζωής αυτού του ταμείου δεν μπορούμε να ορίσουμε. Μια προοδευτική ίσως ε, μείωση που θα εκταθεί σε αρκετά χρόνια. Αυτά και από την κυρία Φανμπρέντ αλλά και τον κύριο Κανσιόν άκουσα την ιδέα της καινοτομία και νομίζω μπορούμε αυτή την πτυχή από την πρότασή μας να την ενισχύσουμε. Επίσης ακούστηκε μια ερώτηση για την τεχνική στήριξη, ένα σημαντικό στοιχείο 10%, 15%, 20%, δεν ξέρω ακριβώς ποιο ποσοστό θα καλύψει ε, χωρίς να είναι ουσιοδέστερη πτυχή της, ε, του Ταμείου ή τεχνική βοήθεια, εφόσον τη χρειάζεται η αγορά, θα διατεθεί. Η διάρκεια. Το πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο λαμβάνουμε την πρωτοβουλία. Έχουμε απόλυτη προθεσμία το τέλος του 2010 γιατί στο τέλος του 2010 δεν θα μπορούμε να ανακτήσουμε τα κονδύλια αυτά δυνάμει των δημοσιονομικών κανόνων. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει μέχρι τα τέλη του έτους να εγκριθεί αυτή η πρόταση και ευχαριστώ ιδιαίτερο σαν προκειμένου τις πολιτικές ομάδες, την κυρία Συγήτρια και τις πολιτικές ομάδες και την Επιτροπή σας για τις προσπάθειες τις οποίες ξέρω ότι έχει αποδειθεί και βέβαια και υπογραμμίστηκε ήδη και από πλευρά τη Βελγική Προεδρία ότι καταβάλλεται τέτοιε προσπάθειε έτσι ώστε το στόχο χρονικά να μπορέσουμε να τον τηρήσουμε. Ευχαριστώ κυρία Βαν για άλλη μια φορά. Είμαι πολύ σύντομη κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ θετικά και ενθαρρυντικά αυτό το οποίο ακούμε. Δηλαδή ότι οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν με αυτή την πρόταση. Αυτό είναι προϋπόθεση επιτυχίας. Έχω να πω στην κυρία Χολ όσον αφορά τις επαφές με το Συμβούλιο, τις άτυπες επαφές και εξελίξεις, Εγώ έχω καλές σχέσεις με την Προεδρία και ακούσατε τι μας είπαν οι εκπρόσωποι της Προεδρίας. Δεν ξέρω για τα άλλα κρατημέλη, αλλά έχω τους συναδέλφους που έχουν έτσι επαφή με τους ομολόγους των δικών τους χωρών, Γερμανία, Ισπανία και προσπάθησαν να τους πείσουν να τα βρουν οι υπουργοί στο Συμβούλιο. Γιατί στα όλα αυτά. Δεν πρόκειται για κάποιο τρομερό ποσό. Μίλαμε για 140 μέλη. 140 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ε, θα πονέσει κανένα κράτος μέλος. Φραγκοδίφραγγι είναι τα περισσοτερα τη κράτη-μέλη αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω αυτά τα χρήματα θα πάνε σε ένα ταμείο. Έτσι θα υπάρχει κάποιο είδου ε, μόχλευση για να μπορέσουμε να έχουμε περαιτέρω χρηματοδότηση σε τοπικό επίπεδο. Επομένω, α μην γκρινιάζουν τα κράτη-μέλη και να ζητούν δίθεν τα λεφτά πίσω. Παρακαλώ, το ίδιο να κάνουν ε, όπω κάνω εγώ για το Βέλγιο και οι άλλε. χώρε. οι άλλοι, οι άλλοι συνέχεια με τι άλλε χώρε τώρα, όσον αφορά την τεχνική αρρωγή. Ε, θα, πρέπει να το δούμε αυτό. Ο ρόλο μα είναι να προσπαθούμε να επενδύσουμε σε τοπικό επίπεδο. Να, τι πρέπει να γίνει. Και θα πρέπει και να έχουμε μια σχετική τροπολογία. Ευχαριστώ πολύ. 14 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, το μεσημέρι στις 12, λίγουν οι προθεσμίες για την κατάθεση τροπολογιών. Ευχαριστώ και προχωρώ στο σημείο 7 με τον κύριο, τον κύριο Φράνκο ως συζητητή, στον οποίο δίνω μέσω στο λόγο. Έχετε το λόγο κύριε Φράνκο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στις 23 Ιουνίου Είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το πρόγραμμα δράση Ευρωπαϊκή Ένωση σχέση με την χημική, βιολογική, ραδιολογική και πυρηνική ασφάλεια. Δεν πρόκειται να σα κρατήσω ε, σήμερα, δεν πρόκειται να με γρηγορήσω. Έχω συζητήσει με αρκετού παράγοντε στον τομέα αυτό. Θα έχετε δει το σχέδιο τη γνωμοδοτήσεω ε, που στηρίζεται σε τέσσερι βασικού άξονε. Καταρχά, το νεφή συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και αμοιβαία διάθεση μέσων και ικανοτήτων στον τομέα αυτής της ασφάλειας. Δεύτερον, δημιουργία μιας πραγματικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον κλάδο της πολιτικής ασφάλειας, γιατί παραμένει κατακαιρματισμένη η αγορά και ιδιαίτερα υπογραμμίζω την ανάγκη για κοινέ προδιαγραφές και διαδικασία πιστοποίησης τεχνολογιών και εξοπλισμού, όπως επίσης και στην ανάγκη να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην καινοτομία και ιδιαίτερα στην ασφάλεια. Επίσης ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την ταξινόμηση των διαφορών ε, υπηρεσιών να εξετάσει ε, τις καταστάσεις των παραγόντων αυτών σε περιπτώσει στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και κυρίως στο βιολογικό και τον ε, χημικό τομέα. Επίσης ζητούμε την δια, αμοιβαία διάθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας και στον στρατιωτικό και στον πολιτικό χώρο και επίσης ζητούμε την κατάρτιση των ειδικών αλλά και του κοινού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έξω από αυτήν χάρη στα κέντρα αριστείας γιατί βέβαια η ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ε, ειδωθεί αποκομμένη από την ασφάλεια στον υπόλοιπο κόσμο, λόγω της υπερσυνοριακής διάστασης που μπορούν να προσλάβουν αυτές, αυτοί οι κίνδυνοι, αυτές οι απειλές ε, χημικές, μηχανικές, ε, ραδιολογικές και πυρηνικές. 14 Οκτωβρίου λοιπόν θα έχουμε την ψηφοφορία. Περιμένω τις ε, τροπολογίες των συναδέλφων. Εγώ προσωπικώς θα καταθέσω αρκετές τροπολογίες καθώς στο σχέδιο της νομοδότησης είχα περιορισμό έκτασης για τις ε, προδιαγραφές κατά της διασποράς, αλλά και στην προστασία των προσωπικών και πολιτών δεδομένων των σχετικών με τις ε, επιχειρήσεις ασφάλειας CPRN θα είναι οι τροπολογίες μου και τώρα παρακαλώ ο κύριος Έντσουν λάβει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ καταρχάς τον συνάδελφο για την πρόταση γνωμοδότησης, το σχέδιο γνωμοδότησης. Είναι καλό το κείμενο, μου φαίνεται καλύπτει όλες τις πτυχές. Θα αναφερθώ σε κάποιες πτυχές που εγώ θεωρώ ιδιαίτερες σημαντικές και από την Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη πρέπει πιστεύω να προσδιοριστούν οι αρμόδιοι που θα χειρίζονται τέτοιου είδου. περιστατικά. Και πρέπει να επισημάνουμε ότι ε, υπάρχουν περιστατικά τα οποία ξεπερνούν τις ε, δυνατότητες και τα όρια των κρατών μελών και δεν θα μπορούν κάτι να τα καταπολεμήσουν με επαρκή σπόρους στα κράτη ακριβώς ή και λόγω της οικονομικής κρίσης. Άρα, ίσως θα πρέπει να εξεταστεί ε, στο πλαίσιο αυτής της νομοδότησης η και λόγω της οικονομικής κρίσης. Άρα, ίσως θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο αυτής της νομοδότησης η βοήθεια που μπορεί να προσφερθεί από άλλα κράτη-μέλη. Ένα παράδειγμα, εν προκειμένου, η ενεργοποίηση της πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ρουμανία, όπου είδαμε πως έλαβαν μέρος στις προσπάθειές μας και άλλα κράτη-μέλη. Η συνεργασία λοιπόν μεταξύ κρατών μελών έχει στη σημασία για μένα και για την ασφάλεια, για την αντιμετώπιση των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών. Τόσο στον ε, τομέα της έρευνας, όσο και στην ανάπτυξη εργαστηρίων ή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Εδώ πιστεύω ότι και η κοινωνία των πολιτών μπορεί να προσφέρει πολλά, όπως και ο ιδιωτικό τομέας. Αλλά πρέπει να μεριμνούμε ώστε να, να ώστε να μην προκύψουν προβλήματα ασφαλείας στα εργαστήρια αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ρωτώ εάν η Επιτροπή, ο κ. Χάρμαν, θέλει να λάβει το λόγο να προσθέσει κάτι. Όχι. Ε, δύο λεπτά έχετε, εν πάση περιπτώσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν επιμείνετε, επιμείνετε να πω ότι αυτά που είπαν τα μέλη της Επιτροπής τα κατανοούμε. Σημαντικά θέματα και για μας όταν ετοιμάζαμε το σχέδιο δράσης. Την περασμένη φορά εδώ έδωσα κάποιες πληροφορίες. Αφορούσαν στις δραστηριότητε μας για την εκτέλεση των μέτρων. στο το σχέδιο γνωμοδοτήσεως και περιμένοντας και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών, θα ακούσουμε τα σχόλιά σας. Θα τα λάβουμε υπόψη. Και θα σταματήσω. Danke. Franco, möchten Sie noch mal bitte sehr. Ευχαριστώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε συνάδελφε. Όχι, απλώ να ευχαριστήσω τον εξαίρετο συνάδελφο και να του πω ότι θα λάβω υπόψη όσο γίνεται περισσότερο τα όσα είπε. Gut, Σας ευχαριστώ θερμά. Και συμπληρώνω ότι έχουμε στις 2 του την προθεσμία για τις τροπολογίες. Δύο. Ενάτου. Ενάτου Σεπτεμβρίου διορθώνει ο Πρόεδρος. Τι να σας δείξω, την ημέρα, την ημέρα ή το μήνα. 2. Σεπτεμβρίου έστω φθινόπωρο θα γίνει η, η συζήτηση του θέματος. Πώς θα καταφέραμε λοιπόν τώρα και ολοκληρώσαμε πριν ακόμη από την ώρα μας. Δυστυχώς όμως ο προσεχής μας προσκεκλημένος που είχε ο ίδιος περιορισμένο χρόνο του. Ο κύριο Μπάρτ Γκόρντον, πρόεδρο τη Επιτροπή Επιστήμη και Τεχνολογία Συμβουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, δεν έχει ακόμα εδώ. Η, Επιτροπ... η γραμματεία μα βγήκε ει αναζήτηση ει άγραν του κυρίου Μπάρτ Γκόρντον. Θα διακόψουμε μέχρι να τον εξαναβρούμε, αλλά παρακαλώ μη μου φύγετε. Μη μου φύγετε, λίγοι είμαστε τόσοι άλλως. Καθίστε εδώ. Και είναι σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. το θέμα της συνεργασίας με τις επιτροπές εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ηνωμένων Πολιτειών. Συχνά λέμε στην Επιτροπή μας ότι πρέπει να ενισχυθεί. Μια καλή ευκαιρία τώρα που τον έχουμε. Βλέπω ότι ήρθε και η κυρία Μαντουρέλ. Και οι άλλοι συνάδελφοι δυστυχώ έχουν φύγει. Αλλά ήθελα να ευχαριστήσω, να συγχαρώ μάλλον του Ισπανού συναδέλφου για το παγκόσμιο κύπελο. Όσο και να το λέω με σφιγμένη καρδιά. Θερμά συγχαρητήρια. Μεγάλη επιτυχία σας. That's a problem. Okay, also eine kleine Pause. Bitte um Geduld. Μικρό διάλειμμα λοιπόν και παρακαλώ να δείξετε υπομονή. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συνεχίσουμε τις εργασίες. Καλωσορίζω τον Μπαρτ Γκόρντον, μέλος του Κογκρέσου της Βουλής των Αντιπροσώπων τον είπα Καλώς ήρθατε. Μεγάλη χαρά για μας που ο πρόεδρος Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων μπόρεσε να έρθει εδώ και να μας μιλήσει τιμή για εμάς. Δύσκολο να ρυθμίσουμε τις ημερομηνίε, δύσκολο να βρούμε μια ημερομηνία που μας ικανοποιεί. Είναι πολύ καλό ότι μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας σήμερα το θέμα συνεργασίας πολιτικών των Ηνωμένων Πολιτειών με Ευρωπαίους πολιτικούς είναι επίκαιρο, σημαντικό και σημαντικό και για το μέλλον. Και γι' αυτό χαιρόμαστε και δεχτήκαμε την προσφορά σας και χαιρόμαστε που θα περάσουμε 45 λεπτά μαζί σας συζητώντας. Κύριε Γκόρντον, θα σας δώσω το λόγο, θα δώσω τη δυνατότητα να τοποθετηθείτε. Να μας μιλήσετε και μετά θα συζητήσουμε. Και θα έχουμε 45 λεπτά περίπου στη διάθεσή μας συνολικά. Ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Ξεκινάμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, σαν εισαγωγή. Μακάρι να τα είχα ακούσει όλα. Δεν είχα αφορέσει εγκαίρω τα ακουστικά και στα αξιότιμα μέλη τη Επιτροπή Βιομηχανία και Έρευνα. Και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σα που ήρθα εδώ και να σα μιλήσω και να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων. Είχα τη δυνατότητα να είμαι με τον πρόεδρο Μπούζεκ περίπου εδώ και μια μισή εβδομάδα. Ήταν στη Ουάσιγκτον και συζητούσαμε τη συνεργασία Ευρωπαϊκή Ενώσεω Ηνωμένων Πολιτειών. Και στο τέλο των συζητήσεων μου ρώτησε κατά πόσο ενδιαφερόμουν εγώ για τη συνεργασία Ευρωπαϊκή Ενώσεω και είπα και τη διατλαντική συνεργασία. Είπα ότι εγώ είχα 9 χρονική κόρη που αγαπώ και υποψιάζομαι ότι εκείνοι όπως και τα δικά σας παιδιά ή τα εγγόνια σας θα μπορούσαν να κληρονομήσουν εθνικό επίπεδο διαβίωσης που είναι χαμηλότερο από των γονιών της αντιστροφή του αμερικανικού ονείρου που αποκαλούσαμε, αλλά είναι και δικό σα όνειρο πιστεύω. Γιατί, διότι είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, οι μισοί από αυτού που εργάζονται βγάζουν λιγότερο από 2 δολάρια την ημέρα. Οπότε σίγουρα δεν θέλουμε να ανταγωνιζόμαστε όσον αφορά τα ημερομίστια, τα εργατικά. Θέλουμε να εργαστούμε με πιο παραγωγικό τρόπο και γι' αυτό με ενδιαφέρει τη συνεργασία με την Ευρώπη. Μερικέ από τις χώρες που έχουν χαμηλά ημερομίσθια επενδύουν πάρα πολύ στην τεχνολογία και την έρευνα καθώς και στη χρήση του μεγέθους τη αγοράς τους για να αποκτήσουν ε, μεταφορά τεχνογνωσίας και καμιά φορά προσπαθούν τα δικά τους πρότυπα να τα κάνουν διεθνή και στι δικέ προδιαγραφές. Άλλες χώρες είναι μεγάλη εξαγωγή ενέργεια και ανησυχώ διότι αυτέ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τι εξαγωγέ αυτέ ούτω ώστε να επηρεάσουν τον ασφαλή φοδιασμό σε ενέργεια. Εμεί, η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολλού κοινού στόχου, αξίε και επίπεδα διαβίωση και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε αμοιβαία ωφέλη από τη συνεργασία μα. Κυρίω σε τομεί όπω είναι η έρευνα, να μην δημιουργούμε ωφέλη εκείνου που διαθέτει ένα προϊόν προ αγορά, αλλά να ωφεληθούμε όλοι. Είχαμε κοινά ωφέλη όπως την ενεργειακό αφοδιασμό, αλλαγή του κλίματος για τα κοινό, καθαρό νερό και την ε, βιωσιμότητα του πλανήτη. Είναι κοινή στόχη. Ποιοι είναι οι φραγμοί για τη συνεργασία σαν νομοθέτες. Πρώτα απ' όλα, ο εκτελεστικό κλάδο συνήθω είναι το όχημα για τι ε, διάφορε συμφωνίε και την επιλογή των συμφωνιών. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει εποπτεία, παροχή συμβουλών και θέσπιση νομοθεσία στον ίδιο κλάδο. Η γλώσσα επίση δημιουργεί ένα πρόβλημα. Όμω με τι συνθήκε τη Αβώνα τώρα είναι ευκολότερο η ΕΠΑ, το Κογκρέσο τον ΗΠΑ να έχει ένα σημείο επαφή και να έρχεται σε επαφή με πολλά κοινοβούλια. Πριν ήταν δύσκολο να ε, μπορέσει κανεί να πλοηγήσει μεταξύ των διαφόρων κοινοβουλίων. Στα 26 χρόνια μου στην ανταλλαγή αυτή συνεργασία τη κοινοβουλευτική θεώρησα ότι μεγαλύτερο φραγμό για συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι η έλλειψη ευθυγράμμιση των συζητήσεων των μελών με, την, ε, με τον νομοθετικό κλάδο. Θα ήταν ενδιαφέρον να συζητήσουμε σήμερα ε, κοινό συντονισμό των κανόνων που θα χρησιμοποιούνται για την εποπτεία των μεγάλων χρηματοστικών ε, ιδρυμάτων. Όμως ούτε η δική σας επιτροπή ούτε η δική μας έχει ε, νομοθετική εξουσία σε αυτό το τομέα. Δεν θα προχωρούσαν πολύ. Πιο παραγωγικό θα ήταν να ευθυγραμμιστεί η νομοθεσία με τους εφικτούς στόχους ξεκινήσαμε με, το, με την Επιτροπή Τεχνολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Έγιναν παράλληλες ακροάσεις όσον αφορά τις, για τους γενετικά του οργανισμούς. Η Επιτροπή Επιστήμης και Τεχνολογίας εξέτασε μακροπρόθεσμο που έγινε όσον αφορά την έρευνα και τεχνολογία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξέτασε θέματα διεθνούς για Θα παραγάγουμε μια κοινή έκθεση σύντομα, την οποία θα σας δώσω στην Επιτροπή σας και νομίζω ότι υπάρχουν και διάφοροι άλλοι ενδιαφέροντες τομείς που μπορούν να εξεταστούν από κοινό. Ένα κοινό σύνθημα είναι τα διάφορα ορυκτά και στατικικά υλικά. Η πρόσφατη ομάδα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έκθεσή τη, καθώς και μια έρευνα γεωλογική των ΗΠΑ δείχνουν ότι η Κίνα έχει 90 με 95% όλων των, της παραγωγής σπανίων ορυκτών. Και είδαμε αρχικά ότι ήθελαν να περιορίσουν τι εξαγωγέ. Είχαμε αυτέ τι υποψίε και αυτό ανησυχεί και τι δύο οικονομίε μα, διότι τα σπάνια ορυκτά σε πολύ μικρέ ποσότητε έχουν σημαντική, παίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση απόδοση διαφόρων ενεργειακών πηγών εναλλακτικών στην τηλεπικοινωνία και τα σχετικά προϊόντα και για άλλε χρήσει που θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα σπάνια υλικά, τα ορυκτά. Αν θεωρείτε ότι θα είναι υποφελέ αμοιβαία να έχουμε παράλληλε ακροάσει, θα χρησιμοποιούσα αυτό το μοντέλο για να ενθαρρύνω και άλλους πρόεδρους επιτροπών να κινηθούν από κοινού στις αρμοδιότητές τους. Ένας πρόεδρος μου είπε ότι στα πνευματικά δικαιώματα είναι κάτι που τον ενδιαφέρει. Και ο πρέσβης Κονάρτ θα ήθελε να ξεκινήσει συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφαλείας. Και τελικά ευχαριστώ τον Χαρτ Μπούντενχόφερ και την Επιτροπή και τη Γραμματεία της Ήτρε για τη βοήθειά της να οργανώσει ανταλλαγή προσωπικού για να καταλάβουμε καλύτερα σε επίπεδα προσωπικού πώς λειτουργούν οι αντίστοιχε επιτροπές μας και θα ήθελα εν κατακλείδη να πω ότι η μακρά φιλία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης έχει προφανείς καταγωγές όταν οι γονείς, οι παππούδες, οι Αμερικανοί ήταν, είχαν γεννηθεί στην Ευρώπη αυτοί που ήταν στην Αμερική. Οπότε υπάρχουν πολιτισμικές ομοιότητες αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις που δεν ανήκουν σε μια ήπειρο, σε μια χώρα, είτε συζητάμε το μέλλον των ενεργειακών πηγών, είτε την προστασία των απειλών όσον αφορά τον κυβερνοχώρο και την αλλαγή του κλίματος και πιστεύω γι' αυτό ότι θα, όταν φίλοι δουλεύουν μαζί, ενισχύουν ένα τον άλλον. Ευχαριστώ ξανά κύριε Πρόεδρε Ρόιλ και με τα χαράς να ακούσω αν υπάρχουν ερωτήσεις ή προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκόρντον, για αυτή την σύντομη αλλά πλήρη παρουσίαση. Μας δώσατε κάποια πρακτικά παραδείγματα που δείχνουν ότι πραγματικά έχουμε κοινά προβλήματα, οπότε γίνεται όλο και πιο αναγκαίο να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ε, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης όσον αφορά τις πρώτες ύλες, ενέργεια, τυποποίηση, πνευματικά δικαιώματα είναι όλο θέμα που, θέματα που μας απασχόλησαν τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες και θα εξακολουθούν να μας απασχολούν στο μέλλον και θα ήταν σόφρον, θα ήταν πάρα πολύ σόφρον η... εάν υπάρξει συνεργασία, είπα και Ευρώπης. Μεγαλύτερη συνεργασία. Όχι μόνο σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά και σε διακοινοβουλευτικό επίπεδο. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή, γίνονται ήδη πολλές επισκέψεις και ανταλλαγές. Μπορούμε να μάθουμε πολλά ημένα από τους δε όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων σε καθημερινό επίπεδο. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Κάποιοι συνάδελφοι ήδη ζήτησαν το λόγο. Ο πρόεδρος λοιπόν θα πρέπει να πιστοχωρήσει και να αφήσει και άλλους να έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν και να συμβάλλουν στη συζήτηση. Επιτρέψτε μου όμως να, να καλωσορίσω την κυρία Σαβάλα που είναι αντιπρόεδρος κυρία επιτροπή, Κυρία Τζαβέλα καλωσορίζω θα συνεργαστούμε και μαζί σας, είσαστε και μέλος της δικής μας Επιτροπής, όχι μόνο στην αντιπροσωπεία για τη ΣΥΠΑ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μαντουρέλ, η οποία είναι η σοσιαλίστρια συντονίστρια της Επιτροπής, ε, είναι από την Ισπανία και θα πάρει το λόγο πρώτη. Και όπως ξέρετε, η Ισπανία κέρδισε και το παγκόσμιο κύπελο στο ποδόσφαιρο, θα το ξέρετε λοιπόν, φαντάζομαι. Κάποιοι λένε ότι ήταν τυχεροί, κάποιοι λένε ότι το άξισαν, τέλος πάντων συγχαρητήρια στην Ισπανία. Ε, ταξίδευα το βράδυ, είμαι λίγο ζαλισμένος ε, σήμερα το πρωί. Μαντουρέλ, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εσάς κύριε Γκόρντον. Και βέβαια ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στην ε, Επιτροπή μας. Έτσι μπορούμε να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων που είναι τόσο ενδιαφέρουσα για τη δουλειά μας, αλλά επίσης και είναι πάρα πολύ αξιόλογα τα όσα μας λέτε σαν αξιολογήσεις που συμφωνούμε μαζί σας και θέλουμε να υπάρξει και συνέχεια. Οφείλω να σας πω ότι το μοντέλο της δικής σας χώρας για τους τομείς αρμοδιότητας της Επιτροπής μας είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το λάβουμε υπόψη τη δουλειά μας και γι' αυτό και είναι καλό το οποίο σήμερα εμείς μπορούμε από πρώτο χέρι να μάθουμε τι γίνεται και έτσι να μπορούμε να σας πούμε και κάποια ερωτήματα που έχουμε. Εγώ δε θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στην πολιτική έρευνα και ανάπτυξης, μια πολιτική στην οποία έχετε μια μακρά παράδοση ε, σε σχέση και με κάποιες πρωτοβουλίες που υπάρχουν και στις οποίες έχετε ε, πετύχει κάποια θετικά αποτελέσματα και έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου προσπαθούμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την επιστημονική πολιτική. Έχουμε το πρόγραμμα πλαίσιο το οποίο το ξέρετε πάρα πολύ καλά και σε βάθος οπότε δε αφορά και κάτι που συγκεντρώνει τη Γενική Συνένεση δηλαδή το πώς θα οι διαδικασίες και για τα προγράμματα και για τα παραστατικά που αφορούν τη χρηματοδότηση και τα δικαιολογητικά. Με σημείο αφορά λοιπόν τη χώρα σας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τέτοια προγράμματα, για ένα σύστημα το οποίο να βασίζεται στην εμπιστοσύνη προς τους επιστήμονες. Να θεωρήσουμε ότι δεν γίνεται παρά να αναλυφθούν κάποια ρίσκα και να σταματήσει η γραφειοκρατία ταυτόχρονα. Έτσι να λειτουργήσει το μοντέλο δικό σας μοντέλο για τέτοια πράγματα. Πολλέ φορέ οι αξιολογήσει όταν κανεί βλέπει τα πράγματα απ' έξω είναι καλύτερε. Άλλο τώρα. Χρειαζόμαστε ερευνητέ. Έχουμε πολύ λιγότερου αναχίλιου κατοίκου από όσου τα θέλαμε και από όσου έχετε και εσεί στη χώρα σα από ό,τι είπατε. Οπότε θα πρέπει τώρα να αυξηθεί η περισσότερο για αυτόν τον σκοπό και επίση σταματήσουμε να έχουμε αυτή τη, την τη, τη διαρροή των ερευνητών. Εσείς τι λέτε όσον αφορά τους ερευνητές, τι προγράμματα ε, απέδωσαν για τη δική σας περίπτωση. Επίσης, για πέστε μας επί τη βάση της δικής σας μακράς εμπειρίας, τι γίνεται όσον αφορά την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα για έρευνα και ανάπτυξη. Για πέστε μας τη γνώμη σας, γιατί έχουμε δοκιμάσει κάποια πράγματα. Αλλά για πες μας εσείς τι θα αλλάζετε όσον αφορά το δικό σας πρότυπο. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν στο έργο μας. Και φυσικά και θα είναι θετικά για την μέλουσα συνεργασία μας. Θα απαντάτε κάθε φορά. Ναι. Εάν είναι τόσε πολλέ ερωτήσει, μάλλον καλύτερα να απαντάω στην κάθε μία χωριστά. Είναι πολλές ερωτήσεις της ε, συναδέλφου. Καταρχά επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι οι επιστήμονες σε όλε τι χώρε θεωρούν ότι είναι υπερβολική η γραφειοκρατία εκτεταμένη και αυτό είναι ένα ζήτημα που βλέπουμε παντού. Ένα άλλο ζήτημα που θέσατε είναι οι νέοι μα. Το ίδιο πρόβλημα μα απασχολεί και εμά Στα τέλη τη δεκαετία του 50 όταν ε, εκτόξευσε το Sputnik ε, η Σοβιετική τότε Ένωση, οι ε, Ηνωμένε Πολιτείε έπαθαν σοκ. Εμεί νομίζαμε ότι είχαμε μια τεχνολογία προηγμένη και ξαφνικά αισθανθήκαμε φόβο για την ίδια μα την ασφάλεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο παρακολούθησα εγώ από το Κογκρέσο. Αλλά εκτός από το Κογκρέσο και η ΝΑΣΑ επίσης έδινε ε, ελπίδες για μια ολόκληρη γενεά επιστημόνων, οι οποίοι όμως τώρα πλέον ε, δεν έχουν περάσει βέβαια οι γενές και δεν βλέπουμε να αντικαθιστούνται από την τωρινή γενεά. Γι' αυτό μας απασχολεί το ερώτημα το τι θα συμβεί με τους νέους μας. Και το 2005 που είχα μια σχετική συζήτηση στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών, νομίζω ότι είναι σχετικό το θέμα αυτά που λέτε, ε, ζήτησα μια έκθεση για τους νέους και την τεχνολογία και την επιστήμη στη δεκαετία του 2020. Πώς μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξη. Και μου είπαν ότι εάν συνεχίσουμε με το ρυθμό που πάμε, θα τα βρούμε σκούρα στο μέλλον. Και για τις επενδύσεις για την έρευνα, οι ομοσπονδιακές επενδύσεις ήταν πολύ χαμηλές. Ο ιδιωτικός τομέας ο είχε μάλλον φθήνουσες επενδύσεις στην έρευνα και αυτό τουλάχιστον δική μου γνώμη είναι ότι οφείλεται στις, ε, στην απόλυτη εξάρτησή τους από τις τριμενιαίες εκθέσεις επιτυχίας και έτσι δεν τολμούν οι επιχειρήσεις να κάνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις γιατί φοβούνται ότι το επόμενο τρίμηνο δεν θα φανεί η επένδυση στις, ε, στους συλλογισμούς. Γι' αυτό στις εκθέσεις. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει και να επενδύσουμε τα διπλάσια για την έρευνα μέσα σε μια δεκαετία, μακροπρόθεσμα δηλαδή, και να έχουμε τη σχετική νομοθεσία, πράγμα στο οποίο έχουμε προχωρήσει ήδη βέβαια, αλλά πρέπει επίση να πω ότι με τι ε, δεινέ οικονομικέ συνθήκε που αντιμετωπίζουμε θα είναι δύσκολο να επιτύχουμε τόσε υψηλέ επιδόσει επενδυτικέ. Επίση, μου είπε η Ακαδημία των Επιστημών ότι τα παιδιά μα έχουν χαμηλέ επιδόσει στι φυσικέ επιστήμε, τα μαθηματικά κτλ. Τα μισά σχεδόν τη μισή σχεδόν επιτυχία από τα δικά σας παιδιά στην Ευρώπη. Ψάχναμε να βρούμε ποιο είναι ο λόγο. Ε, δεν είμαστε λιγότερο έξυπνοι από σε τελευταία ανάλυση από σα είμαστε. Ε, τα 50% λοιπόν, των ε, καθηγητών της μέσης εκπαίδευσης δεν είχαν την ειδίκευση για να διδάξουν μαθηματικά. Δεν είχαν πολλέ φορέ πτυχίο μαθηματικών σχολών. Ούτε των φυσικών επιστημών. Δεν είχαν το υπόβαθρο, δεν είχαν το πτυχίο αλλά τι θα, άρα τι θα διδάξουν, πώς θα εμπνεύσουν τα παιδιά αυτό. Ένα παράδειγμα πολύ σύντομα. Ο πατέρας μου ήταν αγρότης. Ήρθε ο πόλεμος, επιστρατεύτηκε, γύρισε πίσω με το λεγόμενο πιστοποιητικό του GI, που ήταν το, ε, το χαρτί από την ε, αποστρατεία, και θέλησε να σπουδάσει να μην είναι πια αγρότη. Η γυναίκα του όμω, η μητέρα μου έχασε τη δουλειά τη, ο ίδιο αναγκάστηκε να πιάσει δεύτερη δουλειά πέραν της των ενεργικών εργασιών για να μπορέσει να ε, συντηρήσει την οικογένεια και η δουλειά που βρήκε ήταν δάσκαλο στο σχολείο και μάλιστα δάσκαλο φυσική αγωγή πήγε να μάθει μπάσκετ χωρίς τα παιδιά, μπάσκετ που ο ίδιο δεν γνώριζε. Ε, το ίδιο πράγμα κάνουμε ύστερα από 40-50 χρόνια. Φαίνεται ότι δεν έχουμε πάρει τα δάγματα του παρελθόντος. Ναι, μεν εκπαιδεύουμε καλού δασκάλου, αλλά δεν του δίνουμε υπόβαθρο και γνώσει ειδικά στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες κτλ. Έτσι λοιπόν δώσαμε την ευκαιρία με ένα σύστημα υποτροφιών στι θερινέ του διακοπέ αυτοί οι δάσκαλοι να κάνουν την εξειδίκευση στα μαθηματικά και τι φυσικέ επιστήμε για να ενισχύουν τι γνώσει και το υπόβαθρό του, την ειδίκευσή του. Το ίδιο με ένα πρόγραμμα για ε, ενίσχυση της παραμονής των δασκάλων και καθηγητών τη μέσης εκπαίδευση και για να μένουν πιο πολλά χρόνια, γιατί συνήθω μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια οι δάσκαλοι φεύγουν από τα σχολεία. Επίσης αναζητήσαμε εκείνου οι οποίοι έχουν, ε, έχουν ειδίκευση στα, στα μαθηματικά ή στι επιστήμες επιστήμε, θετικέ επιστήμε, που όμως απασχολούνται κάπου αλλού, στο στρατόφερη, πίνει αλλού, για να τους προσελκύσουμε στα σχολεία. Ελπίζω αυτό σαν λύσει να σας εμπνεύσει και εσάς ε, πρέπει δεν να σημειώσω ότι στην εκπαίδευση να δώσουμε το βάρος. Οποτεδήποτε εμείς είδαμε στην Επιτροπή μας ε, επιστήμονες και μάλιστα βραβευμένους με βραβεία Νόμπελ που ήρθαν μερικές φορές να μας μιλήσουν, πάντοτε μας έλεγαν ότι την έμπνευση τους την άντλησαν από τους δασκάλους και τους καθηγητές τους. Όσα λεφτά και να δώσουμε λοιπόν στην εκπαίδευση δεν αρκούνε εάν δεν έχουμε τις καλές ιδέες, εάν δεν έχουμε τους καλούς δασκάλους. Και πρέπει το χρήμα που διατίθεται να το αξιοποιήσουμε στο δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Είδαμε ότι υπάρχουν 25 διαφορετικές υπηρεσίες που ασχολούνται με την ε, έρευνα στην ανατεχνολογία, εκ των οποίων οι 15 είχαν άμεση χρηματοδότηση, οι 10 είχαν ε, να ασχοληθούν με, την, ε, με τις διατάξεις, την νομοθεσία κτλ. Και έτσι ορίσαμε ένα συντονιστικό όργανο μεταξύ αυτών των υπηρεσιών, ελπίζοντας ότι θα εξασφαλίσουμε τη συνεργασία μεταξύ τους και το συντονισμό, ίσως μεταξύ των κρατών μελών. Θα μπορούσατε να ε, κάνετε κάποια αντίστοιχη ε, προσπάθεια, ένα συντονιστικό όργανο. Επίσης, ορίσαμε, διορίσαμε και ένα συμβουλευτικό όργανο για την ε, από πλευρά τη βιομηχανία, ε, δηλαδή ε, ένα συμβουλευτικό όργανο, δεν είμαστε δεσμευμένοι από τι προτάσει του, το οποίο θα μα έλεγε προ τα που θα ήταν σκόπιμο να αξιοποιηθεί η έρευνα που έχουμε στη θέση μα. Να δούμε πού μπορεί να, έχει, να πιάσει περισσότερο τόπο. Άρα, ο ιδιωτικό τομέα μα λέει Φερρυπίν, αυτή η τεχνολογία, εάν καταφέρετε να την προχωρήσετε κτλ. Εμείς βλέπουμε αυτές και εκείνες τις εφαρμογές. Κάποια προγράμματα συγκεκριμένα που χρειαζόμαστε για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων είναι αυτά και αυτά. Αυτό είναι ένα καλό τρόπο να αξιοποιήσουμε καλά τα, τα δημόσια χρήματα και βέβαια να εμπλέξουμε και τον ιδιωτικό τομέα. Από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει η βούληση για ανεξαρτητοποίηση από την ενέργεια. Υπάρχει μια υπηρεσία ομοσπονδιακή η οποία ονομάζεται DARPA και είναι εκείνη η οποία ανέπτυξε την τεχνολογία εχμή το GPS, το Γαλιλαίο, όλα αυτά. Ο δε λόγος για τον οποίο επέτυχε στι προσπαθίε της είναι ότι ήταν οι επιχειρήσει της υψηλού κινδύνου και υψηλή ανταμοιβή. Και από ό,τι βλέπω από τους Ευρωπαίους φίλους, η τάση είναι εδώ μάλλον να μην λαμβάνεται, να μην αναλαμβάνεται κίνδυνο. Ή αν κανείς ε, ανέλαβε κίνδυνο και ε, χρεοκόπησε, συνήθως δεν έχει άλλη δεύτερη ευκαιρία να αναπτύξει δραστηριότητε το να αποφεύγουν κτλ. Ε, αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε από πλευράς κυβέρνηση να συμβάλλουμε με μικρή συμβολή κάθε φορά με την ελπίδα ότι μπορούμε να συμβάλλουμε σε εναλλακτικέ μορφέ ενέργεια, και τέτοια πράγματα και έτσι θεσπίσαμε μία υπηρεσία που αντιγράψαμε από την Τάρμπα ε, για το τομέα της ενέργειας, γνωρίζοντας ότι με υψηλό κίνδυνο μπορεί κανείς να έχει και υψηλή απόδοση, υψηλά, καλά αποτελέσματα. Και χωρίς να θέλω να σας καθυστερήσω περισσότερο τώρα, θα ήθελα να πω ότι είναι χρήσιμο ένα τμήμα του προπολογισμού σας να το ορίσετε για κάτι τέτοιο. Εγώ ζητώ, επαραδείγματι, από τη συγκεκριμένη αυτή, στο ε, συγκεκριμένο αυτό το τομέα ένα κομμάτι του προπολογισμού να, να αφιερώνεται ειδικά σε αυτή την υπηρεσία υψηλού ε, κινδύνου και υψηλών αποτελεσμάτων στην έρευνα. Ο κύριος Ρούμπι το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θερμά. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ χρήσιμε η και τα αλλαγή απόψεων. Πολύ σημαντική για όλους μας. Συναντηθήκαμε βέβαια και στο παρελθόν στι ΗΠΑ. Είναι καλό πάντα να έχουμε αυτή τη συνεργασία στον ε, μεγαλύτερο τομέα των οικονομικών των οικονομικών προγραμμάτων, να μπορούμε δηλαδή να κάνουμε επενδύσεις, ναι, ε, ναι, ναι, να βρίσκουμε, τις, ε, τα προβλήματα που μπορούμε να επικοινωνήσουμε, που μπορούμε να συνεργαστούμε στην έρευνα για την ηλιακή ενέργεια, για τη σύνδεξη. Όλα αυτά τα μεγάλα προγράμματα τα οποία βέβαια μας καθοδηγούν για το μέλλον, ε, τα οποία ακολουθούμε με ενθουσιασμό, αλλά και όπου θέλουμε να αναπτύξουμε τις νέες ε, δομές και τις νέες οργανώσεις. Ταυτόχρονα mm. υπάρχει και η άλλη πτυχή, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι τα μεγάλα σχέδια, αλλά οι μικρέ και μεσέ επιχειρήσει, τι οποίε θέλουμε επίση να ενισχύσουμε για την έρευνα και τεχνολογία. Εδώ τι μπορείτε να μα συμβουλεύσετε, ο πρόεδρο. Κοιτάξτε να σας πω, έχω πολλούς εγγεγραμμένους στον κατάλογο για τις ερωτήσεις. Αν είναι καλύτερο να απαντήσετε σε αρκετούς συναδέλφους μαζί. Η κυρία Χέρτσοκ έχει το λόγο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και τον κύριο Γκόρντον που ήρθε για να μας πει τις απόψεις του. Πάντοτε είναι καλό να μιλάμε από ανθρώπους που έρχονται από την έρευνα γιατί τα βρίσκουμε μαζί τους. Γιατί όταν τα λέμε με τους, τους υπουργούς οικονομικών και τους σχετικούς δεν τα βρίσκουμε. Είναι εκείνοι οι οποίοι σκοτώνουν τις ιδέες μας. Άρα θέλουμε στην επόμενη δεκαετία να έχουμε διπλασιασμό των όσων δίνουμε για την έρευνα. Να δούμε αυτό πώς θα περάσει τους υπουργούς οικονομικών. Τώρα όσον αφορά την διαχείριση των οικονομικών αυτό πρέπει να κάνουμε είναι ε, το όραμα ίτερ, το τι θα γίνει για τις υποδομές. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Εδώ στις συζητήσεις μας είπα τι λένε όσον αφορά το μέλλον της ε, ενέργειας και το καντάς. Επίσης, υπάρχουν κάποια βασικά θέματα τα οποία ίσως είναι αμοιβαίων ενδιαφέροντος. καλύτερα να έχουν προσέγγιση βάσει της αποδοχής του ρίσκου παρά της αρχής της ε, σοφροσύνης. Επίσης, τι λέτε για την κλωνοποίηση και τα θέματα, τις επιστήμες που έχουν σχέση με τη ζωή, γιατί εδώ υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά βασικά θέματα. Οι ερευνητές πάντοτε είναι ένα βήμα μπροστά και για τα ηθικά. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Γκόρντον. Νομίζω ότι είναι χρησιμότατο το να συνεργαστούμε όπως είπατε κι εσείς και να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με τη χώρα σας κυρίως ευθυγράμμιση επί εργασιών και στόχων αποτελεσμάτων. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και τις δικές μας εργασίες. Πρέπει να επικεντρωθούμε επί κάποιου θέματος που είναι σημαντικό πριν αναφερθήκατε στην έρευνα. Είπατε τρεις φορές όμως αναφερθήκατε στην ασφάλεια. Ασφάλεια όσον αφορά την έρευνα. Αναφερθήκατε στην έρευνα όσον αφορά τον τομέα της πληροφορικής. Μπορούσαμε να μιλήσουμε για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλα. Ερώτηση. Θέλουμε να δώσουμε ασφάλεια, αλλά και θέλουμε και σεβασμό της ιδιωτικής ζωής. Αναφέρθηκε σε ηθικά θέματα συνάδελφος πριν. Αυτά είναι δύο πράγματα αλληλένδετα. Θέλουμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια από τη μια και να σεβαστούμε την ιδιωτική ζωή από την άλλη. Αυτό είναι κυρίαρχο θέμα, θεμελιώδες. Κύριε Πρόεδρε, Ποια είναι η άποψή σας για να καταλάβω που βρίσκεται η ισορροπία, μέχρι πού μπορούμε να σπροχτούμε, να προωθήσουμε και πού μπορούμε να αφήσουμε να χαθεί λίγο η ασφάλεια για να σεβαστούμε οι ίδιοι την ιδιωτική μα ζωή και τους εαυτούς μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ουντή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και σας κύριε Κόντο που ήρθατε τον Τζο Μπάιντεν τον είχαμε δείχνει πρώτη τον είπα στην, ε, στο ημικύκλιο και είδαμε κάποια αλλαγή. Αλλαγή τόνου της Αμερικανικής κυβερνήσεως. Και βλέπουμε ότι δημιουργούνται νέες σχέσεις. Μεγάλη, οι ε, μεγάλες προκλήσεις της ανθρωπότητας επηρεούνται από την επιστήμη. Και θέλω την άποψή σας για δύο πράγματα. Εμείς Ευρωπαίοι θέλουμε να πολύ την πνευματική ιδιοκτησία. Έχουμε πρόβλημα περιφερειακό που είναι πρόβλημα των γλωσσών και είναι πρόβλημα ρυθμίσεως των γλωσσών όσον αφορά το δίπλωμα Ο Μισελ Μπαρνιέ, ο επίτροπος εσωτερικής αγοράς, θέλει να συμφωνήσουμε με τριών γλώσσων όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Ποια είναι η θέση σας? Κυρίως έναντι των Κινέζων και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεύτερον, κρατικές ενισχύσεις για τα μεγάλα επιστημονικά προγράμματα. Γίνονται, υπάρχουν διαφορές μεταξύ Boeing και Airbus, γίνονται δίκες στο ΠΟΕ για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται από τη ΣΥΠΑ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχασε στο πρώτο βάθμιο η Airbus. Θα δούμε τι θα γίνει με την Boeing. Λοιπόν, σχέση ιδιωτικού δημόσιου τομέα όσον αφορά την πρόοδο στον επιστημονικό τομέα. Θα ακούσουμε ακόμη μία παρέμβαση. Ο κύριος Μπιτσικόφερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω, Πρόεδρε, ότι έτσι έχουμε πολύτιμη ευκαιρία με την ανταλλαγή των απόψεων. Τώρα που έχουμε την να μιλήσουμε με τον επερχόμενο πρόεδρο της Επιτροπής αυτής, τον κύριο Γκόρτον, ο οποίος έχει εμπλακεί με τον ε, διατλαντικό νομοθετικό διάλογο τόσο πολύ καιρό και ήρθε σήμερα να μας δει στην Επιτροπή μας και για άλλη μια φορά. Ε, γίνεται μια μηχανή για καλύτερη συνεργασία μεταξύ του δικού μας Κοινοβουλίου και του Αμερικανικού Κογκρέσου μια που θεωρώ ότι επίσης αυτό αποτελεί απόδειξη του γεγονότος το ότι με την συνθήκη της Λισαβόνας και την έναρξη τη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να είναι ένας σημαντικός παίκτη για πολλά ζητήματα και επομένως ε, αξίζει να συνεργάζεται κανείς μαζί του και διαπιστώνω ότι τώρα έχουμε ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα γιατί ό,τι χρειάζεται να υπάρχει μια ευρύτερη συνεργασία και όχι μόνο μεταξύ της δικής σας και της δικής μας Επιτροπής αλλά μεταξύ όλων των επιτροπών των κοινοβουλευτικών των δικών σας και αυτού εδώ του Κοινοβουλίου και ακριβώς όπως αναφέρατε και εσείς έχουμε μια σειρά ζητημάτων τα οποία θα πρέπει να τα θέσουμε επιτάπητος για να ενδυναμώσουμε αυτή μας την συνεργασία και να μπορούμε να απευθυνθεί ο, ο ένας στον άλλο που είναι κάθε φορά αρμόδιος και έτσι να περνάνε τα θέματα αυτά από τη διατατική συνεργασία και να κάνουμε ακόμα ευρύτερε ανταλλαγές προσωπικού, να έχουμε κοινέ ακροάσεις και επίσης περιμένουμε εναγωνίως πώς το επόμενο κογκρέσο θα φτιάξει μια υπηρεσία στις Βρυξέλλες, όπως έχουμε εμείς μια υπηρεσία στην Ουάσιγκτον. Και έχουμε πολλά θέματα από τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η συνεργασία και από τους μεν και από τους δε. Και έτσι να μπορούμε να έχουμε καλύτερη κατανόηση. Να εξυπηρετήσουμε έτσι καλύτερα τους πολίτες. Και θέλω να σταθώ στην πρότασή σας για κάποια σπάνια ορυκτά και μέταλλα. Είναι κάτι που είναι θέμα καυτής επικαιρότητα και στατικής σημασίας. Να κάτσουμε για να τόσο το διαφορά μας όσο γίνεται περισσότερο σε αυτό το θέμα. Όπως κάνουμε και για τη νέα τεχνολογία. Την χρήση cradle του cradle και looping. Να ωφεληθεί τη βιομηχανία ακριβώ όπως λέμε για την ανοτεχνολογία, το αέριο cell. Είναι το αέριο από κάποια πετρώματα. Και έτσι να μπορούμε να γίνουμε ε, ατμομηχανοί που θα προωθήσει όλα τα θέματα τα οποία κρυβούν στην ατζέντα μας. Ευχαριστώ, έχετε το λόγο. Ας προσπαθήσω όμως να πιο σύντομος, γιατί καλύψαμε πολλά θέματα εδώ. Ε, επιχειρήσεις ε, και δομ, επιχειρηματικότητα μάλλον και δομές. Αυτό στηρίζεται περισσότερο σε αυτό που ονομάζουμε εθνικά εργαστήρια, που έχετε και εσείς ασφαλώς στην πανεπιστημιακή μας έρευνα επίσης και έχουμε προσθέσει ένα ακόμη στοιχείο με τους, με τους νόμους. Οργανώνουμε λοιπόν γύρω από ένα πανεπιστήμιο ή εθνικό εργαστήριο ε, δομές για ένα συγκεκριμένο τομέα, φερειπίν την ηλιακή ενέργεια και εκεί μαζεύουμε τους πιο καλούς, τους πιο λαμπρούς επιστήμονες που θα ασχοληθούν με την ηλιακή ενέργεια. Αλλά επίσης χρειάζεται και κάποια πρόοδος φερειπίν ή κάποια ρηξικέλευτη επιλογή όπως φερειπίν ε, συνδυασμός της νανοτεχνολογίας με την ηλιακή ενέργεια. και εκεί έχουμε τα λεγόμενα μεθοριακά κέντρα. Δηλαδή εκεί έχουμε για ε, συγκεκριμένο στόχο το συνδυασμό δηλαδή τεχνολογίας με την ηλιακή ενέργεια και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τους πιο λαμπρούς επιστήμονες και τους ζητούμε να ασχοληθούν με αυτή τη ε, ζώνη μεταξύ των δύο κλάδων. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερη σημασία τους δίνουμε και προσπαθούμε να τις ενισχύσουμε με διάφορους τρόπους στις προσπάθειές τους. Έχουμε φέρει φερειπίν μία επιδότηση για παραγωγή φερρυπίν του τάδε προϊόντος ε, με, την, με μια συγκεκριμένη τεχνολογία, εν, μια ένα ποσοστό αυτής της επιδότησης πηγαίνει αποκλειστικά και μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που μπορούσα επίσης να προσθέσω είναι ότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται κάθε πολιτεία, το λεγόμενο πρόγραμμα MEP, το οποίο έχει τον εξή σκοπό. Ορισμένε μικροεπιχειρήσει μπορεί να μην έχουν αρκετού πόρου για γραφίστα, για οικονομολόγο, για μηχανολόγο μηχανικό. Έχουμε λοιπόν μια ομάδα των ειδικών αυτών από τους διάφορους τομείς, η οποία είναι διαθέσιμη και προσφέρει τις υπηρεσίες της στη μικρομεσαία επιχείρηση. Το ποσοστό το ορίζει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, δύο τρίτα από την τοπική κοινωνία και ένα τρίτο από την Ομοσπονδιακή Δομή, αναλόγως. Κάποιο λοιπόν ο οποίο δεν μπορεί να έχει το γραφείο στα διάθεσή του συνέχεια στην επιχείρησή του, μπορεί απευθυνόμενο σε αυτή την ομάδα να αξιοποιήσει τι υπηρεσίε κάποιου γραφίστα, ενδεχομένω με έκπτωση κτλ. για τις τεχνολογίες. Η σύνθηξη, είμαι σίγουρο ότι θα κρατήσει αρκετά χρόνια για να την εξασφαλίσουμε, είναι υψηλού κινδύνου και υψηλής απόδοσης τομέας, στον οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Είτε μας ε, φαίνονται προτιμότερες η ηλιακή και η αιωλική ενέργεια, είτε όχι, δεν μπορούμε να λησμονούμε το γεγονό ότι ο ήλιο δεν λάμπει πάντοτε και ο άνεμο δεν φυσάει πάντοτε. Γι' αυτό πρέπει να μα απασχολήσει οπωσδήποτε το ζήτημα τη σύνδεξη. στην διερεύνηση νέων οδών. Βεβαίως μπορεί να έχουμε ε, ζητήματα δεοντολογικά και να μας απασχολούν πάντα στις ΗΠΑ, αλλά μην λησμονούμε ότι όταν υπάρχει κάποιος τρόπος και κάποιος διάβλος, οπωσδήποτε κάποιος τελικά θα τον ακολουθήσει. Δεν μπορούμε να κλείσουμε κάθε ε, διέξοδο δηλαδή. Γι' αυτό καλό θα είναι να επιτρέπουμε την πρόοδο με προστασία βεβαίως των ε, διοντολογικών μας ανησυχιών. Για τη βιοτεχνολογία επίσης νομίζω ότι θα ήταν καλό να συνεργαστούμε μαζί και για τη βιοτεχνολογία και για την νανοτεχνολογία που έχουμε την πρωτοπορία και εσείς και εμείς και να κοιτάξουμε διάφορους τομείς έτσι ώστε να μην επαναληφθεί το πρόβλημα του Μορτζάνο. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα για το οποίο πολλοί έχουν ανησυχίες ε, και επιφυλάξεις. Και πρέπει να έχουμε καλή έρευνα στην τεχνολογία για να ξέρουμε τι επιφυλάξεις υπάρχουν και τι συνέπειες. Ε, ένα παράδειγμα θα σας πω. Εάν βάλετε αμφιλιακή κρέμα, να είστε βέβαιοι ότι έχει στοιχεία νανοτεχνολογίας μέσα της. Επομένως, η ανανοτεχνολογία είναι παρούσα παντού. Για το SWIFT και τα υπόλοιπα θέματα δεν θα συζητήσω αλλά έχουμε μία διαφορά ως προς την αντίληψή μας ορισμένα θέματα, όπως για παραδείγμα στο θέμα του ιδιωτικού βίου στις ΗΠΑ, τον οποίο ασφαλώς και υποστηρίζουμε, αλλά η δική σας περιγραφή του ιδιωτικού βίου να είναι διαφορετική μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα Σήμερα έβλεπα στην εφημερίδα κάποιο νεαρό Γερμανό που μιλούσε για την ε, ε, προστασία του ιδιωτικού του βίου, ενώ ταυτόχρονα είχε όλη του την ε, ζωή στο facebook, συμμετείχε σε διάφορες άλλες αντίστοιχες ιστοσελίδες κτλ. Ε, και όμως έλεγε ότι πρέπει να προστατεύονται προσωπικά του δεδομένα. αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει όλους κατά τρόπο σοβαρό. Αλλαγή τόνου, διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων έχει η παρούσα κυβέρνηση από ό,τι παρθούσα. Εγώ είμαι δημοκρατικό και υποστηρίζω αυτόν τον πρόεδρο. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι ζούμε σε έναν κόσμο μαζί με άλλους και ότι δεν μπορούμε να είμαστε ο cowboy ο οποίος επιβάλλει το τι πρόκειται να γίνει. Και ειλικρινά πρέπει να πω ότι πήγαμε με την αποστολή του Απόλλωνα πήγαμε στο φεγγάρι Εκτό από του Γερμανού επιστήμονες που μας βοήθησαν τότε, μόνοι μας είχαν και με τα δικά μας χρήματα. Μελλοντική διαστημική έρευνα θα είναι πάρα πολύ δαπανηρή. Άρα θα πρέπει να συνεργαστούμε και η απορρόφηση του άνθρακα και η αποθήκευση του άνθρακα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αλλαγή του κλίματος. Είναι κάτι που συζήτησαν οι G8, θα πρέπει να συνεργαστούμε. Όπως λέμε, ε, αυτός που προσπαθεί τα καταφέρνει. Σε αυτούς τους οικονομικούς καιρούς με, με σύννεφο που καλύπτει τα πάντα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε. Όσον αφορά την Boeing και την Airbus, η Airbus είχε το δικό της πρόβλημα, θα δούμε τι θα γίνει με την Boeing. Αν με ρωτάτε προσωπικά, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε εθνικές επενδύσεις για να βοηθήσουμε έναν τομέα, κάποια βιομηχανία θα πρέπει να γίνονται εθνικέ επενδύσεις για να βοηθούν οι επενδύσει στην έρευνα, για να χρησιμοποιηθεί έρευνα από όλου. Κάποιος θα θεωρούσε αυτό σαν όφελος και κάποιο άλλος αν όχι. Πνευματικά δικαιώματα, πάρα πολύ ισχυρό το θέμα αυτό στη ΣΥΠΑ, είναι ένα τομέα όπου χρειάζεται αμοιβαία συζήτηση, είναι πολύ επικαιρό το θέμα στη ΣΥΠΑ και μας προσβάλλει το ότι τα έργα των συγγραφέων μας, των συγγραφέων του θεάτρου, των τραγουδιστών μας, των κινηματογραφιστών μας, όλα αυτά τα έργα βλέπουμε ότι αφαιρούνται. Τα παίρνει και τα αντιγράφει κάποιος. Ελπίζω να συνεργαστούμε σε αυτό το τομέα. Και άλλο θέμα. Η συνεργασία, το ανέφερε ο Ράινχαρτ, το προσωπικό μας να συνεργαστεί και κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει πολλοί ερευνητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γνωρίζουν σε ποιον να απευθυνθούν στη ΣΥΠΑ. Πολύ συχνά γίνεται επαφή πανεπιστημίου με πανεπιστήμιο. Καμιά φορά πάει κανείς στο Υπουργείο Εξωτερικών. Υπήρχε μια, ένας οργανισμός, OSTP, που είναι συμβουλευτικό φορέα τη Γερουσία για τον Πρόεδρο. Και υπήρχε μια υποεπιτροπή η οποία ασχολιόταν με την διεθνή συνεργασία. Και στην προηγούμενη κυβέρνηση ατρόφησε. Δεν χρησιμοποιήθηκε αυτό ο φορέα. Ο Dr. John Holden ζητήθηκε να αποκαταστήσει αυτό το φορέα. Ήδη υπάρχει μια ιστοσελίδα, δεν είναι πλήρη, είναι σε πρώιμο στάδιο, αλλά ελπίζουμε ότι θα υπάρχει αυτή η πύλη στο διαδίκτυο. Αν σας ενδιαφέρει η νανοτεχνολογία κάποιο θέμα, έχετε ένα σημείο να πάτε και μπορούν να σας κατευθύνουν από εκεί και πέρα. Το θέμα του γραφείου στις Βρυξέλλες, σίγουρα αυτό θα έπρεπε να γίνει, είμαστε φίλοι, να σας πω την αλήθεια. Ε, έχω την εξουσία να το κάνω αυτό και την νομοθεσία στο παρόν κλίμα όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο εμείς πολιτικώς να πούμε ότι θα αυξήσουμε τη γραφειοκρατία μας. Οπότε δεν πρόκειται να συμβεί τώρα κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι ο πρέσβης κ. Σκουνάρ Γνωρίζω ότι ο πρέσβης κ. Σκουνάρ θα ήθελε ένα γραφ, το, να υπάρχει ένα γραφείο εδώ, ελπίζω σε μεταγενέστερη προθεσμία, σύμφωνα με το δικό σας μοντέλο να ακολουθήσουμε και εμείς ένα παρόμοιο. Νομίζω ότι κάλυψα όλα τα ερωτήματα που ετέθησαν. Ευχαριστώ κυρία Νίμπλερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Κόρντιν που ήρθατε, που μας δώσατε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Μπροστά σας κάθομαι. Η διατλαντική συνεργασία είναι νομίζω ένας. Η διατλαντική συνεργασία είναι, πιστεύω, πολύ σημαντική για μας από την ευρωπαϊκή πλευρά. Πάντοτε την εκτιμούμε ιδιαίτερως και ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε. Έχω πολύ ερωτήσεις, τρεις στον αριθμό. Καταρχάς εδώ Πολλέ φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για αρκετά χρόνια προσπαθούμε να οικοδομήσουμε τον ευρωπαϊκό χώρο της έρευνας. Από την ευκαιρία που είχαμε αποστολές, ταξίδια ως μέλος της Επιτροπής αυτής αλλά και ως πρόεδρος της ε, προσωπίας για τη με τα Ευρωπαϊκά κράτη, βλέπω ότι μπορούμε με προγράμματα να υποστηρίξουμε ερευνητικές προσπάθειες από ερευνητές σε ολόκληρο τον κόσμο που ίσως να μην είναι πολύ δημοφιλείς και που να μην έχουν την ευκαιρία να προσελκύσουν κονδύλια. Εσείς ως ε, Ηνωμένες Πολιτείες τι προτίμηση δείχνετε στην ερευνητική πολιτική. Λέτε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, ε, Έρευνας είναι έννοια γνωστή στις ΗΠΑ και ενδιαφέρει τους νέους ερευνητές. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Και επίσης, με τη φυσική καταστροφή που έχετε στον κόλπο του Μεξικού, εσείς στο Κογκρέσο τι συζητάτε και κυρίως σε τι συμπεράσματα καταλήγετε από αυτή τη μεγάλη πετρελαιοκυλίδα. Είναι πολλές οι ανησυχίες που εκφράζονται σε σχέση με ε, εξόριξη πετρελαίου στις θάλασσες και ίσως να πρέπει να αντιλήσουμε κάποια διδάγματα από το ατύχημα αυτό. Πολλά ακούγονται επίσης πολλές φορές για εναλλακτικά σενάρια σε σχέση με τις πλατφόρμες εξόριξης, πιο ασφαλείς λύσεις. Εσείς στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ τι συζητήσεις κάνετε. Και επίσης ένα ζήτημα συνείδησης, αν θέλετε, ένα ερώτημα συνείδησης. Εγώ είμαι Βαβαρή, προχωρώ από τη Βαβαρία, είμαι Γερμανίδα. Ε, βλέπω λοιπόν ότι στην Ευρώπη μεγάλο κομμάτι της έρευνας χρηματοδοτείται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στις ΗΠΑ Πολιτείες τι είδους ε, αναλογίες έχετε ως προς την ε, χρηματοδότηση των επενδύσεων ιδιωτικό τομέα, δημόσιο τομέα κλπ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και σύντομα παρακαλώ για να προλάβουμε να ακούσουμε όλες τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Κύριε Στροσχόνης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε. Είναι όντως... Γιατί είναι πολύτιμη εμπειρία του να έρχεται εδώ και να συμμετέχει στη ζήτησή μας και αναφερθήκατε προηγουμένως, αγαπητέ, εις ε, αυτήν την ε, συμβολή που αναδεικνύεται από την συνεργασία. Και εγώ πέρασα και έζησα τον ψυχρό πόλεμο και είδα τι θα πει ανταγωνισμός μεταξύ των πρωταγωνιστών της γεωπολιτικής. Περίπλοκα τα πράγματα και συνεργαστικά και είναι τα χρόνια της νιώτης μου και επίσης τότε σπούδαζα τις δυτικές επιστήμες, ξέρετε, και, αυτό ήταν συναρπαστικό. Έχω την εντύπωση πάντως, δεν ξέρω σωστά, είναι υποκειμενική αυτή η γνώμη μου, αυτή μου η άποψη, ότι έχουμε μία συγκεκριμένη μονόπλευρη αντιμετώπιση των επιστημών. Πέστε μα τη γνώμη σα. Γιατί το θέμα να δούμε τι θα κάνουμε τα προγράμματα, τι θα κάνουμε τους νέους, πώ θα τους δώσουμε κίνητρα. Εσείς, τι θεωρείτε ότι μπορούμε να κάνουμε. Τι σύμβολα μπορούμε να αναδείξουμε. Είναι σημαία η πρόοδος των επιστημών για τη ΣΥΠΑ, η αναζήτηση νέων δρόμων, η ΝΑΣΑ. Και θα πρέπει βέβαια να ξέρει κανείς προσπάθειες που κατατείνουν. Είναι βέβαια θέμα οικονομικό, είναι θέμα περίπλοκο, όμως τελικά θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα όπως γίνεται με την ΝΑΣΑ ή με κάτι άλλο το ίδιο σημαντικό κίνητρα και έτσι κανείς να μπορεί να πείσει τους επιστήμονες. Και βεβαίως σας ρωτώ πώς βλέπετε τη συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και ΝΑΣΑ στο μέλλον. Κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Γκόρντον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. σημειώνω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε και την Επιτροπή ΣΤΟΑ, στην οποία συμμετέχουν 13 βουλευτές, έχουν τον πρόεδρό τους και αξιολογούν τις προτάσεις στον τομέα των επιστημών, διατυπώνουν συστάσεις προς τις κοινοβουλευτικές επιτροπές για να διαμορφώνουμε εμείς τις απόψεις μας. Και ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει αντίστοιχη δομή στο Κογκρέσο. Επίσης, βλέπω ότι η Επιτροπή της οποίας εσείς ε, προεδρεύετε έχει και την εσωτερική ασφάλεια στον τομέα των αρμοδιοτήτων της. Μπορώ να ρωτήσω λοιπόν τι είδους ερευνητικά προγράμματα έχετε στην κύβερνο ασφάλεια, cyber security ιδιαίτερος. Και μια τελευταία ερώτηση σχετική με τη συνεργασία για την τυποποίηση, διεθνή τυποποίηση, όπου έχουμε καλή συνεργασία με τις Ηνωμένες και βέβαια πάντα θα έχουμε την ε, διάσταση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η κυρία Τζεβέλα παρακαλώ. Πρόεδρε και καλώς ορίζω τον ε, κύριο Γκόρντον ε, στην Επιτροπή μας. Πράγματι είναι χαρά μας και φαίνεται και από την ανταπόκριση των συμμετεχόντων ότι υπάρχει έδαφος για μια καλή και συγκεκριμένη συνεργασία. Ε, δύο σημεία θέλω να τονίσω και να ενημερώσω στα πλαίσια της ενδυνάμωσης της Ευρωατλαντικής Συνεργασίας η Επιτροπή ΙΤΡΕ κεφαλαιοποιεί την επίσκεψη του κυρίου Γκόρντον σε συγκεκριμένη βάση. Δηλαδή, συνήθως έχουμε μιλητές, ανταλλάσσουμε απόψεις, έχουμε καλές προθέσεις συνεργασίας, αλλά κάπου χανόμαστε στο follow-up. Σε αυτή την περίπτωση ε, εκμεταλλευτήκαμε την επίσκεψη του κυρίου Γκόρντον. Έχουν προβλεφθεί τα επόμενα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν σε ένα συγκεκριμένο project και ίσως αυτό συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και ίσως αυτό είναι και ένα pilot project το οποίο καθοδηγήσει και τις άλλες επιτροπές από την πλευρά του Κογκρέσου και την πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου πώς μπορούμε να συνεργαστούμε πιο στενά. Το δεύτερο που θέλω να σας ενημερώσω είναι ως ένα follow-up βήμα στην επίσκεψη και την αρχική μας συζήτηση με τον κύριο Γκόρντον, στις 16 Νοεμβρίου έχει προβλεφθεί η επίσκεψη του Dr. Holdren... ο οποίος είναι ο επικεφαλής, 16 Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία, είναι ο επικεφαλής της έρευνας και τεχνολογίας του Λευκού Οικού, ο σύμβουλος του κυρίου Ομπάμα, σε αυτόν που αναφέρθηκε ο κύριος Γκόρντον και ο οποίος έχει αναλάβει και τον συντονισμό της έρευνας και ε, ε, innovation στις Ηνωμένε Πολιτείε. Οπότε 16 Νοεμβρίου θα έχουμε πάλι έναν ομιλητή, ένα κεντρικό ομιλητή επί του θέματος και θα δούμε πού έχουμε φτάσει το follow-up της δουλειάς που ξεκινήσαμε με τον κύριο Γκόρντον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Bedanke mich ευχαριστώ και εγώ. Κύριε έχετε και πάλι το λόγο Ευχαριστώ. Ρωτήσατε τι γίνεται όσον αφορά το συντονισμό έρευνα μεταξύ ΙΠΑ ΕΕ και Ευρωπαϊκή Ενώσεω σε μεγάλο βαθμό. Αυτό βασίζεται στα πανεπιστήμια και δεν περνά από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Ήμουνα στο Cambridge το Σάββατο. Και ένα από τα πανεπιστήμια εκεί έχει άμεση σχέση με το MIT. Οπότε πολλά από αυτά είναι επαφές πανεπιστήμιο με πανεπιστήμιο. Και πολλά από τα εθνικά ιδρύματα, ε, επιστημονικά ιδρύματα, εργάζονται με τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα. Και μπορεί βέβαια να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμός, κυρίως στους μεγάλους τομείς η σύλληψη και αποθήκευση του άνθρακος, εκεί το συζήτησαν οι G8, αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε μέσω των ομοθετικών μας ακροάσεων, ίσως και εσείς, είναι να τους πιέσουμε να κάνουν κάτι, διότι αυτό είναι κάτι δαπανηρό. Ο άνθρακας θα υπάρχει μακρόν στη ΣΥΠΑ, στην Πολωνία και σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης. Ο άνθρακας είναι μεγάλο ποσοστό, αποτελεί μεγάλο ποσοστό της κινέζικης ενεργειακής πηγής στο μέλλον, ενεργειακών πηγών στο μέλλον. Αν αναπτύξουμε λοιπόν κάποιο είδη σύστημα σύλληψη και αποθήκευση του άνθρακου, θα είναι εποφελές προ όλου. Αργότερα, αυτό το μήνα νομίζω, θα, θα περάσει στην Επιτροπή μα μια διαδικασία διοδότησης για την πυρηνική ενέργεια, επίμαχο ζήτημα, αλλά σε πολυεθνή προσέγγιση θα πρέπει να το εξετάσουμε. Όταν μιλάω για έρευνα, μιλώ για τέταρτη γενιά οι εγκαταστάσεις να είναι φθηνότερες, οι αντιδραστήρες φθηνότεροι, μετά ε, πανεκατεργασία τους ώστε να απαλλαγούμε από το πρόβλημα της διάδοσης των πυρηνικών όπλων και μετά είναι το θέμα της αποθήκευσης. Καμία χώρα δεν έχει ε, κάποια, κάποιο χώρο αποθήκευση που χρησιμοποιείται κεντρικό σημείο. Χρειάζεται πολυεθνική προσέγγιση και μάλλον ε, διακρατική προσέγγιση και θα είναι κάτι ακριβό. Λοιπόν, Όσον αφορά τα άλλα θέματα, είμαστε μεταξύ φίλων. Η ΕΠΑ χρησιμοποιεί, δίνει μεγαλύτερη αξία στην έρευνά της από ό,τι άλλους τομείς. Ε, συμμετέχουμε. Αλλά η κατάσταση είναι γνωστή. Τώρα όσον αφορά και το πρόβλημα αυτό της διαρροής του πετρελαίου στον κόλπο ε, υπάρχουν, είναι σοβαρό πρόβλημα. Ήδη πέντε επιτροπές του Κογκρέσου εξετάζουν διάφορες στοιχές πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Τις επόμενες δύο εβδομάδες θα θεσπίσουμε κάποια νομοθεσία όλοι μαζί. Ένα κομμάτι του προβλήματός μας ποιο ήταν. Δεν ήταν η διαδικασία διοδότησης που δεν ήταν αρκετά αυστηρή θα έλεγα ότι οι γραφειοκράτες μας δεν παρακολούθησαν, δεν τήρησαν τους κανόνες. Ήτανε πολύ δέσμοι της βιομηχανίας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το να γνωρίζουμε, θα γίνουν κάποιες αλλαγές, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτού του είδους οι διεθνείς προδιαγραφές να εφαρμόζονται και να υπάρχουν. Ίσως από τις ακτές της Κούβας να υπάρξει μεγαλύτερη παραγωγή. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει εκεί, αλλά αυτό η παραγωγή στην Κούβα θα επηρεάσει εμάς. Θα πρέπει να υπάρχουν διεθνείς προδιαγραφές για την αδειοδότηση, διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα σχετικά με το πώς γίνονται οι γεωτρήσεις. Και μετά, προσωπική άποψη, θα πρέπει να λέμε σε μια εταιρεία. Αν διαλέξετε να μην συμμορφωθείτε όσον αφορά τι προδιαγραφέ, κοντά στι ακτέ τη Αγγλία ή ξέρω εγώ οπουδήποτε αλλού, θα λέμε αν δεν κινηθείτε σωστά εκεί δεν μπορείτε να έρθετε στα δικά μας παράκτια ύδατα ούτε. Και θα πρέπει εκεί να είμαστε μαζί ενωμένοι. Θα γίνουν αλλαγές πιστεύω. Όσον αφορά το ποσοστό έρευνας, περίπου τα δύο τρίτα της έρευνάς μας στη χώρα μας διεξάγεται το ιδιωτικό τομέα. Ένα τρίτο περίπου από το δημόσιο. Όμως, εδώ υπάρχει ένας όρος. Το συντριπτικό ποσοστό της βασικής έρευνας γίνεται στο δημόσιο τομέα, από δημόσια χρήματα. Και τα περισσότερα ιδιωτικά χρήματα χρησιμοποιούνται να πάρουν αυτή τη βασική έρευνα και να τη μετατρέψουν σε εφαρμοσμένη έρευνα. Έχω ένα σημείωμα εδώ. Τι έχω σημειώσει. Με βάση τον κίνδυνο, δεν θυμάμαι περί σε πρόκειται η ΝΑΣΑ. Α, κίνδυνος Τέλο πάντων, είναι εθνικό θησαυρό η αν θέλετε. Ε, εθνικό κοιμήλιο. Εμεί έχουμε μεγάλες δυσκολίες για να αποφασίσουμε το μέλλον της ΝΑΣΑ. Ποιο είναι το πρόβλημα, είναι το εξή. Δεν το λέω κομματικά. Τις χρονιές όμως, τα χρόνια του Μπούς, η ΝΑΣΑ ε, της ανέθεταν περισσότερες αποστολές από ό,τι χρήματα. Και κάπου πρέπει να πληρωθεί ο λογαριασμός. Οπότε είστε στα χέρια μας. 17 δις δολάρια προπολογισμό, με 23 δις όμως αποστολέ. Οπότε προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Σχέση μεταξύ ΝΑΣΑ και εμπορικού τομέα. Σχέση μεταξύ ΝΑΣΑ και διεθνών εταίρων. Κάποια κυρία, εσείς αναφέρατε, κάτι, ότι φαίνεται ότι έχουμε κολλήσει. Ναι, χρειαζόμαστε μια αποστολή. Θα πάμε, στο, θα πάμε σε αστεροειδή, θα πάμε στη σελήνη, πού θα πάμε. Προσπαθούμε αυτό να εξετάσουμε τώρα. Όσον αφορά το ΣΤΟΑ, το δικό σας, εμείς δεν έχουμε κάποια παρόμοια επιτροπή. Αλλά μέσω της δικής μας επιτροπής αδειοδοτούμε διάφορες έρευνες και δίνουμε κάποιες κατευθύνσεις. Εμείς είμαστε, είμαστε πιο ήπιοι, πιο ελαστικοί όσον αφορά τη διάθεση των πόρων στον Εθνικό Φορέα έρευνα. Και τους αφήνουμε να κάνουν αυτό που θεωρούν καλύτερο. Όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, Πέρασε η Επιτροπή μα για την έρευνα τη σχετική, πέρασε νομοθεσία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, σημαντικό διεθνεί προδιαγραφέ, είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία. θέλουμε να καταλήξουμε σε κάποια ωφέλη από την εφαρμογή των προδιαγραφών. Ελπίζω ότι θα γίνουν περισσότερα πράγματα σε συνεργασία μεταξύ μας σε αυτούς τους τομείς, στον τομέα των προδιαγραφών υπάρχει φορέας εντός της Ομοσπονδιακή Κυβερνήσεως, Εθνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Προδιαγραφών, που ανήκει στη δικαιοδοσία μας και τους προωθούμε σημαντικά. Είναι ε, εθελοντική η χρήση του. Ε, έρχονται επιχειρήσεις και χώρες χωρίς έλεγχο. Η νίκη μάλιστα πρέπει να δεχτείτε τα συγχαρητήριά μου που βοήθησε αυτό, δηλαδή να εξε... που πρόθεσε αυτό να εξετάσουμε τα αποτελέσματα που παίρνουμε όσον αφορά τα χρήματά μας. Έχουμε ένα σύστημα μέτρησης, ο πρόεδρος Ομπάμα έδωσε ένας έδωσε πόρους για να τονωθεί η έρευνα και τώρα θέλει να δει τα αποτελέσματα, να δει τι, τι καρπούς δρέπουμε για τις προσπάθειές μας. Είναι διτή προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να βοηθηθούμε πολιτικά για να πούμε έχουμε τόσα προϊόντα, τόσες απασχόλησεις Λοιπόν, αν επενδύσετε περισσότερο, θα δείτε περισσότερα αποτελέσματα. Και το άλλο, χρειάζεται μεγαλύτερη κατανόηση ότι ένα δολάριο που επενδύεται κάπου μπορεί κάπου να πάρει ένα και δέκα και κάπου αλλού να γίνει τρία δολάρια. Οπότε Νίκη ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια να συνεργαστεί με το εθνικό μας Ίδρυμα η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξετάσουμε αυτό το σύστημα μέτρησης και σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές και όπως είπε η Νίκη, θα έρθει και ο Δόκτωρ Χόλτρε να σας δει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο και ξέρω ικανότατο πρόσωπο και πολύ σημαντικό στον τομέα τον ερευνητικό. Είναι σύμβουλος του Προέδρου. Είναι μέλος της, του, του Royal Society της Βρετανίας και καταλαβαίνει και εκείνος και ο Πρόεδρος ότι χρειάζεται συνεργασία μεταξύ μας. Είναι δύσκολο από πολιτική σκοπιά, λόγω δύσκολων οικονομικών καιρών, αλλά θα είναι καλός ε, εκπρόσωπός μας για να μπορέσετε να συζητήσετε μαζί του αυτά τα θέματα. Επιτρέψτε μου, Mr. Congressman, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Είναι, θα έλεγα, μια πολύ καλή ευκαιρία, μια πρώτη ευκαιρία για μας βέβαια, αλλά ελπίζω να μην είναι η τελευταία. Εσείς από ό,τι φαίνεται έχετε ήδη επισημάνει την ανάγκη για θεσμοθέτηση αυτής της συνάντησης συνεργασίας. Ε, μια πιο τακτική μάλιστα επικοινωνία θα ήταν σκόπιμη, όχι μια περιστασιακή αλλά τακτική οργανωμένη συνάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Εύχομαι κάθε καλό στις εργασίες σας.